Uh, good morning, um, Καλημέρα σε όλους. Είναι πάνω κάτω η ώρα να αρχίσουμε. Περιμένουμε και τον κύριο Μάντελς να κάτσει. Λοιπόν, κανονικά έχετε ένα επικαιροποιημένο πρόγραμμα για σήμερα στις θέσεις σας. Θα πρέπει να διορίσουμε εισηγητές ε, σήμερα για διάφορους ε, φακέλους που θα συζητήσουμε σήμερα το πρωί και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Θα ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για τα κλωστοϊφαντουργικά και θα συζητήσουμε και κάποια άλλα ζητήματα ε, σήμερα το απόγευμα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με την οδηγία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Είναι βασικό ε, φάκελο για μα. Έχουμε οργανώσει ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος ε, ο εισηγητής, θα ηγηθεί τη συζήτηση. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας για σήμερα. Πάμε στο πρώτο σημείο θα συνεχίσουμε ουσιαστικά ε, τις εργασίες ε, που είχαν αρχίσει την προηγούμενη θητεία για την ε, πρόταση της Επιτροπής για τη σήμανση των προϊόντων της κλωστοϊφαντουργίας από πλευρά της Επιτροπής. Αλλάζει ο εισηγητής. Ο κύριος Τουάιν Μάντερς που τα περασμένα πέντε χρόνια είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή μας, τώρα αναλαμβάνει η ε, σε αυτό το φάκελο και έχουμε και τους κοιόδες εισηγητής, κυρία Κούνη, ε, μία από τις ε, ε, αντιπρόεδρους, ε, η κυρία Σαλντεμόζα. Κυρία Σαλντεμόζα. Θα δώσω το λόγο σε όποιον το επιθυμεί μετά από την παρουσίασή μου. Επίσης έχουμε την Επιτροπή, τον κύριο Λουίς Φιλίπ Τζεράου, Ελπίζω να το πρόφερα σωστά. Θα μιλήσετε εξ ονόμως Επιτροπής, έτσι δεν είναι. Από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Επιχειρήσεων. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Επιχειρήσεων, λοιπόν, ο κύριος Τζεράρ που είναι προϊστάμενος εκεί. Θα ακούσουμε την ε, τοποθέτηση του εισηγητή, τον, ε, του σκιώδη εισηγητή και μετά πάλι την Επιτροπή. Κύριε Μάντες, παρακαλώ. Θα αρχίσετε τη συζήτηση. Uh, Ευχαριστώ, Μάλκομ. Ευχαριστώ που μου δίνεις το λόγο. Φυσικά μιλάμε για τη σήμανση των κλωστοϊφαντουργικών. Ε, όσοι δεν γνωρίζουν το θέμα, σας έφερα και ένα παράδειγμα. Μία, δύο, τρεις ετικέτες, τέσσερις ετικέτες, πέντε ετικέτες για... Για... και με γράμματα τόσο μικρά που πρέπει να βάλω και γυαλιά για να τα διαβάσω. Και μπορείτε να δείτε στα Ιταλικά, ε, Γαλλικά, όπως λέμε τον πολυεστέρα, αλλά δεν... Απλά ε, ήθελα να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να διευκρινίσω το αντικείμενο της συζήτησή. Μπορείτε να το δώσετε και στους συναδέλφους να το μελετήσουν, λέει ο Πρόεδρος. Yeah. So actually what I ask myself, uh, who is... Αναρωτιέμαι. Ποιο κάθεται να διαβάσει αυτή την εφημερίδα, γιατί η εφημερίδα είναι με τόσε ετικέτε όταν πάει κανεί να κάνει jogging το πρωί. Οι περισσότερε πληροφορίε είναι υποχρεωτικέ. Ε, Κάποιε βασίζονται στην αυτορύθμιση, γιατί έτσι θέλουν η παραγωγή, αλλά στο τέλο θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα. Κύριε Γκράου, σας ευχαριστώ. Είναι ο προκάτοχός μου που ήδη έκανε πολύ καλή δουλειά και πάνω κάτω είναι όλα έτοιμα ήδη και μπορούμε να ε, βασιστούμε σε αυτά που ήδη έχει κάνει για το μέλλον. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της έκθεσης? να επισπεύσουμε τη διαδικασία θέση εμπορία νέων υφασμάτων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Αν το πετύχουμε αυτό, και τυποποιήσουμε τις κανονιστικές ρυθμίσεις για τη θέση εμπορία των νέων υφασμάτων στην Ευρώπη, στην εσωτερική αγορά. Αυτό θα είναι υποφελές για τη βιομηχανία. Μία άδεια θα χρειάζεται πλέον και μπορείτε να αγγίξετε 500 εκατομμύρια καταναλωτές σε όλη την χώρια αγορά υπάρχει κάτι παράξενο. Δεν είναι και η μήτρική μου τα αγγλικά όπως θα έχετε καταλάβει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την οδηγία. Ε, παράρτημα 8, ε, τμήμα 2, κεφάλαιο 2. Ε, τι λέει εκεί, ότι αυτό ισχύει για ε, τις σε ε, κάθε είδους ε, στο μέτρο που δεν είναι μείγμα, mixture, Θέλω να συνεχίσω. Και ε, έχουμε τις πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μειωθούν γιατί ο καταναλωτή πλημμυρίζεται από τόσε πληροφορίε. Έχουμε τον πολυεστέρα που γράφεται πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο, διάφορε ίνες πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη προσέγγιση στην εσωτερική αγορά, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, αν είναι δυνατόν, να ξεφορτωθούμε όλες αυτές τις υποχρεωτικές μεταφράσεις στις διάφορες γλώσσες που μας επιβάλλει ο κανονισμός. Ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μειωθούν μία γλώσσα, παραδείγματος χάρη, ή απλά ε, να αναφερόμαστε στην ε, Ίνα και ίσως να φτιάξουμε μια ιστοσελίδα και άμα θέλουν οι καταναλωτές να πάνε να βρουν στην ε, μητρική τους γλώσσα όλες τις ε, πληροφορίες για ε, το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη τεχνική ονομασία αυτής της ίνας. Μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές μια τέτοια ιστοσελίδα και Καλό θα ήταν να ξέρουμε τι θέλουν οι καταναλωτές. Αν τους αρέσουν όλες αυτές οι γλώσσες στην ετικέτα, ίσως δεν πρέπει να αλλάξουμε τίποτα. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται. Ε, κυρίως μιλώντας για τις μεταφράσεις, έτσι, στις ετικέτες. Θέλουμε να τυποποιηθούν οι μέθοδοι και να τις απλουστεύσουμε τις μεθόδους της εμπορία και να τις επισπεύσουμε. Τώρα χρειάζονται τρία-τέσσερα χρόνια πριν πάρετε την άδεια για να εισάγετε στην αγορά νέα ή να... Αν μπορούμε να μειώσουμε την περίοδο σε έξι μήνες ή κατανότα το όριο ένα χρόνο, θα ήταν καλό για τους καταναλωτές, για τη βιομηχανία, για ολόκληρη την κοινωνία. Μετά, έχουμε την ετικέτα για το πώς πλένει κανείς το ρούχο, πώς το φροντίζει. Ε, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά το βάζουν όλοι οι παραγωγοί. Η γυναίκα μου, Φερρυπίν, μου είπε ότι χαίρεται που υπάρχει η ετικέτα γιατί είναι πιο εύκολο έτσι να ξέρει πώς ακριβώς να το πλύνει για να μην χάσει το χρώμα του και τη φόρμα του ρούχο. Είναι χρήσιμο. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι πρέπει να πληρώνουν οι καταναλωτές για τις ταμπελίτσες γιατί υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα πρέπει να πληρώσουν το αντίτιμο σε κάποια οργάνωση και θα ήταν χρήσιμο να σκεφτούμε το εξής οι ετικέτες κοινοτικέ που θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, δωρεάν όμως για τους καταναλωτές και αυτό θα ήταν πλεονέκτημα για αυτούς. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό σε κάποιες χώρες είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται, σε άλλες όχι. Ε, γι' αυτό και πρέπει να ε, πετύχουμε μια εναρμόνιση για ολόκληρη την ενιαία αγορά. Αν ε, μπορούμε να το ξεφορτωθούμε, δεν ξέρω με ποιο τίμημα, ποια τι πληρώνει ο καταναλωτής για τα πνευματικά δικαιώματα, για αυτά τα... Για αυτά τα εικονογράμματα. θα μπορούσαμε ίσως να σχεδιάσουμε καινούργια που θα έχουν τις ίδιες πληροφορίε και έτσι ε, να βοηθήσουμε τους καταναλωτές. Μετά έχουμε τα παραρτήματα, το 5 παραδείγματο χάρη, όπου περιγράφονται τα κλωστοφαντουργικά προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται καμία σήμανση. Ε, και κάποια παιχνίδια, ε, τα γάντια παραδείγματο χάρη, για το φούρνο. Ε, μπορούμε να το συζητήσουμε με τους ε, σκιώδεις εισηγητές αν χρειάζεται σήμανση ή όχι για κάποια προϊόντα. Πρέπει να το σκεφτούμε. Πάντω είχαμε και αυτή την ιδέα. Ζήτησα από τη γραμματεία της Επιτροπής μας να ε, φτιάξει ένα ενημερωτικό σημείωμα για κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να ελέγξουμε αν πρέπει να εναρμονίσουμε αυτές τις ετικέτες για τη φροντίδα των ρούχων, πλήση λοιπά. Γιατί ε, θέλουμε να προετοιμάσουμε σωστά τα προϊόντα για τους καταναλωτές, αλλά ίσως αυτό δεν αντιστοιχεί στις προσδοκίες τους. Μπορεί να τους αρέσει το σύστημα όσο έχει. Ε, αυτό το ξέρουμε ακόμη. Ε, χρειάζεται λοιπόν εναρμόνιση στον τομέα αυτό. Επίση, απαιτήσει ε, για την υγεία ε, ή για την υγιεινή. Ε, του ενδιαφέρουν τους καταναλωτέ αυτές τις ρυθμίσει. Η Eurostat, η μπορεί να έχει ήδη στη διάθεσή της ε, πολλές πληροφορίες και η γραμματεία μπορεί να βρει τέτοιες πληροφορίες, να καταλάβουμε ε, τι πιστεύουν οι καταναλωτές για τις απαιτήσει για την υγιεινή παραδείγματο χάρη και κάτι άλλο στο οποίο αναφέρθηκα ήδη. Στο παράρτημα 5 έχουμε τον κατάλογο των προϊόντων ε, που αποκλείονται από την υποχρέωση σήμανσης, να δούμε αν χρειάζεται η σήμανση σύμφωνα με τους καταναλωτές και κάτι άλλο. η χώρα προέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ή όχι ε, στο προϊόν. Μετά, ε, όταν λέμε χώρα προέλευση εννοούμε χώρα παραγωγής ή εκεί πέρα που ε, προσθέθηκε, ε, δηλαδή όπου προέρχεται η οχι στο προιον μετα οταν λεμε αξία, ένα κομμάτι της παραγωγής δηλαδή. σε μία επίσκεψη στην Κίνα, παραδείγματο χάρη, είδαμε ένα τεράστιο εργοστάσιο όπου εκατοντάδε, ε, χιλιάδε κουστούμια Hugo Boss παράγονταν ε, και έλεγε πάνω Made in Germany, ότι έχει φτιαχτεί στη Γερμανία γιατί βάλαν κάτι κουμπιά στη Γερμανία και άρα πήρε την ονομασία σαν να είχε παραχθεί στη Γερμανία. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Απλά ε, τι θα θεωρήσουμε, ότι έχει παραχθεί ε, στη Γερμανία ή εκεί ε, έχουμε την προσθέμενη αξία στο προϊόν. Κάπως θα πρέπει να ενημερωθούν και οι σε σχέση με αυτό. Να λοιπόν κάποιες σκέψεις που είχα τις περασμένες εβδομάδες. Σίγουρα θα βρούμε λύση γιατί είπαμε είναι καλό για τη βιομηχανία και για τους καταναλωτές και ελπίζω να τα καταφέρουμε να συνοηθούμε με όλους τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους υπόλοιπους που ε, γνωρίζουν το θέμα. Είμαι πεπισμένο ότι τις προσεχεί εβδομάδες, μήνες ε, θα έχουμε νέα. Ε, έχω και ένα χρονοδιάγραμμα σας προτείνω αν θέλετε. Το έχουμε ήδη συζητήσει. 15 Οκτωβρίου να στείλουμε για μετάφραση την έκθεση. 4 Νοεμβρίου εξέταση του σχεδίου έκθεσης. 16 Νοεμβρίου καταληκτική ημερομηνία για υποβολή τροπολογιών. Δεκεμβρίου εξέταση των τροπολογιών. Την επόμενη μέρα ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και τον Ιανουάριο, αν γίνεται, ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Επισπεύουμε τη διαδικασία. Ήδη έχουμε επεξεργαστεί το φάκελο και απλά πρέπει να το τελειοποιήσουμε. Ε, να το... Και να ε, έχουν τελειώσει όλα τον Ιανουάριο. Λοιπόν, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Good. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί ε, ξεκινήσατε αυτή τη συζήτηση με το χαρακτηριστικό σας στυλ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, τώρα νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα από μεριά μα δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Να αφήσω όμω του σκιώδει ηγητέ να το σχολιάσουν. Και επίση, όσον αφορά ε, του συντονιστέ χθε, αποφάσισαν να να, να φροντίσουμε να υπάρξει ένα ενημερωτικό σημείο. Έχουμε κάποιου πόρου και θα μπορούσαμε να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίε ε, για το θέμα αυτό. Με την προπόθεση βεβαίω ότι συμφωνείτε με του σκιώδει όσον αφορά τι προδιαγραφέ ε, τη εργασία αυτή, εμεί πολύ γρήγορα θα φροντίσουμε να υπάρξει. Ε, να ακούσουμε του σκιώδε και πρώτα απ' όλα να ε, ζητήσω την κυρία, από την κυρία Κόμη να συμβάλλει στη συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια καινούργια εμπειρία για μένα. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα εργασία θα είναι πάρα πολύ καλή, θα εργαστούμε όλοι από κοινού ε, και θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Ήδη βλέπετε ότι ασχολούμαστε με τα πρακτικά θέματα και αυτό όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πιστεύω ότι η πρόταση αυτή, την οποία την ανέλησε και ανέλησε σε λεπτομέρειε στον κανονισμό, Σίγουρα πιστεύω ότι η πρόταση αυτή ε, είναι εξαιρετική. Δηλαδή πράγματι πρέπει να ε, αναπτύξουμε, να προωθήσουμε αυτές τις νέες σύνες, αλλά και να προστατεύσουμε όλους και τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις, να βοηθήσουμε δηλαδή αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με, τις νέες, ε, με τα νέα αυτά προϊόντα. Ταυτόχρονα συμφωνώ ότι θα πρέπει να απλοποιήσουμε τα πράγματα και από γραφειοκρατική άποψη και να δούμε όλες τις διαδικασίες ε, που έχουν να κάνουν με την ονομασία αυτών των νέων ινών και βεβαίω ε, το γραφειοκρατικό ζήτημα σχετίζεται άμεσα και με τα εικονογράμματα, με τα σύμβολα αυτά. Σύμφωνο λοιπόν ότι πρέπει να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία και όσον αφορά την ετικέτα. Αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη νομοθεσία, οι οδηγίες, κυρίως οι τρεις οδηγίες για τα κλώστα εφαντουργικά, αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό εργαλείο. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε, ένα, σε μια επιτυχή που έχει να κάνει με τη νέα τεχνολογία. Αφορά λοιπόν τις νέες ίνες. Είμαι από την Ιταλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα εκλοστιφοντουργικά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο τομέας παρουσιάζει κρίση. Οι δυσκολίες είναι πολλές και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι, βιοτέχνε, και οι βιοτέχνες. Όλοι αυτοί δηλαδή ε, που ασχολούνται σε μικρή κλίμακα με την, με την παραγωγή κλωστεφαντουργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε με την ομάδα εργασία κατά πόσον θα πρέπει να αναφερθούμε και στις επενδύσεις και στι χρηματοδοτήσει, αν θέλετε, προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Έτσι ώστε και αυτέ να μπορέσουν, πώ μπορούμε να τι βοηθήσουμε, έτσι ώστε να αναπτύξουν αυτέ τι νέε ίνε με την ε, πλέον εξελιγμένη τεχνολογία. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα βοηθήσουμε μόνο τι μεγάλε επιχειρήσει, αυτού δηλαδή που έχουν τα απαραίτητα κονδύλια για να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και δεν θα βοηθήσουμε καθόλου του βιοτέχνε και αυτέ τι μικρέ επιχειρήσει που τουλάχιστον στη χώρα μου ε, αποτελούν το 80% των επιχειρήσεων και αναπτύσσουν δραστηριότητες ε, και παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια πιο ευέλικτη διαδικασία. Έτσι ώστε να βοηθούν αυτέ οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα ήθελα να το αναλύσουμε καλύτερα στι λεπτομέρειέ του. Συμφωνώ. Βεβαίω, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίε και να και τον Ιανουάριο να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Ταυτόχρονα όμως ε, θα ήθελα ε, να ακούσουμε και τις απόψεις του κλάδου, ε, των διαφόρων οργανώσεων, των καταναλωτών, δηλαδή ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή μα, έτσι ώστε να πούν όλη τη γνώμη τους και τελικά να καταλήξουμε σε μια νομοθεσία, σε ένα κανονισμό με τον οποίο να συμφωνούν όλοι. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, να υπάρξουν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, που να μας βοηθήσουν να τα πετύχουμε όλα αυτά. Να υπάρξουν οι διάφορες συναντήσεις, τα διάφορα ραντεβού αν θέλετε, και μετά βεβαίως και να έχουμε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Συμφωνούμε να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο, πολύ ωραία. Αλλά ε, όσον αφορά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Συμφωνώ Απολύτω, ε, με όλε αυτέ τι διαδικασίε. Όσον αφορά την ετικέτα, βεβαίω είναι μεγάλε αυτέ οι ετικέτε και αναφέρουν πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Πιστεύω όμω ότι για να είναι καλό το αποτέλεσμα τη εργασία μα πρέπει να ακούσουμε και του καταναλωτέ. Τι πιστεύουν οι καταναλωτέ. Και βεβαίω ε, οι διάφοροι εκπρόσωποι του κλάδου παραγωγή. Και οι μόδα, αν θέλετε, που συνδέονται με όλα αυτά. Προστασία κυρίω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί στον κλωτοφαντουργικό τομέα πλήττονται ιδιαίτερα νομοθεσία που να βοηθά και τους καταναλωτές, αλλά και όλους αυτούς που παράγουν αυτές τις νέες ίνες. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστώ κυρία Κόμη. Η επόμενη ομιλητρία. Ε, ε, ευχαριστώ. Θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Ρομάντες για μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτού του ζητήματος. Έχουμε πολλά σημεία τα οποία θίγονται σε σχέση με αυτή την πρόταση, αλλά ίσως ε, σας διέφυγε μία πτυχή. Εδώ στην αίθουσά μας ε, λοιπόν υπάρχει μία επιπρόσθετη πτυχή την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, ε, δηλαδή το μέγεθος των χαρακτήρων και το γεγονός ε, που αναφέρατε ότι θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει τα γυαλιά του για να ε, διαβάσει το τι αναφέρεται. Αυτό λοιπόν το ζήτημα του μεγέθους των χαρακτήρων σας διέφυγε νομίζω μέσα σε αυτή την πρόταση, αλλά κατά τα άλλα συμφωνούμε πάρα πολύ με το πνεύμα αυτή τη πρόταση, γιατί πραγματικά θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ό,τι αφορά τη σήμανση κλωστοϊφαριδοτικών προϊόντων. Όμως ε, τελικά το ζητούμενο για μας είναι ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στον καταναλωτή. Δηλαδή το κατά πόσο τελικά είναι χρηστικές ε, και μπορούν να αξιοποιηθούν από τον καταναλωτή οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτές τις ετικέτες. Καλό θα ήταν λοιπόν να εξετάσουμε κάποια στιγμή ε, τι ακριβώς συμβαίνει από την πλευρά των καταναλωτών σε σχέση με αυτές τις ετικέτες. Τις εξετάζουν, τις διαβάζουν ε, να βλέπουμε δηλαδή κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν από το καταναλωτή. Από εκεί και μετά, σε σχέση με τα ζητήματα υγεία, συμφωνούμε και εδώ με την στάση σας. Είπατε δηλαδή ότι ε, εν λόγω στατικές ουσίες δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνες και μετά από, την, ε, από τον εμποτισμό των ούχων με χημικές ε, χρωστικές ουσίες και ούτω καθεξής. Ναι, δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά δηλαδή την ε, ασφάλεια του καταναλωτή και από εκεί και μετά την ε, ονομασία της ε, προέλευσης προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο να αναφέρεται θα πρέπει να βρούμε μια λύση αλλά σίγουρα αυτή η λύση θα πρέπει να είναι ορατή από τον καταναλωτή. Δηλαδή θα πρέπει ο καταναλωτή να γνωρίζει κατά πόσο το εν λόγω ρούχο έχει παραχθεί στην Ινδία ή στη Γερμανία ή τίποτα άλλο. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των γλωσσών που αναφέρονται στι ετικέτε επί της αρχής ε, συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει να, αναφέρεται, να αναφέρονται ίδιες πληροφορίες ε, σε, σε 5-6 γλώσσες ε, και σε 5-6 διαφορετικές ετικέτες καθώς πολλές φορές είναι ενοχλητικές αυτές οι ετικέτες αλλά ταυτόχρονα κάτι τέτοιο είναι δημιουργεί κάποια προβλήματα ενδεχομένω. Μπερδεύει δηλαδή το καταναλωτή αν έχουμε πολλέ γλώσσε. Όμω θα πρέπει να το συζητήσουμε λίγο πιο εντελεχώ αυτό το ζήτημα, γιατί ναι μεν δεν θέλουμε να δώσουμε υπερβολική πληθώρα πληροφοριών στον καταναλωτή, αλλά ούτε θα πρέπει να τον περιορίσουμε ως προς την ενημέρωσή του. Τώρα, το τι θα κάνουμε με αυτή την ε, πρόταση. Συμφωνούμε καταρχήν ε, με τα όσα προτείνεται. Ε, υπάρχουν πολλές πτυχές ε, που αφορούν αυτό το ζήτημα και που θα πρέπει να συζητηθούν. Άλλωστε δεν βρισκόμαστε υπό πίεση χρόνου. Ε, ας εξετάσουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα με την ησυχία μας. Ε, το χρονοδιάγραμμα λοιπόν που προτείνεται είναι ε, σωστό και βέβαια αν θεωρήσουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο μπορούμε να το αναβάλουμε λιγάκι. Δηλαδή, για παράδειγμα, να θέσουμε την προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών το Δεκέμβριο κάπου. Αλλά κατά τα άλλα, σα λέω, σε γενικέ γραμμέ μα αρέσει αυτή η πρόταση για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Α, κυρία Ρούλα θέλει το λόγο. Μάλιστα. Θα καλύψει λοιπόν το θέμα για τους πράσινους. Δεν ξέρω, κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Είσαι άργουε. Ωραία. Λοιπόν, θα ζητήσω από την κυρία Ρούλε να τοποθετηθεί και μετά ε, θα έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα να αναφέρω μόνο ένα ζήτημα. Όταν συζητούμε λοιπόν τη σήμανση, σήμανση προϊόντων, θα πρέπει να γνωρίζουμε πω έχουμε όλο και περισσότερου ανθρώπου οι οποίοι υποφέρουν από αλλεργίε. Και αυτέ οι αλλεργίε σχετίζονται πολύ συχνά με γλυκοσυφαρτητικά προϊόντα και όχι μόνο με τι χωριστικέ ουσίε επάνω σε αυτά, αλλά και με τα ίδια τα συστατικά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει, είναι σημαντικό να γνωρίζουν από τι αποτελείται ένα συγκεκριμένο ρούχο. Ακριβώς γιατί ε, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες νέες τεχνολογίες ε, στην ε, παραγωγή των ρούχων. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καταναλωτής, δηλαδή κατά πόσο είναι ένα συγκεκριμένο ρούχο καλό για την υγεία του ή όχι. Και συμφωνούμε μετά όσο προτείνει εδώ ο κύριος Μάντερς. Ε, σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση όμως ότι δηλαδή θα μπορούσαμε να περικόψουμε το κόστος ε, μέσω ε, της δημιουργίας κάποιων νέων συμβόλων είμαστε πολύ επιφυλακτικοί γιατί θέλουμε να έχουμε διεθνή σύμβολα καθώς κανείς προβαίνει σήμερα σε αγορές σε όλο τον κόσμο και άρα θα πρέπει τα σύμβολα να είναι ίδια όπου και αν κάνει τις αγορές του είτε είναι στις ΗΠΑ είτε στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενιαία σύμβολα ε, παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Uh, uh, Καλώς ολοκληρώσαμε εδώ με τον ε, ε, κύριο τη συζήτηση ό,τι αφορά του στιώδει συζητητέ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον ε, συγητή αλλά και την σκιώδη συγκήτριά μα ε, για τη δουλειά που έχει γίνει και το γεγονός ότι θα μπορέσουμε ήδη από τον Ιανουάριο να πάμε σε σφοφορία. Βέβαια, σε σχέση με αυτό το ζήτημα προκύπτουν μία σειρά από επιμέρους ζητήματα που έχουμε συζητήσει στο πλαίσιο των συντονιστών. Για παράδειγμα, η πρόταση του κυρίου Μάντερ για την δημιουργία ε, νέων ε, ετικετών ε, συμπίπτει και με τις προτάσεις που έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά την εκ νέου εξέταση των ετικετών και τη σήμανση γενικά στα καταναλωτικά προϊόντα στην Ευρώπη. και δεν είναι προφανώς θετικό κάθε φορά που έχουμε μία νέα συστατική ουσία να υπάρχει μία νέα πρόταση σε ό,τι αφορά την σήμανση. Ε, κάτι τέτοιο δεν δίνει δηλαδή το σωστό μήνυμα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι πολύ ετερογενής εδώ η αγορά. Δηλαδή έχουμε, κάποιο, έχουμε τους μεγάλους ε, ε, πολιτές της Μεγάλης οι οποίες προβαίνουν σε εισαγωγές από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας ενώ έχουμε ταυτόχρονα ανταγωνισμό ε, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εισάγουν από την ε, Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν ενδεχομένως τα ζητήματα που αφορούν αυτήν την ετερογένεια θα μπορούσαν ενδεχομένως να καλυφθούν από αυτή την πρόταση και όχι μόνο να περιοριστούμε απλά στην, ε, στις ετικέτες που θα αφορούν σε νέες, κάποιες νέες κλωστές ή οτιδήποτε άλλο σε ό,τι ε, είπατε σε σχέση με μια σχετική διοργάνωση, ναι, θεωρώ πως θα ήταν πολύ θετικό να υπάρξει και μια τέτοια αποστολή, ενδεχομένω ε, όπως ε, ανέφερε και η κυρία ακόμη, θα μπορούσαμε δηλαδή να ρίξουμε μια ματιά, αλλά ε, κυρία Ρούλε, είχατε δίκιο σε αυτά που είπατε και υπάρχει και βέβαια διαφορά ανάμεσα στα όσα αφορούν άντρες και γυναίκες. Γιατί εγώ φοράω για παράδειγμα πολύ συχνά βαμβακερά και με ενοχλούν πάντοτε οι ετικέτες και θα πρέπει να τις ε, κόβω. Όμως ε, θα πρέπει να θυμίζουμε ότι κατά τα τελευταία 5-6 χρόνια οι αλλεργίες που σχετίζονται με τα ρούχα ε, έχουν μειωθεί σε αντίθεση με την σημαντική του αύξηση κατά τη δεκαετία του 90. Ε, εγώ λοιπόν ε, ε, νιώθω μια ασφάλεια σήμερα σε ό,τι αφορά τα ρούχα που φορά τα δικά μου παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, εν γέννη συμφωνώ με τα όσα προτείνονται μέσα σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, κυρία Γεπχάρη. ευχαριστώ. Βλέπω πως πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο για το οποίο υπάρχει κάποια συναισθηματική φόρτιση στη συζήτηση, γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο βέβαια αφορά την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων και κατά συνέπεια δημιουργεί μια διαφόρτιση. φόρτιση. Ε, σε σχέση με τα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Μάντερσε και ο κύριος Σφάμπ, ε, να πω ότι εγώ ε, ναι ρίχνω πάντα μια ματιά στι ετικέτε γιατί έχω πρόβλημα με ορισμένες ε, είναι, οπότε για μένα είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμες αυτές τι πληροφορίες και μάλιστα σε γλώσσε τι οποίες ε, κατανοώ. Άρα λοιπόν πραγματικά δεν μπορούμε να μην έχουμε αυτές τις πληροφορίες επάνω στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε Και σα λέω ότι μερικές φορές ε, κοιτώ, διαβάζω την ετικέτα πρωτού καν αγγίξω ένα συγκεκριμένο ρούχο. Άρα λοιπόν υπάρχουν εδώ άνθρωποι και μέσα εδώ στο κοινοβούλιο ε, για του οποίου αποτελεί ζήτημα υγεία το να υπάρχουν ε, και να περιλαμβάνονται τέτοιου είδους πληροφορίε στι ε, Από εκεί και μετά. Αυτό η τεράστια πληθώρα ετικετών που έχει σημειωθεί δεν νομίζω πως οφείλεται στους, στον νομοθέτη αλλά στους ε, προς το τους τους παραγωγούς των ρούχων. Εμείς ε, δεν είπαμε για παράδειγμα στη Γερμανία δεν υποχρεώνουμε ε, κάποιον ε, παραγωγό ε, να ε, διαθέτει αυτές τις πληροφορίες σε άλλες γλώσσες. Στη Γερμανία ζητούμε στα γερμανικά, στην Ιταλία ζητούν στα ιταλικά, στη Μάλτα στα μαλτέτσικα και ούτω καθεξής. Οι ίδιοι οι παραγωγοί αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να έχουν διαφορετικές ετικέτες για διαφορετικές αγορές, αλλά να μπορούν να διαθέτουν το ίδιο προϊόν γενικά σε όλες τις αγορές. Και αν αυτό επιλέγει να κάνει ο παραγωγός, τότε δεν μπορούμε να τον εμποδίσουμε αλλά βέβαια να έχουμε απλούστευση η οποία να μας λέει ότι θα έχουμε μία γλώσσα που να ισχύει παντού, όχι, κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί βέβαια ε, θα πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ομιλούν ξένες γλώσσες, ε, τουλάχιστον αυτή είναι η πραγματικότητα ε, για ένα μέρος των ανθρώπων και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα λοιπόν μια τέτοια λύση δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Αυτό το ζήτημα για, κατά την άποψή μου δεν αποτελεί ζήτημα ουσιαστικά. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποφασίζουν οι παραγωγοί και θα πρέπει εκείνοι να δουν τι θέλουν να κάνουν. Ε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει μια διάταξη λοιπόν η οποία να ε, καταργεί τέτοιου είδου δικαιώματα. Τώρα σε ό,τι αφορά την ε, πρόταση που έχουμε εδώ, σε ό,τι αφορά την ε, ε, διάθεση στην αγορά νέων ε, κλωστοφαντουργικών υλών. Θα πρέπει εδώ να δούμε κατά πόσο θα ήταν δυνατό να έχουμε μια κοινή ονομασία για αυτές τις νέες είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς θα, πρόκειται, θα για ένα νέο προϊόν για το οποίο δεν θα χρειάζεται πλέον μετάφραση κατά συνέπεια. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Και νομίζω για τους ε, ε και για τους παραγωγούς, αλλά γνωρίζω πως υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν το επιθυμούν. Γιατί υπάρχουν κάποιοι α, πολίτες οι οποίοι επιθυμούν ακριβώς αυτή την διαφοροποίηση για λόγους διαφήμισης. Ε, δηλαδή η η χρήση των ε, γραμμάτων και η χρήση των διαφόρων λέξεων είναι διαφορετική ανάμεσα στις χώρες. Άρα λοιπόν για κάποιους μπορεί αυτή η πρόταση να μην είναι καν ενδιαφέρουσα, ακόμα και αν θα ήταν η πιο αποτελεσματική από άποψη απογραφειοκρατικοποίησης σε ό,τι αφορά την ε, διάθεση στην αγορά νέων ινών. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε, ώστε να αποφασίσουμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε και καλό θα ήταν να γίνει μια συζήτηση και με τους παραγωγούς και με εκείνους οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την ε, ε, ανάπτυξη, για την ε, δημιουργία νέων γλωσσοφαλωτικών ινόντος, ώστε να αποφύγουμε να μην ληφθούν υπόψη οι πολίτες στο πλαίσιο αυτό. Και κλείνοντας επιτρέψτε μου να πω ότι είναι απαραίτητη μια σαφής σήμανση των προϊόντων, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν ε, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω προϊόντα, εάν δηλαδή μπορούν να τα βάλουν για παράδειγμα στο πλυντήριο ή όχι. Αλλά ταυτόχρονα συμφωνώ με τους Σάντεμος και Σφάμπ ότι ε, το να έχουμε νέα εικονογράμματα νέα σύμβολα δηλαδή τα οποία θα συμπεριλάβουμε στι ετικέτε δεν θα ήταν τόσο χρήσιμο. Θα πρέπει δηλαδή να μείνουμε στα εικονογράμματα τα οποία είναι γνωστά σήμερα στου ε, πολίτε ε, και τα οποία γνωρίζουν πώ να χειριστούν. Το να έχουμε τώρα να δημιουργήσουμε, να εφεύρουμε νέα σύμβολα νομίζω πω δεν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ όλου ιδιαίτερα. Νομίζω ότι συνεισφέρατε όλοι με πάρα πολλέ παρεμβάσει. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο θέλει το λόγο. Αν όχι, τότε νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τουράου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει όσα άκουσε μέχρι στιγμή και ίσω να μα δώσει και ορισμένε ενδείξει για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι συζητήσει. Έχετε το λόγο. Αλλά προηγουμένω, συγγνώμη, ξέχασα να καλωσορίσω το Συμβούλιο, τον εκπρόσωπο ε, του Συμβουλίου, που ήταν πρόεδρο τη ομάδα εργασία. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ε, είστε εδώ με την ιδιότητα του παρατηρητή των εργασιών μας. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ γιατί μας δίνει την ευκαιρία να σας δώσουμε ορισμένε πληροφορίε και να κάνουμε και ορισμένα σχόλια σε όσον αφορά, όσον αφορά τη συζήτηση για τον κανονισμό αυτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι από τη δική μα ε, την οπτική γωνία ο συγκεκριμένο κανονισμό καταρτίστηκε στα πλαίσια του προγράμματο απλοποίηση και απλούστευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Στόχος είναι να ε, ε οι οδηγίες να οδηγήσουν σε ένα κανονισμό έτσι ώστε να έχουμε εξοικονόμηση χρόνου και για τους παραγωγούς και για τις εθνικές διοικήσεις και ταυτόχρονα να προωθήσουμε και επομένως μάλλον να προωθήσουμε την καινοτομία για το συμφέρον των καταναλωτών έτσι ώστε να έρθουν αυτέ οι νέες ίνε στην αγορά, ε, ώστε να τον πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Θα ήθελα να σας πω ότι Μα ανησυχεί ιδιαίτερα η συζήτηση για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού. Διότι αυτή τη στιγμή, όπω σα είπα, ε, πρόκειται για μια άσκηση απλούστευση τη νομοθεσία και όχι απόπειρα ρύθμιση για την κάλυψη όλων των πιθανοτήτων ετικετοθεσίας των κλωστοφαντουργικών προϊόντων, όλων των περιπτώσεων. Από ό,τι γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να αρχίσει η συζήτηση για την ετικετοθεσία των κλωστοφαντουργικών προϊόντων σε γενικό επίπεδο. Αλλά θέλουμε αυτός ο κανονισμός να περάσει ώστε να πιο γρήγορα, γιατί θα ωφεληθούν σαφώς όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και γιατί μας φοβίζει η συζήτηση για τον κανονισμό να ταυτιστεί με την ευρύτερη συζήτηση για, την, για τις ετικέτες των κλωστιφαντουργικών. Ενώ λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα οι συζητήσει με του εμπλεκόμενου και με του με τους ενδιαφερόμενου και με τα κράτη-μέλη στο παρελθόν για όλα αυτά τα διάφορα ζητήματα. Μας έχει δείξει ότι υπάρχει σαφής διάσταση απόψεων ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους και στα κράτη-μέλη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 υπέβαλε μία πρόταση για την ε, ε ετικετοθεσία όσον αφορά τη χώρα πλεύρευση των κροτοφαντουργικών προϊόντων. Αυτή η πρόταση από το 2005 βρίσκεται στο Συμβούλιο και μέχρι στιγμή τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η ετικέτα. συγκεκριμένη. Επίσης, εάν πρόκειται να συζητήσουμε τις άλλες ετικέτες, απαιτείται χρόνος. Βεβαίως, θέλουμε ιδιαίτερα να γίνει η συζήτηση αυτή. Αλλά όπως σας είπα, εκτός της συζήτησης, στα περιθώρια της συζήτησης για τον κανονισμό αυτό, γιατί σας είπα, θα ωφεληθούν όλοι, τα κρατημέλη, οι διοικήσεις, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Δηλαδή, να απλοποιήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία, μέσω του κανονισμού αυτού. Όπως σας είπα, ο μοναδικός στόχος είναι η απλοποίηση της νομοθεσίας. Για να αξιολογήσουμε όμως, για παράδειγμα, ζητήματα όπως ε, οι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, με το περιβάλλον, ε, με τις οδηγίες για το πλήσιμο, σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε μελέτες ε, αντικτύπου. Γιατί μόνο με αυτές τις μελέτες μπορούμε να πείσουμε τους ενδιαφερόμενους αλλά και τα κράτη-μέλη για τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μία ή η άλλη λύση. Και, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα καθυστερήσει και η έγκριση συγκεκριμένου κανονισμού ε, για δύο ή τρία χρόνια. Όσον αφορά το θέμα της τυποποίησης, ε, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε τον κανονισμό στο Συμβούλιο. Οι συζητήσεις διεξάγονται ιδιαίτερα καλά μέχρι στιγμής. Έχουμε ε, συγκεκριμένες λεπτομέρειες που θα εισάγουμε στο κείμενο, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει ε, ευρεία συνένεση, ευρεία συμφωνία για αλλαγή στα πλαίσια της διαδικασίας της επιτροπολογίας, για αλλαγή του παραρτήματος, που είναι το μεγαλύτερο. Μετά λοιπόν την έγκριση του κανονισμού θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά τις γλώσσες, οι υποχρεωτικές γλώσσες κάθε κράτους μέλους ε, οι αντιπροσωπείε των ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θέλουν και πάντα μας λένε ότι οι ετικέτε πρέπει να είναι στη γλώσσα τη συγκεκριμένη χώρα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να συμφωνήσουν. Είναι σαφέ αυτό. Βεβαίω, ε, είμαι στη διάθεσή σας να σας δώσω οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή εδώ ή οπουδήποτε αλλού. εάν θέλετε να έχετε περισσότερε ε, διασαφηνήσει. Βεβαίως μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να έρθετε σε επαφή μαζί μου και να σας δώσω ό,τι πληροφορίες θέλετε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σεράρε. Ευχαριστούμε για την προσφορά σας να συνεργαστείτε στενά με την Επιτροπή μας. Κύριε Μάντερς, θέλετε να κάνετε σχόλια, παρατηρήσεις... Και μετά θα κλείσουμε μιλώντας για το χρονοδιάγραμμα και την πρόταση που κάνατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Καταρχάς να σας πω ότι για την εσωτερική αγορά χρειαζόμαστε κανονισμούς μάλλον και όχι οδηγίες που μεταφέρονται σε, κάθε εθνική νομοθεσία και χαίρομαι που μιλάμε για κανονισμό εδώ. Είναι καλύτερο να έχουμε κανονισμούς αντί να έχουμε ένα patchwork ε, από οδηγίε, γιατί μεταφέρονται με διαφορετικό τρόπο στι εθνικές νομοθεσίες. Είπανε κάποιοι ότι δεν χρειαζόμαστε νέα στοιχεία. Ούτε εγώ τα χρειάζομαι. Είπα ότι πρέπει να απλουστεύσουμε τι ετικέτε ή δυνατόν. Δεν θέλουμε νέα στοιχεία, απλά απλούστευση ζητάμε. Και νέες μεθόδους ευρωπαϊκής τυποποίησης ε, των μεθόδων αδειοδότησης. Όλοι όσοι πήραν το λόγο, τον ίδιο στόχο έχουν. Το γνωρίζω και γι' αυτό ζήτησα ενημερωτικό σημείωμα. Εάν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές όλοι επιμένουν να έχουμε τις πληροφορίες στις 23 επίσημες γλώσσες, ας το κάνουν. Έτσι είναι η αγορά. Αλλά Θέλω να βασιστούμε στις γνώσεις που έχουμε για να πάρουμε την απόφαση. Γι' αυτό ζήτησα ενημέρωση, να ξέρουμε τι πιστεύουν οι παραγωγοί, τι πιστεύουν οι καταναλωτές για τα ζητήματα αυτά. χαίρομαι που οι συντονιστές ήδη αποφάσισαν την εκπόνηση αυτού του briefing paper, του ενημερωτικού σημειώματος και η Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει γιατί εδώ και χρόνια ασχολείται με το ζήτημα. με αυτή την ευρεία βάση πληροφοριών από πλευρά παραγωγών και καταναλωτών μπορούμε να πάρουμε ορθέ αποφάσει. Υπάρχει και μια σχέση με το REACH είπε στην συναδελφός μου ότι πρέπει να φροντίσουμε... Τι πώς το είπε ένα λεπτάκι... Τα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία αν πρόκειται για νέο, ε, νέα χημική ουσία, χρειάζεται συμμόρφωση με το ρίτσο τόσο ή άλλως. Ε, ας μην έχουμε επικαλύψεις, η απλούστευση είναι ο στόχος μας. Δεν θέλω καινούργια εικονογράμματα, δε, καινούργια συμβολάκια. Απλά μίλησα για το κόστος των πνευματικών δικαιωμάτων των ε, συμβόλων πάνω στην ετικέτα. Αν δεν είναι υπερβολικά υψηλό, να μείνουν ως έχουν. Και εγώ προτιμώ, γιατί ξέρουμε τι σημαίνουν ήδη. Αν δεν είναι υψηλό το κόστος, να κρατήσουμε τα ίδια σύμβολα. Αν προκύψει ότι ε, παρά είναι ακριβά, τότε να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικέ μέθοδοι. Συμφωνούμε δηλαδή ότι δεν πρέπει άδικα να αλλάξουν τα σύμβολα. Και αν έχετε περισσότερες πληροφορίες από αυτού, παρακαλώ να μου τις δώσετε. Θα είμαι ευγνώμων. Επίσης, να... ακούστηκε αν θα ήταν ενδιαφέρον να συνδυάσουμε αυτή τη δράση με επενδύσεις για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα αυτό είναι θέμα της, μάλλον, της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού. Όχι δικό μας. Το χρονοδιάγραμμα τώρα ο συνήθως είναι στενό το χρονοδιάγραμμα. Βλέπουμε τις προτεραιότητες κάθε φορά, αλλά άμα δείτε ότι είναι αδύνατο να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, ας το καθυστερήσουμε. Αν ήδη τώρα το καθυστερήσουμε, θα χρειαστεί και στο τέλος νέα καθυστέρηση, λόγω της ε, πίεσης ε, που έχουμε. Τις προτεραιότητες τις ιεραρχούμε βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Και μην ξεχνάτε ότι είναι επιτάπητο στο ζήτημα εδώ και χρόνια. Γι' αυτό είπα να προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο στην Ολομέλεια. Αλλά ε, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να είναι ισορροπημένη η πρόταση επί της οποίας θα ψηφίσουμε και αν χρειάζεται αναβολή ενός μήνα, δύο μηνών, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά εν γέννη πρότεινα να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και προσβλέπω με ανυπομονησία στη συνεργασία με τους ε, σκιώδεις εισηγητέ και όλους τους εμπλακόμενους. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε. Θα σας προτείνω κάτι για τα, την διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Έχουμε άλλη μία συνεδρίαση σε μία εβδομάδα, έτσι. Μία ημέρα. Προτείνω να σας δώσουμε μια σύντομη χρονοθυρίδα στο πρόγραμμα, όχι να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Απλά μόλις δείτε τους και συναντηθείτε με τους σκιώδεις, να μας ενημερώσετε και εμάς την επόμενη φορά για το χρονοδιάγραμμα και θα βοηθούσε αν εστιάζαμε λίγο τη συζήτηση στη συνολικότερη προσέγγιση. Όπως ε, μας υπενθύμισε ο κύριος Ζεράρο, είναι πρόταση απλοποίησης για τη σήμανση των φλωστόιφαντουργικών προϊόντων. Δεν έχει σχέση με ζητήματα ασφάλειας, ρίτς ε, κτλ. Ξέρω επίσης ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τα σήματα, τα οικολογικά και τα σήματα για τη φροντίδα των ρούχων. Και υπήρχε μια σχετική αμφιλεγόμενη πρόταση τη Επιτροπή. Η Επιτροπή μα μπορεί να δράξει την ευκαιρία και να εκπονήσει ξεχωριστή έκθεση πρωτοβουλία, ε, ιδέα πρωτοβουλία και να την προωθήσουμε εκ παραλίλου με αυτήν δεν κάνω πρόταση προς τα εκεί. Μη με παρανοήσετε. Απλά ε, προτείνω ε, να συμφωνήσετε με τους κοιόδης για τη συνολικότερη προσέγγιση που θα ακολουθήσετε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Γιατί έχει συγκεκριμένο πεδίο η πρόταση της ε, Επιτροπής ε, και αν το αποφασίσετε θα μείνετε σε αυτό μπορείτε να διαρθρώσετε και το χρονοδιάγραμμά σας αναλόγως. Όπως μας είπε ο κύριος Ζεράρα από την Επιτροπή, Πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να εξετάσουμε τις επιπτώσεις ενδεχόμενης επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της πρότασης. Κάθε φορά ε, ε, από την εμπειρία μας έτσι που κάναμε αυτό, ε, δαπανίσαμε πόρους γιατί χρειάζεται αξιολόγηση και λοιπά. Να άλλο ένα όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εσείς ε, κύριε Σιγητά θα πρέπει να μας πείτε ακριβώς τι θέλετε να έχει μέσα το briefing paper. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε τις σκέψεις σας ή η γραμματεια στη διάθεσή σας είναι απλά τι χρειάζεστε. Συζητήστε με τους ε, σκιώδεις και πείτε μας τι χρειάζεστε αλλά να μας δώσετε και μια ρεαλιστική προθεσμία και ε, υποψιάζομαι ότι ήδη υπάρχουν οι πληροφορίε που θέλετε. Απλά η γραμματεία θα τι ενοποιήσει και η Επιτροπή σίγουρα θα μα επικουρήσει. Απλά ε, αυτή τη βδομάδα σας παρακαλούμε, αν γίνεται, να συναντηθείτε με τους σκιώδεις, να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και θα σας δώσουμε λίγο χρόνο την τρίτη το πρωί την ερχόμενη εβδομάδα για να ενημερώσετε την Επιτροπή, να μας πείτε ποιο είναι το πρόγραμμα εργασιών σας. Έτσι θα βοηθηθούν όλοι νομίζω. Και ε, απευθύνομαι γενικότερα σε όλους τους συζητητές της Επιτροπής. Αυτό θα σας ζητάω κάθε φορά. Αν προγραμματίζουμε σωστά τις εργασίες μας, τελικά θα εργαζόμαστε και καλύτερα και θα έχουμε καλύτερες ευκαιρίες ε, να κάνουμε τη διαφορά. Ελπίζω να δεχτείτε την πρότασή μου. Βεβαίως, ε, με μεγάλη χαρά να τη δεχτώ. Απλά το σκέφτομαι διότι κάποια κράτη-μέλη, παρότι δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο μέσα στην πρόταση κανονισμού, κάποια κράτη-μέλη για τις ε, έχουν ε, κάνει υποχρεωτικέ τι ετικέτε για τη φροντίδα και το πλήσιμο των ρούχων, ενώ άλλα κράτη-μέλη όχι. Γι' αυτό μίλησα για επέκταση, ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογή, γιατί μπορεί να ε, παρουσιάζει ενδιαφέρον για την κοινωνία, για του καταναλωτέ και τη βιομηχανία. Πρόεδρος, ωραία. Ε, με αυτό το σχόλιο κλείνει το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο, κατάργηση των οδηγιών για τη... μεθόδους μέτρηση για την μετρολογία ε, και Ε, κυρία Βάις Γκέρμπερ έχει αναλάβει πάρα πολλές εκθέσεις στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν έχουμε τους σκιώδεις εδώ. Η κυρία Ρούλα βλέπω και πάλι θα πάρει το λόγο. Ο κύριος Μπιζόικ. Ο κύριος Κόζης Νίκε. Από τους σοσιαλιστές δεν είναι κανένας σκιώδης. Α, η κυρία Γκέπαρτ. Ωραία. Επίσης, ε, δεν... από τη γάμα δέλτα επιχειρήσεων ε, θα μιλήσει κανείς. Ο κύριος... Α, ο κύριος Αντούνες είναι εδώ πέρα που είναι επικεφαλής ε, του φακέλου. Ήρθε ο ίδιος, μάλιστα. Θα, θα σας ακούσουμε στη συνέχεια. Και από το Συμβούλιο δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε κάποιον. Νομίζω θα έρθει ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για αυτό το θέμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Η συγγήτρια, οι σκιώδεις θα πάρουν το λόγο και μετά οποιοδήποτε μέλος επιτροπής το επιθυμεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε σε αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για ένα θέμα αρκετά τεχνικό, αλλά παρόλα αυτά ενδιαφέρον. Ε, στην αρχή θεωρούσα ότι θα πρέπει να υπάρχει γενική συμφωνία καθώς η εν λόγω πρόταση θα οδηγήσει σε λιγότερη γραφειοκρατία στην Ευρώπη καθώς ε, η πρόταση αυτή προβλέπει την κατάργηση 8 διαφορετικών οδηγιών που ισχύουν σήμερα για τη μετρολογία και οι οποίες είναι βασικά απαρχαιωμένες και μπορούν να καταργηθούν αφού βέβαια εξεταστούν προσεκτικά. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον αυτό το θέμα γιατί πολλοί ε, μιλούν για μείωση της γραφειοκρατίας ε, και νομίζω πως ε, αυτός ο στόχος βρίσκει σύμφωνα σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Δηλαδή να καταργήσουμε διατάξεις κοινοτικέ οι οποίες είναι δυνατόν να καταργηθούν. Όμως, όμως είναι ενδιαφέρον το, το γεγονός ότι από την πλευρά διαφόρων κρατών μελών ή από την πλευρά διαφόρων φορέων να ε, υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες να υψώνονται κατά της κατάργησης. Γιατί λοιπόν ε, έχει νόημα αυτή η κατάργηση. Όλες αυτές οι οχτώ οδηγίες ε, αναφέρονται σε διάφορους τρόπους μέτρησης, για παράδειγμα όπως η μέτρηση της χωρητικότητας δεξαμενών σε πλοία, ε, όργανα μέτρηση σε ό,τι αφορά την πίεση του αέρα σε πίσω οχημάτων και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ορισμένα ίδια οργάνωτα, τα οποία χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο ε, τη σήμερα ημέρα. Ε, πολλά από αυτά ουσιαστικά έχουν ξεπεραστεί από την σύγχρονη τεχνολογία και ο αντίκτυπος από την κατάργηση αυτών των ειδικιών δεν θα είχε ιδιαίτερες επιπτώσεις καθώς ε, σε όλη την Ευρώπη η αγορά η οποία θίγεται από αυτό τον αντίκτυπο ανέρχεται μόνο στα 20 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες ε, κατασκευάζουν μόνο τέτοιου είδους απαρχαιωμένα ε, όργανα μέτρησης. Είχαμε την οδηγία για τα όργανα μέτρησης τη δεκαετία του 70 και τότε βέβαια κάτι τέτοιο είχε νόημα εκείνη την περίοδο καθώς θέλαμε να αποφύγουμε διαφορετικές διατάξεις σε αυτό το τομέα ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτές όμως οι τυποποιήσεις σήμερα έχουν πλέον ξεπεραστεί καθώς σε όλους αυτούς τους τομείς έχουν πλέον θεσπιστεί διεθνούς ε, εμβέλειας ε, πρότυπα. Ε, και κατά συνέπεια οι κοινοτικές διατάξεις δεν έχουν πλέον νόημα. Πολύ συχνά δηλαδή προβαίνουμε σε τέτοιου είδους τυποποιήσεις σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να οδηγήσουν σε κάποια στιγμή σε διεθνές παγκόσμιο επίπεδο. Ε, σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν ακριβώς ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία, έκλεισε αυτός ο κύκλος καθώς από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα έχουν πλέον θεσπιστεί διεθνή πρότυπα σε πολλούς ε, τομείς. Έχουμε κάνει ενδιαφέρουσες συζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ έχω να θέσω και κάποια ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα οποία θα ήθελα να διευκρινίσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν διεθνή πρότυπα σε όλους τους τομείς, δηλαδή που καλύπτουν και οι 8 οδηγίες και επίσης θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνονται από πλευρά ποιότητα στα ευρωπαϊκά πρότυπα, γιατί ακούσαμε πλευρά διαφόρων κρατών μελών ότι τα δικά μας, τα κοινοτικά δηλαδή πρότυπα υπερβαίνουν ποιοτικά τα διεθνή ε, πρότυπα και αυτό θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Ε, καθώς ε, βέβαια απόκληση από τα πρότυπα του ε, ΠΟΕ επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολόγηση για λόγους ασφαλείας και ούτω καθεξής. Επίσης, ερώτημα που θα πρέπει να φοβούμε. Θα πρέπει να φοβούμαστε με την κατάργηση αυτών των ειδηγιών σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Αυτό, για παράδειγμα, θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να θεσπίσουν εθνικού ε, εθνικά ε, πρότυπα, εθνική εμβέλεια ε, πρότυπα, κάτι το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί το στόχο μας. Ανάλογα λοιπόν με τι απαντήσει που θα λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να αναλογιστούμε ποια θα είναι η πρόταση που θα κάνουμε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτω ώστε πράγματι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώ αυτή την πρωτοβουλία για απογραφειοκρατικοποίηση. Κατά τη δική μου άποψη, δύο εναλλακτικέ ε, υπάρχουν ενώπιόν μα. Η μία, γιατί είναι βασικά αλληλοσυμπληρωματικέ αυτέ οι δύο, η μία να καταργήσουμε όλε αυτέ τι οδηγίε, ή εκείνε τις οδηγίες, δηλαδή δύο ή τρει, για τις οποίες πραγματικά δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη ύπαρξής τους, όπως για παράδειγμα η οδηγία για τα όργανα μέτρησης ή α, εκείνες οι οποίες ε, καλύπτουν στου οποίου υπάρχουν πράγματι διεθνή πρότυπα επαρχού τη ποιότητα. Η άλλη αναλλακτική είναι αυτοί που αφορά διατάξει, οι οποιες καλυπτουν τομεις στου οποιου υπαρχουν πραγματι διεθνη προτυπα υπαρκους ποιοτητα η αλλη εναλλακτικη ειναι αυτη που αφορα διαταξει οι οποιε ειναι αντιστοιχε ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το ε, εύρος ε, των αυλακιών, σε ό,τι αφορά την, τις συγκεκριμένες καλλιέργειες ή σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε διάφορες ουσίες στα δημητριακά. Όπως αναφέρθηκε και από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη θεωρούμε πως εκεί που υπάρχουν πραγματικά επαρκή ε, ποιοτικά ε, πρότυπα μπορούμε πράγματι να καταργήσουμε τις οδηγίες χωρίς να υπάρξει αντικατάστασή τους. Ακριβώς αυτό το χωρίς αντικατάσταση όμως είναι εκείνο που δημιουργεί κάποιες αντιδράσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι τα τελείως απαρχαιωμένα πρότυπα καταργούνται αλλά εάν θεωρηθεί απαραίτητο πως θα πρέπει να υπάρξει ε, ρύθμιση σε αυτούς τους τομείς θα μπορούσαμε να έχουμε ε, ρύθμισή τους μέσω της οδηγίας σε πλαίσιο του 2004 για τα αναμετρήσεις, ε, η οποία βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης και αυτό μας εξυπηρετεί πάρα πολύ γιατί πρόκειται για μια πραγματικά ευρύτατη οδηγία σε ό,τι αφορά τα όργανα της μέτρηση, η οποία έχει οθετηθεί μέσω του New Approach, της νέας προσέγγισης, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί και μελλοντικά πολύ εύκολα. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η πρότασή μου. Καταργούμε πράγματι αυτά τα παλιά πρότυπα τι παλιέ οδηγίε, αλλά εάν θεωρηθεί πω υπάρχει ανάγκη ρύθμιση των ελόγω τομέων από νέα πρότυπα, καθώ δεν θεωρούμε πω μα καλύπτουν επαρκώ τα διεθνή πρότυπα, ε, ε, τα ενσωματώνουμε μέσα στην ελόγω οδηγία πλαίσιο για τα ε, όργανα μέτρηση, για την οποία μάλιστα τρέχουν αυτή την περίοδο διαβουλεύσεις και αύριο θα υπάρξει μια συζήτηση στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν τα διάφορα κράτη-μέλη. Βέβαια θα υπάρξει περαιτέρω εξέταση, ε, δηλαδή θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν τα κράτη-μέλη και στο πλαίσιο της μελέτης αντικτύπου, η οποία θα εκπονηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ή εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης ε, ορισμένων κοινωτικών προτύπων, να το κάνουμε μέσω αυτής της οδηγίας σε πλαίσιο. αυτή η προσέγγιση είναι που προτείνεται. Δηλαδή, καταρχήν κατάργηση και αν υπάρξει ανάγκη ενσωμάτωση μέσα στην οδηγία πλαίσιο. Και αν δημιουργείται κάποιο νομικό κενό, ε, να λέμε ότι είναι δυνατή η κατάρχηση μόνο εφόσον πράγματι μπορεί να συμπεριληφθεί το εν λόγω πρότυπο μέσα στη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας σε πλαίσιο. Αυτές είναι οι δικές μου προτάσεις μετά από α, κάποιες πρώτες συζητήσεις οι οποίες έγιναν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες κατέδειξαν ότι υπάρχει ανοιχτή στάση διαλλακτική από την και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, Κλείνοντα, θα ήθελα να καλέσω όλου του συναδέλφου εδώ μέσα σε αυτή την προπαρασκευαστική αν θέλετε περίοδο των δύο εβδομάδων να απευθυνθούν σε μένα ή να ενδιαφέρονται ε, για να ενσωματώσω και δικέ του απόψει μέσα στην έκθεση και αν δεν τα καταφέρουμε να έχουμε από τον προτέρων μια έκθεση η οποία θα βρίσκει σύμφωνα σε όλες τις πολιτικές ομάδες τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε μια κοινή θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πούμε πώς ε, πράγματι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβήκαμε με συνέπεια σε μια πρωτοβουλία, σε μια προσπάθεια απογραφειοκρατικοποίησης, πράγμα το οποίο θα συνιστούσε επιτυχία για το Κοινοβούλιο. Εάν λοιπόν τα καταφέρουμε, ε, θα προτείνω ένα αρκετά σφιχτό ε, χρονοδιάγραμμα ε, σήμερα λοιπόν έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Στις 6 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, μας παρουσιάσει ε, την μελέτη εκτύπου σε ό,τι αφορά την υπάρχουσα οδηγία και μετά στις 16 Οκτωβρίου εγώ θα σας ε, παρουσιάσω τη δική μου έκθεση. Οπότε 3-4 Νοεμβρίου θα λάβει η χώρα επόμενη συζήτηση για αυτή την έκθεση στη δική μας Επιτροπή μετά. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Ε, παρότι βέβαια όπως σας είπα θα ήταν επιθεμητό να γνωρίζω εκ των προτέρων αυτές τις ε, προτάσεις ούτως ώστε να μπορέσω να τις ενσωματώσω. Μετά 16 Νοεμβρίου θα είχαμε επανεξέταση αυτών των amendments και 16 Νοεμβρίου ταυτόχρονα και υιοθέτηση ε, της έκθεσης μέσα στην Επιτροπή μας ώστε την ε, Ολομέλεια του Δεκεμβρίου να έχουμε πλέον έγκριση της έκθεσης. Αυτό σας λέω όμως ε, έχει ως ε, προϋπόθεση το να έχουμε να κινούμαστε λίγο πολύ προ την ίδια κατεύθυνση όλες τις πολιτικέ ομάδες. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, και ελπίζω πως θα έχω τη συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων. Σα ευχαριστώ για αυτή την τόσο συνολική ανάλυση του που βρισκόμαστε και νομίζω ότι ήσασταν και σαφέστατοι και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Επιβεβαιώνω ότι είχαμε προγραμματίσει να έχετε και ορισμένο χρόνο και την άλλη εβδομάδα για την συζήτηση για την ε, ε, αξιολόγηση αντίκτυπου. Τώρα, έχω του σκιώδε. Ε, ξεκινούμε με την κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε την κυρία Βάις για την ε, πολύ καλή παρουσίαση των απόψεων της ε, σε ό,τι αφορά αυτό το τομέα και την ε, παρουσίαση και των διαφόρων εναλλακτικών οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν με βάση τις δικές μας εργασίες. Νομίζω πως όλοι συμφωνούν όταν ο στόχος μας είναι η απογραφειοκρατικοποίηση, δηλαδή η κατάργηση διατάξεων οι οποίες είναι παροχημένες και αυτό είναι το σημείο στο οποίο θα ήθελα να βασιστώ κι εγώ. Θα ήθελα μάλιστα να υπενθυμίσω ένα ερώτημα το οποίο έχω θέσει δύο φορές ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θέτω για τρίτη φορά σήμερα καθώς δεν έχω λάβει σαφή απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διάφορες συζητήσεις που κάνουμε για αυτό το ζήτημα μας είπε ξανά και ξανά πως ε, ναι είναι δυνατό, μπορούμε να καταργήσουμε αυτές τις 8 οδηγίες, ναι είναι όλες τους παροχημένες, είναι όλες τους απαρχιωμένες, δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Αυτό ισχύει νομίζω για ένα τμήμα τους. Όμως ακούμε ταυτόχρονα ότι τα κράτη-μέλη ή καλύτερα ορισμένα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική άποψη και λένε όχι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτή δηλαδή τη συλλήτηνη κατάργηση. Και θέτω λοιπόν ξανά το ίδιο ερώτημα που έχω θέσει. Ποια είναι, πόσα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με αυτήν την ε, ομαδική κατάργηση των 8 οδηγιών και ποια είναι η αιτιολόγηση, ποια είναι τα επιχειρήματα των κρατών μελών όταν λένε ότι δεν συμφωνούν με την κατάργηση. Χρειάζομαι να λάβω αυτή την πληροφορία προτού μπορέσω να προβώ στη λήψη μια απόφασης. Ε, δεν μου, δεν μου φτάνει δηλαδή η εξήγηση που μου δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλες αυτές οι οδηγίες είναι παροχημένες και είναι περιτές. Ε, γιατί Προφανώ δεν ισχύει αυτό. Αν ισχύει, δεν θα υπήρχαν διαφωνίε από την πλευρά των κρατών μελών. Θέλω να ξέρω λοιπόν τι συμβαίνει εδώ, τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί βέβαια, αν προβούμε στην κατάργηση θα υπάρξει ένα νομικό κενό. Αυτή τη στιγμή έχουμε εναρμόνιση σε ό,τι αφορά τα ε, όργανα μέτρηση και ε, με την κατάργηση θα προκύψει ένα κενό το οποίο ενδεχομένω να ε, κληθούν να καλύψουν τα κράτη-μέλη μέσω εθνικών διατάξεων. Πράγμα που θα οδηγήσει και πάλι σε διαφοροποίηση εντός ε, της ενιαίας αγοράς. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του θα συνιστά, δηλαδή οι εθνικές διατάξεις θα συνιστούν ε, προστατευτισμό, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε. Άρα λοιπόν, ε, λέω σε εσά, κυρία Βαζικέρμπερ, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την κατάρριξη αυτών των ιδιών, θα πρέπει να εξετάσουμε τι θα κάνουμε και κατά συνέπεια δεν μπορώ να σας πω σήμερα τουλάχιστον ε, ω σκιώδη εισηγήτρια τη δική μου πολιτική ομάδα κατά πόσο μπορώ να συμφωνήσω με το δικό σα χρονοδιάγραμμα ή όχι. Σα λέω ότι χρειάζομαι, και να το κάνω αυτό, τι συγκεκριμένε πληροφορίε τι οποίε έχω ζητήσει ξανά και ξανά και τι οποίε δυστυχώ δεν έχω λάβει ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Μπουζό, έχει το λόγο. Θα μιλήσω στα ρουμανικά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Βάισπεργκερ για ε, την παρουσίαση του θέματος. Σε μεγάλο μέρος οι αρχές που ανέπτυξε δεν μας δημιουργούν κανένα πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν από την εισηγήτρια και αντίθετα πιστεύω ότι τα θέματα τα οποία ανέφερε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει όμως να πάρουμε μια απάντηση πριν ε, πάρουμε την ε, τελική μας απόφαση. Από ό,τι γνωρίζω, τα κράτη-μέλη ήδη μπόρεσαν να, να υιοθετήσουν τις δικές τους τεχνικές προδιαγραφές, ορισμένες. Και μετά από την θέση σε ισχύ αυτών των οδηγιών έκαναν προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη και την ε, ε, πρόοδο επί του θέματος σε διεθνές επίπεδο. Γνωρίζω εξάλλου ότι αυτές οι οδηγίες μιλούν για μεθόδους μέτρησης ε, που είναι ε, απαρχαιωμένες και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απλοποιεί το κοινοτικό κεκτημένο και να διευκολύνει το, ε, τη ζωή των επιχειρήσεων. Όμως θα πρέπει να αξιολογήσουμε κάθε μία από αυτές τις οδηγίες ξεχωριστά. Για παράδειγμα, η οδηγία σε σχέση με τους πίνακες Γνωρίζω ότι και σε άλλες οδηγίες ε, ε, αναφέρονται οι μετρήσεις αυτές. Άρα η κατάργηση ε, αυτών των οδηγιών δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αναφέρονται, τα, ε, αναφέρονται αυτά τα θέματα αλλού, σε άλλα κείμενα τα οποία θα ε, ισχύουν, εξακολουθήσουν να ισχύουν. Επίσης, να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι παραγωγοί χρησιμοποιούν τα διεθνή πρότυπα σε ε, εθελοντική βάση. Τα διεθνή πρότυπα τα οποία ε, χρησιμοποιούνται στο μέγιστο με το βαθμό στι άλλε χώρε. Άρα δεν χρειάζονται αυτέ οι οδηγίε επί τη ουσία. σα πω ότι η ομάδα μα υποστηρίζει την πρόταση τη Επιτροπή αλλά δεν μπορούμε να λάβουμε τελική απόφαση πριν πάρουμε, την, ε, πριν πάρουμε τις απαντήσεις στα θέματα τα οποία έχει τη θέση η συγκήτρια. Ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ κύριε Μπουσόη. Κύριε Ρούλα. Ευχαριστούμε για την ε, πολύ καλή προετοιμασία αυτού του ζητήματος από την κυρία Βάζη Κέρμπερ και να πω πως ε, θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσες τις ε, που μας παρουσιάσατε γιατί πάντα ακούγεται ε, ενδιαφέρουσα η μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά βέβαια το να μπαίνουν τελικά από το παράθυρο διατάξεις οι οποίες οδηγούν σε διαφοροποίηση, σε μείωση της εναρμόνισης δεν είναι κάτι το θετικό. Εάν λοιπόν έχουμε μια κατάργηση η οποία τελικά θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων εμποδίων σε εθνικό επίπεδο, ε, θα κάνουμε κάτι το οποίο ακριβώς δεν επιθυμούμε. Ε, άρα λοιπόν θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσες τις εναλλακτικέ που αναφέρατε, δηλαδή η πρόταση περί συμπερίληψης δηλαδή ορισμένων προτύπων στην ε, οδηγία IRD, δηλαδή για τα όργανα μέτρησης ε, προτύπων τα οποία θα καταργήσουμε στις άλλες οδηγίες. Και αναρωτιέμαι γιατί το, δεν το έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Δηλαδή να έχουμε μια τέτοια συνεργασία, αν θέλετε, εργασία σε διάφορα επίπεδα. Τελικά ποιο είναι το ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δείξει απλά στη δημοσιότητα ότι πράγματι να λαμβάνουμε μια πρωτοβουλία στον τομέα της μείωσης της γραφειοκρατίας ήθελε πραγματικά να κάνει κάτι. Γιατί σας λέω, γιατί υπάρχουν τόσες, φορέ, τόσες απόψεις που είναι κατά αυτής της ε, κατάρρυξης. Δεν θα μας ε, οδηγούσε σε μεγαλύτερη ε, συμφωνία, σε μεγαλύτερη συνένεση το να είχαμε ακριβώς συμπερίληψη των προτύπων αυτών στην οδηγία πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βάις Μπέρκερ, την εισηγήτρια, για την εισαγωγή που έκανε πιστεύω ότι θα υπάρξει συνένεση όσον αφορά τις αρχές αυτές, διότι ε, αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα απλοποίησης ε, της ε, νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Να σας παραπέμψω όμως το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης, οι ετικέτες στο κλωστιφοντουργικό τομέα. Και άλλη μια πρόταση λοιπόν προς την απλοποίηση. Αλλά εδώ μπορούμε να βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Όλοι ε, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το κλωστοφαντουργικό τομέα. Φοράμε ίδιοι τα, ε, τα προϊόντα αυτά, αλλά δεν είναι το ίδιο όσον αφορά τα θέματα μετρολογίας. Δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Βεβαίως και πρέπει να απλοποιήσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνω απόλυτα τις αντιρρήσεις που μπορεί να υπάρχουν, τα σχόλια τα οποία ακούσαμε από ορισμένους συναδέλφους πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χρονοδιάγραμμα. Και το καλύτερο θα ήταν να δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαγραφή ε, των ε, οδηγιών, αλλά με την προϋπόθεση αξιολόγησης διαγραφής μετά από πέντε χρόνια, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου για τι τόσο επικοδομητικέ παρατηρήσει. σα. Όλα αυτά δείχνουν ότι πράγματι είναι πολύ, πλοκό το ζήτημα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα. Και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να καλύψετε όλα αυτά τα ζητήματα σήμερα. Έχουμε προγραμματίσει και μια συζήτηση την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε ε, ορισμέ, ένα από τα πιο πρόσφατα ε, στοιχεία αξιολόγηση αντικτύπου κτλ. Θα σα δώσω το λόγο λοιπόν και στο που να αναφερθείτε και σε αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μπέργκερ για την τόσο καλή τη παρουσίαση. Πραγματικά ε, μας έκανε μια πολύ καλή παρουσίαση του προβλήματο μα έθεσε ορισμένε συγκεκριμένε ερωτήσει σε σχέση με την ποιότητα των διεθνών προτύπων. Από ότι, ε, ίσως από ό,τι γνωρίζετε, σε 7 από τι 8 περιπτώσει υπάρχουν διεθνή πρότυπα παρόμοιου ποιοτικού επίπεδου με αυτά τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή στι οδηγίε. Εκτό από το θέμα τη πίεση των ελαστικών. Εκεί δεν υπάρχει ακόμα ε, πρόταση, αλλά και εδώ ε, θα, θα δώσουμε εντολή και θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Τυποποίησης για να έχουμε πιο ενημερωμένα ε, πρότυπα. Έχουν γίνει εξελίξει στον τομέα και θα πρέπει να δούμε το ζήτημα. Και επί τη ευκαιρία σας λέω ότι από διάφορους διεθνείς φορείς ε, και από βιομηχανίες τρίτων χωρών βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για τις εξελίξεις ε, στο θέμα των προτύπων. Να Λαμβάνοντας υπόψη και την ποιότητα των υφιστάμενων προτύπων σε σχέση με το άλλο ε, ερώτημα, δηλαδή τι θα, τι θα συμβεί στην ιστορική αγορά μετά από τη διαγραφή, κοιτάξτε, καταρχήν δεν υπάρχει πρόβλημα. Η, αρχή τη αμοιβαία αναγνώριση υπάρχει. Τα περισσότερα από τα προϊόντα αυτά ε, ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και λειτουργούν όλα αυτά στην πράξη. Πρέπει να σα πω ότι ε, επανειλημμένα θέσαμε το ερώτημα και εμεί τα κράτη-μέλη για να δούμε κατά πόσον υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι εμπορικοί φραγμοί και στην βιομηχανία, στι μικρομεσαίε, στι μικρέ επιχειρήσει θέσαμε το ερώτημα, γιατί όσον αφορά και, ε, και, τα, και, την, ε, και τις 8 αυτές κατηγορίες προϊόντων, ε, μιλάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ε, μικρό μέρος λοιπόν της βιομηχανίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους εσωτερικούς φραγμούς και σε σχέση με το διεθνές εμπόριο. Θέσαμε το ερώτημα στα κράτη-μέλη και μέχρι στιγμής κανείς δεν, έκανε, ε, δεν ανέφερε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Πρόσφατα, προετοιμάζοντας την αναθεώρηση στην οποία αναφέρθηκε και η συγκεκριμένη η κυρία Ρούλα, προετοιμάζοντας λοιπόν την αναθεώρηση της ε, οδηγίας MID, Το κοινοβούλιο μα το ζήτησε και έγινε δεκτό και συμπεριλήφθηκε στην ίδια την οδηγία MID να υποβάλουμε έκθεση ε, μέχρι τον Απρίλιο του 2011 για να συμπεριλαμβάνει και κάποιες, ε, η πρόταση αυτή κάποιε δημοθετικέ ε, υποδείξει, εάν βέβαια δικαιολογούνται όλα αυτά. Τον περασμένο Ιούλιο ξαναθέσαμε το ερώτημα στα κράτη-μέλη να μα δώσουν οποιαδήποτε νέα στοιχεία έχουν για πιθανά εμπόδια στο εμπόριο που προκαλούνται που θα μπορούσαν να προκληθούν από την πρότασή μα για τη διαγραφή. Ακόμα και στι υφιστάμενε οδηγίε, με βάση τι υφιστάμενε οδηγίε, ε, να μα πούν τι γίνεται. Αύριο είναι η καταληκτική προθεσμία. Και μέχρι στιγμή δεν πήραμε καμία συγκεκριμένη απάντηση από κανένα κράτο μέλο. Άρα λοιπόν περιμένουμε και θα σα ενημερώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Όχι μόνο για την αξιολόγηση αντικτύπου τη δική μα πρόταση, όπω άλλωστε κάνουμε ε, και με κάθε πρόταση, αλλά θα σα ενημερώσουμε εάν στο μεταξύ κάποιο κράτο μέλο μα έχει δώσει κάποια νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω πρόταση. Και βεβαίω να σα πω ότι ήδη είπαμε στο Συμβούλιο ότι εάν υπάρχουν νέα στοιχεία, τότε εμεί θα είμαστε έτοιμοι να ε, λάβουμε, να εκμεταλλευτούμε την αναθεώρηση που προβλέπεται το 2011, να προβλέψουμε όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, ακόμα και μια ε, σύντομη αξιολόγηση του δικτύπου που φαίνεται έτοιμη του χρόνου. Θα είμαστε έτοιμοι λοιπόν να σας παρουσιάσουμε την έκθεση και εάν υπάρχουν τέτοια νέα στοιχεία, φυσικά θα συμπεριλάβουμε και κάποια νομοθετική πρόταση, εάν, θεωρηθούμε, εάν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο δικαιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, ε, το μέγεθος των εμποδίων και τον πιθανό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Και όλα τα άλλα στοιχεία, τα οποία πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας. Άρα πρέπει να σα πω ότι είναι κάπω παράξενο και κρίμα, αν μου επιτρέπετε, που η Προεδρία δεν είναι σήμερα εδώ. Ελπίζω να είναι παρούσα την επόμενη εβδομάδα. Γιατί όσον αφορά τα ερωτήματα τη κυρία Γκέπχαρτ, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία βεβαίω σε αυτό το δημόσιο έγγραφο. Το, το έγγραφο με τα ζητήματα κλειδιά που δημοσιεύσαμε τον Αύγουστο 2008. Ανάλογα με την οδηγία, 11 έως 15 κράτη-μέλη είναι υπέρ της διαγραφής και 6 έως 10 ε, προτιμούν μια κανονιστική προσέγγιση, ανάλογα με, το, με τα μέσα. Μιλώ για τις 8 αυτές ε, προτάσεις. Άρα βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα να σας πω και το εξή. Σε κάθε περίπτωση αλλάζουν και τα κράτη-μέλη. Είναι διαφορετικά τα επιχειρήματα Άρα τα πράγματα είναι τελείως συμπερδεμένα αυτή τη στιγμή, δεν είναι απλά. Θα θέλαμε να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις. Οι συζητήσεις σταμάτησαν στο τεχνικό επίπεδο, σε τεχνικό επίπεδο τον Απρίλιο αυτού του χρόνου, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Και περιμένουμε, από ό,τι έχουμε ακούσει, δεν φαίνεται να θεωρεί ότι είναι επίγον ζήτημα η Σουηδική Προεδρία. Όπω είπε η κυρία Ρούλε, βεβαίω δεν είναι επίγον ζήτημα γιατί δεν υπάρχουν προβλήματα στην αγορά. σε κανένα επίπεδο. Αλλά σκεφτήκαμε ότι στα πλαίσια της καλύτερης ε, ε, ρύθμισης και απλοποίησης νομοθεσίας είναι καλό ε, να βγάλουμε από τη μέση όλες αυτές τις οδηγίες που έτσι και παροχημένες και αποκαλύπτονται σε περισσότερες περιπτώσεις από τα διεθνή πρότυπα. Μέχρι στιγμής, όπως σας είπα, δεν πήραμε καμία, ε, κανένα συγκεκριμένο επιχείρημα. Δεν ακούσαμε να υπάρχουν συγκεκριμένα ε, προβλήματα, είτε σχέση με το εμπόριο, είτε σχέση με οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν τα κράτη-μέλη και θα μπορέσουμε να επανέλθουμε με ε, περισσότερε λεπτομέρειε. Πάντω σα πω ότι ε, τώρα εντάξει, μία μέρα πριν την προθεσμία να μην έχουμε πάρει κανένα σχόλιο. Δεν φαντάζομαι. Τέλο πάντων, μπορεί αύριο να έρθουν μαζικά τα στοιχεία αυτά. Την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε. Πάντω σα λέω ότι είμαστε απόλυτα ανοιχτοί και στην πρόταση τη ηγήτρια να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη συμφωνία με το Συμβούλιο. Αλλά και εδώ πρέπει να αντιδράσει το Συμβούλιο, ε, να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Δεν πρότειναν καμία νέα συζήτηση στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο πέρυσι του ζητήσαμε να ε, προωθήσουν το θέμα σε επίπεδο κορεπέρ. Αυτή τη στιγμή που σα είπα, οι συζητήσει έχουν φτάσει μόνο μέχρι, ε, μέχρι το επίπεδο των εμπειρογνωμόνων. Κάναμε συγκεκριμένη πρόταση να ανέβει στο επίπεδο Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Δεν, δεν συμφώνησαν κρίμα. Μακάρι να μπορέσουμε να πείσουμε την Προεδρία, να το προωθήσουμε το ζήτημα και να δούμε σε πολιτικό επίπεδο τι, ποια είναι τα επιχειρήματα. Ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε θέση λοιπόν να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο και βεβαίω είμαστε στη διάθεσή σα και στη διάθεση τη συγκήτρια και των σκιωδών και οποιονδήποτε μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όποιο θέλει περισσότερε λεπτομέρειε, είμαστε στη διάθεσή σα. Και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. ακόμα και αν κάνουμε μια παραπομπή σε περαιτέρω υιοθέτηση ή να το συνδέσουμε με την οδηγία MID. Δεν ξέρω γιατί η Προεδρία δεν θέλει να προωθήσουμε το θέμα. Ελπίζω με τη δική σας ενθάρρυνση και με την προσέγγιση της ηγητρίας, εάν συμφωνήσετε όλοι στο Κοινοβούλιο, να μπορέσουμε να ασκήσουμε έτσι κάποια ε, ήπια πίεση προς το Συμβούλιο, έτσι ώστε να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να λυθεί το ζήτημα. Ευχαριστώ. Well, σας ευχαριστούμε για την ειλικρίνειά σας ε, περιγράφοντας τις εξελίξεις ε, και αυτό που μας προσφέρατε να ακούσουμε μια πιο λεπτομερή παρουσίαση. Φυσικά θα το θέλουμε, θα φροντίσουμε να βρούμε και χρόνο. Βάσει αυτών που μας είπατε, ε, η δική μας Επιτροπή φέρει μεγάλη ευθύνη για το, τις μελλοντικές εξελίξεις. Δηλαδή, αν υπερψηφίσουμε αυτή την πρόταση, θα υποχρεώσουμε το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν κάτι και να προωθήσουν ε, το θέμα. Θέλετε να πείτε κάτι πριν δώσω το λόγο στην κυρία Βάις ε, Μπέργκερ. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι αντιλήφθηκα σωστά τα όσα μόλι τώρα μα είπε ο πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού είναι πολύ σημαντικό. Στην αρχή λοιπόν τη παρέμβασή του μα είπε Πώ μπορούμε πράγματι με ίση και τη συνείδησή μα να καταργήσουμε αυτέ τι οδηγίε γιατί έχουμε ήδη το σύστημα τη αμοιβαία αναγνώριση το οποίο ισχύει. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, οι κοινοί κανόνε αποτελούν εναρμόνιση ενώ αυτό το σύστημα το οποίο μα ανέφερε, δηλαδή τη αμοιβαία αναγνώριση, αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία. Άρα ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό εννοούσατε. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ναι, ναι, βασίζεται στην εθνική νομοθεσία, αλλά καλούμαστε να ακολουθήσουμε τα διεθνή πρότυπα, γιατί η εθνική νομοθεσία δεν μπορεί να ε, ε, δημιουργεί φράγμους ούτε στην εσωτερική αγορά, ούτε σε διεθνές επίπεδο. Οπότε προς το παρόν μπορούμε να εφαρμόσουμε ήδη την αμοιβαία αναγνώριση, γιατί δεν έχουμε εντοπίσει εμπορικά προβλήματα ε, σχετικά με αυτό. Οπότε ναι, απαντώ καταφατικά στην ερώτησή σας. Uh, Mrs. Gerber, Κυρία θα θέλατε να κλείσετε και να πούμε πως το χρονοδιάγραμμα το οποίο μας παρουσιάσατε και το οποίο έχει ήδη συζητηθεί με την γραμματεία φαίνεται λογικό. Για να έχουμε και κάποιο χρόνο για μια πλήρη συζήτηση την ερχόμενη εβδομάδα. Ο λόγος λοιπόν σε εσά, κύριε Βαστήρμπερ, για τα καταρκτικά σχόλια. Ναι, ε, πολύ σύντομα λοιπόν ε, πρωτού συνοψίσω τη συζήτηση, να πω το εξή. Σε ορισμένες διατάξεις, ε, σε ορισμένες οδηγίες, ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη μέτρηση της ε, περιεκτικότητας σε αλκοόλ, υπάρχουν πράγματι ήδη διατάξεις οι οποίες συμπίπτουν με αυτές και όπου υπάρχουν διεθνή πρότυπα, και αυτό μου αποτελούσε και για μένα έκπληξη, ε, πράγματι υπάρχει αντικατάσταση της, ε, των κοινοτικών προτύπων από διεθνή πρότυπα. Δηλαδή, εάν υπάρχουν εθνικά πρότυπα, τότε αυτά ε, ισχύουν κατ' εφαρμογή των διεθνών προτύπων. Άρα, δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις το επίπεδο, αν θέλετε, της εναρμόνισης έχει ανέλθει από το κοινοτικό δηλαδή στο διεθνές επίπεδο. και σας λέω ότι τα ε, κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δικαιούνται με βάση τις διατάξεις ε, του ΠΟΕ ε, να έχουν υψηλότερα πρότυπα μπορούν να το κάνουν μόνο για δικούς λόγους ασφάλειας, προστασίας υγείας και το καταξής. Άρα θα ήθελα να συνοψίσω την όλη συζήτηση που έγινε ως τώρα και την οποία βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, ότι όλοι συμφωνούν με το βασικό στόχο της μείωσης της γραφειοκρατίας και μπορούμε ακριβώς ε, σε ό,τι αφορά ορισμένε ε, οδηγίε να αποδεχτούμε την κατάργηση, αλλά, και εδώ συμφωνώ απολύτω μαζί σα, κυρία Γκέμπχαρτ, μετά από πολύ προσεκτική εξέταση για να δούμε πώ ακριβώ έχουν τα πράγματα εκεί, ούτω ώστε να πούμε ότι στις οδηγίες εκείνες όπου πράγματι έχουν καλυφθεί πλήρως οι διατάξει του από άλλο, χρειαζόμαστε την κατάργηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναμένουμε μόνο την αναθεώρηση, γιατί ορισμένες οδηγίες μπορούν και πρέπει ήδη να καταργηθούν. Στις υπόλοιπες τώρα οδηγίες και διατάξεις που θεωρούμε πως ε, πράγματι και λάβουμε σχετικά στοιχεία ότι χρειάζεται ε, η ύπαρξη περαιτέρω ρυθμίσεως, τότε οι εν λόγω αυτές ρυθμίσεις, τα εν λόγω πρότυπα να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης οδηγίας για τα όργανα μετρησής. Και αυτό δηλαδή να υπάρξει και εδώ να υπάρξει μια συμφωνία στο επίπεδο των ε, θεσμικών οργάνων. Ε, δηλαδή, ε, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μείνουμε στην κατάσταση που είχαμε τη δεκαετία του 1970. Δηλαδή, θα πρέπει να, πρέπει να Έχουμε συμπεριληψή του στην αναθεώρηση. Και εδώ ακριβώς είναι λίγο περίεργο το γεγονός ότι πράγματα, παραπονιούνται τα κράτη-μέλη ε, ε, ότι για παράδειγμα προβαίνουμε σε μια τέτοια κατάσταση και ούτω καθεξής, αλλά τελικά όταν κάνουμε κάτι και όταν αναφερόμαστε σε αναθεώρηση δεν ε, αναφέρεται κανείς από τα κράτη-μέλη σε αυτό. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει επιμονή από την πλευρά των κρατών μελών σε κάτι τέτοιο, εμεί θα πρέπει να προβούμε στην κατάργηση εκείνων των διών που θεωρούμε δεδομένων να γίνει. Και, α, βέβαια, θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σα, ώστε να έχουμε μια έκθεση στην οποία θα έχουν συμφωνήσει όσο γίνεται ε, πιο πολύ ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, παραγωγική μας συζήτηση και αναμένω με χαρά τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενέργεια που αφιερώνετε σε αυτή τη δουλειά και την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια πληρέστερη συζήτηση. Ε, προχωράμε στο επόμενο σημείο. Τώρα έχουμε την ε, δυνατότητα να εξετάσουμε τρεις γνωμοδοτήσεις που προτείνουμε ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τρεις πολύ σημαντικές προτάσεις που σχετίζονται με τα φαρμακευτικά σκευάσματα και τα ζητήματα στον τομέα αυτό που σχετίζονται με τους καταναλωτές. Προς ενημέρωση των νέων μελών της Επιτροπής ε, να ε, εξηγήσω ότι ως Επιτροπή έχουμε τη δυνατότητα να αποστέλουμε αυτές τις γνωμοδοτήσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση στην καθήλια αρμόδια Επιτροπή, δηλαδή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να ε, παρουσιάσουμε την κατάσταση από τη δική μας οπτική γωνία, ε, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τους ε, καταναλωτές και την εσωτερική αγορά. Οι συγητές έχουν σημαντική δουλειά να κάνουν εδώ ε, και σε συνεργασία με τους συζητητές από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για να λεφθούν δεόντως υπόψη οι δικές μας απόψεις και δεν είναι πάντοτε εύκολο, λέω, απευθυνόμενος στους συζητητές, αλλά άμα σας υποστηρίξουμε πλήρως θα τα καταφέρετε. Θα ήθελα να σας προτείνω μια ελαφριά αλλαγή στην τάξη, στη σειρά. Αν συμφωνεί ο κύριος Κορέια Ντεκάμπος, έχουμε δύο αλληλένδετες προτάσεις για την ενημέρωση ε, για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χρειάζονται η ιατρική συνταγή. Έχουμε ένα κανονισμό και τροποποίηση του κοινοτικού κώδικα στον τομέα αυτό. Ο κύριος Μπουζόη που ήταν εισηγητή στην προηγούμενη θητεία Ήδη έχει εκπονήσει έγγραφα εργασία και για τι δύο αυτέ προτάσει. Οι συντονιστέ αποφάσισαν να διορίσουν δύο εισηγητέ. Ο κύριο Μπουζόη ε, ευγενικά δέχτηκε να συνεργαστεί με έναν διαφορετικό ε, εισηγητή για να μοιραστούν και το φόρτο εργασία και ένα νέο μέλο, ο κύριο Κορέι Αντεκάμπο, αναλαμβάνει εισηγητή πρώτη φορά ε, στη θητή αυτό. Οπότε σα προτείνω το εξή. Εφόσον ο κύριο Μπουζόη γνωρίζει, κατέχει ήδη ε, το θέμα και έχει εκπονήσει και τα έγγραφα εργασία, κύριε Κορέι, αν συμφωνείτε να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Μπουζόη που θα μα παρουσιάσει και τι δύο προτάσει θα μας δώσει τη δική του άποψη και στη συνέχεια εσείς θα παρουσιάσετε τη δική σας πρόταση και θα κάνουμε από κοινού συζήτηση διότι να αλληλένδετα τα ζητήματα και ο κύριος Φιέλνερ από το ΕΛΚ είναι ο εισηγητής σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο κύριος Μπάστος είναι επίσης εδώ και θα φτάσουμε και σε εσά για να συζητήσουμε ε, τη δεύτερη πρόταση για τα παραποιημένα φάρμακα που αναλαμβάνει από τον προηγούμενο εισηγητή, τον κύριο Αγγελάκα, που είχε ε, αναλάβει τον ε, φάκελο στην προηγούμενη θητεία. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Μπουζόη, μετά τον κύριο Κορέι Ντεκάμπος και μετά τους σκιώδεις από όλες τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Κυρία Βάις Γκέρμπερ, συγγνώμη. Κάποιος από την Επιτροπή θα μας μιλήσει επίσης ε, για το θέμα, ο κύριος Φέρινγκ για τις δύο προτάσεις θα θέλαμε να τοποθετηθείτε. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Μπουζόη αρχικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήδη είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα στην τωρινή θητεία. Οπότε... Δεν χρειάζεται εγώ να μπω σε λεπτομέρειες. Απλά ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, περί τίνος πρόκειται και θα αποπειραθώ να σας προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συζητήσουν. Έχουμε ήδη συζητήσει με τους συμβούλους για την πολιτική της Επιτροπής μας για το χρονοδιάγραμμα. Επί της ουσίας, η κείμενη νομοθεσία, η οδηγία δηλαδή, ε, καταργεί την, ε, τις διαφημίσεις για το κοινό, για τα φάρμακα που χρειάζονται συνταγή. Ε, όμως, η κείμενη νομοθεσία δεν καλύπτει λεπτομερείς διατάξεις για την ενημέρωση για τα φάρμακα. Λέει μόνο ότι κάποια ανεπίσημη δραστηριότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως διαφήμιση καταργείται, απαγορεύεται. Ε, η κοινοτική νομοθεσία δεν παρεμποδίζει τα κράτη-μέλη από το να ορίσουν τη δική τους ε, προσέγγιση για αυτό το θέμα και τώρα η κατάσταση έχει ως εξής. Η φαρμακοβιομηχανία ε, που ε, πουλά το ίδιο φαρμακευτικό σκεύασμα σε πολλές διαφορετικές ε, χώρες μπορεί να δώσει κάποια ενημέρωση σε ορισμένα κράτη-μέλη αλλά όχι σε άλλα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί εναρμόνιση ε, και θέσπιση σαφών κανόνων σχετικά με το πώς οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται για φαρμακευτικά σκευάσματα που ε, απαιτούν ιατρική συνταγή. Είμαι πεπισμένος ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να επωφελούνται από τις ίδιες πληροφορίες υψηλής ποιότητας για τα φάρμακα. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι ακόμη και τώρα οι ασθενείς επιζητούν πληροφορίες διαφόρων ειδών, στο διαδίκτυο κυρίως. Και πολλές από αυτές τις πληροφορίες, ε, πώς να τις χαρακτηρίζω, δεν είναι επίσημες ε, και μπορεί να ταράξουν ε, τους ασθενείς, μπορεί να βλάψουν τους ασθενείς αυτές οι πληροφορίες γιατί δεν κατοχυρώνεται η ποιότητά τους για τέτοια φάρμακα που χρειάζονται ιατρική συνταγή. Επίσης είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να παραμείνει η απαγόρευση περί διαφήμισης για το κοινό για τέτοια συνταγογραφούμενα φάρμακα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε διαφημίσεις σε αυτό το τόσο ευαίσθητο τομέα. βάσει του μοντέλου των ΗΠΑ που σίγουρα είμαι εγώ πεπισμένος ότι στην κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ε, είναι υποφελής μπορούμε να αναβαθμίσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να θεσπίσουμε σαφείς κανόνες σχετικά με την παροχή πληροφοριών στους ασθενείς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε τους διάβλους πληροφόρησης. Ε, πρέπει να παραμείνει απαγόρευση ε, ε, παροχής πληροφοριών στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο για τα φάρμακα, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε την ανάπτυξη ιστοσελίδων και ειδικευμένων δημοσιευμάτων ιατρικού χαρακτήρα, από όπου θα ενημερώνονται οι ασθενείς. Επίσης, για τα άτομα με αναπηρίες και για τους ηλικιωμένους πρέπει να βρούμε ξεχωριστές λύσεις γιατί δεν μπορούν να έχουν την ίδια πρόσβαση στους ίδιους, ε, στις ίδιες μεθόδους πληροφόρηση. Το διαδίκτυο, παραδείγματο χάρη, δεν είναι μια εναλλακτική λύση για αυτούς, ε, γιατί πόσοι ηλικιωμένοι έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Πρέπει να βρούμε μια διαφορετική λύση ως εκ τούτου για να ε, ενημερώνεται και αυτοί. Επίσης, Πιστεύω ότι ε, οφείλουμε να θεσπίσουμε σαφείς κανόνες για την ενημέρωση στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή ήδη μας προτείνει κάποιους κανόνες Έχουμε ήδη κάποιες ε, προτάσεις για να βελτιώσουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν έχουμε σαφείς κανόνες με σύστημα πρώτερης αδειοδότησης και σύστημα επισήμων ιστοσελίδων όπου θα παρέχονται πληροφορίες για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν ουδέτερες ποιοτικές πληροφορίες για τα φάρμακα. Προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα τώρα ζητώ ε, τη συγκατάθεση των συναδέλφων ε, του κυρίου Μπάστος και του κυρίου Κορέια Αντεκάμπος. Προτείνω να εξεταστούν τα σχέδια γνωμοδοτήσεων στις 4 Νοεμβρίου, ε, να ορίσουμε καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες την 11η Νοεμβρίου να εξετάσουμε τις τροπολογίες την 1η Δεκεμβρίου και να ψηφίσουμε στις 2 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσει για τις εκθέσεις στις 25 Ιανουαρίου. Εάν λοιπόν όλα ε, πάνε καλά κατά το πρόγραμμα, το Φεβρουάριο ή αρχές Μαρτίου θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εφόσον είναι η τρίτη φορά που παρουσιάζω το θέμα, γι' αυτό το λόγο δεν ε, επισέρχομαι σε λεπτομέρειες. Αλλά αν οι συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις, ε, με μεγάλη χαρά θα τις απαντήσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ήσασταν σαφέστατος, ε, στη... Ε, είστε σαφέστατος μέσα στο έγγραφο εργασίας και στην παρουσίαση που κάνατε και ο κύριος Κορέια μάλλον το ίδιο χρονοδιάγραμμα θα μας προτείνει γιατί καθοδηγούμαστε από το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Κύριε Κορέια, ε, σας δίνω το λόγο. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνετε εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ευχαριστώ τον Κρίστιαν Μπουζόη αρχικά για όλη τη δουλειά που έχει κάνει στο φάκελο αυτό. Ας επανέλθουμε στο περιεχόμενο. Θα μιλήσω πορτογαλικά, λέει ο κύριος ε, Κορέντε Κάμπος, γιατί υπάρχει μετάφραση. Λοιπόν, συγχαίρω τον κύριο Μπουζόη και ήθελα να εξηγήσω το εξής. Ο στόχος αυτών των δύο νομοθετημάτων βασίζεται στην δημιουργία μιας δομής ενημέρωσης για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, για τις ενημέρωσης λοιπόν του κοινού για τα φάρμακα. Ποιος ε, είναι ο στόχος για την παροχή πληροφοριών ε, όσοι έχουν άδεια θέση σε εμπορία των φαρμάκων. Και γιατί πράγματα μιλάμε, γιατί προϊόντα μιλάμε, Μιλάμε για φάρμακα που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής ε, συνταγής ε, και ο, η πληθυσμιακή ομάδα στόχος, αν θέλει, είναι ολόκληρο το κοινό. Ε, ποιοι είναι οι περιορισμοί που δεχόμαστε. Πρώτον, να διατηρηθεί η απαγόρευση της άμεσης διαφήμισης προς τους καταναλωτές. Αυτή είναι η κανόνες του παιχνιδιού, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογεί αυτή την τροποποίηση του κανονισμού καταρχάς από την ανάγκη που υπάρχει για την εναρμόνιση της πρόσβασης πληροφορίας για τα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχει σχετική ασυμμετρία, όπως ακούσαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση. Δεύτερον, Υπάρχει η Γενική Αρχή των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων του Καταναλωτή ε, και η εξασφάλιση ισότητας των καταναλωτών χάρη στην ισότιμη ενημέρωση και τρίτον, ο παραγωγός είναι στην καλύτερη θέση, η βιομηχανία θέλει είναι στην καλύτερη ε, θέση να δώσει αξιόπιστες ε, πληροφορίες. Επίσης, έχουμε το περιεχόμενο του διαδικτύου που μας πλημμυρίζει και πρέπει να ρυθμίσουμε και πέμπτον, υπάρχουν αρχέ αρχές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο που έχουν την δυνατότητα, έχουν την αρμοδιότητα να ρυθμίσουν το περιεχόμενο ε, των πληροφοριών σε αυτές τις ιστοσελίδες. Όμως, όμως, η θέση του Συμβουλίου και δεν ξέρω αν ε, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Ε, στο Συμβούλιο ε, με την προηγούμενη Προεδρία η πλειοψηφία των κρατών μελών αντιτίθετο σφόδρα στην τροποποίηση του κανονισμού. γιατί ισχυρίζονται ότι ε, αυτή η επιχειρηματολογία δεν αιτιολογεί τροποποίηση του κανονισμού, ότι είναι δυσδιάκριτη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση και στη διαφήμιση. Επίσης, ε, θα μπορέσει κανείς να παρακάμπτει εύκολα ε, τον νέο κανονισμό. Επίσης λένε ότι οι μηχανισμοί ελέγχου των ρυθμιστικών αρχών συνεπάγονται μεγάλο κόστος και μεγάλο διοικητικό άχθος. Επίσης, οι σχέσεις ανάμεσα στους παρόχους επαγγελματίας του τομέα της υγείας και των ασθενών θα ε, ζημιωθεί ε, και τελικά θα ζημιωθεί η υγεία του ε, ασθενούς και τέλος αλλά εξίσου σημαντικό θα αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για τα, τα φάρμακα η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών στο Συμβουλίο στις 28 Μαΐου του 2009 ε, ισχυρίστηκε ότι η εν λόγω πρόταση δεν επαρκεί γιατί δεν κατοχυρώνει ε, καλή ποιότητα, για πληρότητα και αξιοπιστία για τις πληροφορίες πέραν ε, της διαφήμισης. Οπότε βρισκόμαστε προ ενός διλήμματος αν θέλετε θα σας πω τι κατά τη γνώμη μου σε αυτό το στάδιο μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για τις μελλοντικέ μας εργασίες. Ε, πρώτον, η αναθεώρηση του κανονισμού και της οδηγίας κατά τη γνώμη μου δεν είναι απαραίτητες. και ούτως ή άλλως μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις στις προτάσεις ε, της Επιτροπής. Επίσης, είναι απαραίτητη η άλλω μπορουμε του κοινού στις προτασεις τη επιτροπη επιση ειναι απαραιτητη η προσβαση του κοινου στις πληροφοριε και το ίδιο απαραίτητη είναι και η πρόσβαση ε, στις ε, πληροφορίε των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Και έχουμε καλά παραδείγματα συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία, στο ρυθμιστή, στη ρυθμιστική αρχή, στον πάροχο και στον ασθενή. Και πρέπει να προάγουμε τέτοιες καλέ πρακτικέ που ήδη έχουν σημειωθεί. όμω η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κατοχυρώνει ε, παρκή η ε, εχέγγυα για αυτή την ε, διάκριση που είπαμε ανάμεσα στην ενημέρωση και στην διαφήμιση. οπότε υπολείπεται μεγάλο έργο. Έχουμε δύο προτάσεις, δύο μάλλον από απόψεις εκ διαμέτρου αντίθετες. Ε, έχουμε από τη μία πλευρά το Συμβούλιο και από την άλλη όλους τους υπόλοιπους. Ε, όσοι ε, έχουν την εκτελεστική εξουσία χρησιμοποιούν επιχειρήματα που δεν μας πείθουν πάντοτε, αλλά δεν υπάρχει και επαρκής υποστήριξη για να διατηρηθεί ο κανονισμός ως έχει. Γι' αυτό το λόγο συμφωνώ προφανώς με το χρονοδιάγραμμα που μας ε, προτάθηκε για τις 4 Νοεμβρίου, αλλά να ρωτιέμαι, δεν θα ήταν καλύτερο να προτείνουμε μία έκτακτη συνεδρίαση μισή ημέρα, ούτω ώστε να ακούσουμε αυτέ τι εκδιαμέτρου αντίθετε απόψει ε, ε, και να τι εξετάσουμε. Αυτό προτείνω. Σα ευχαριστούμε. Uh, yes. well, um, thank you. Σας ευχαριστούμε για τις ε, τόσο ε, συνολικές απόψεις σας. Και ε, να κάνω ένα πρακτικό σχόλιο. Βεβαίως πρόκειται για γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν πρέπει να υπακούσουμε στο δικό τους χρονοδιάγραμμα. Γιατί πρέπει να τα προλάβουμε. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει ζήτημα να θέλουμε περισσότερο χρόνο, Πρέπει να το διαπραγματευτείτε και εσείς κύριε Μπουδόη με την ε, υπεύθυνη επί της ουσίας επιτροπή. Αν επιμένουν στην προθεσμία 25, 25 Ιανουαρίου, σαφώς είμαστε αναγκασμένοι να υπακούσουμε σε αυτούς τους περιορισμούς. Αυτή είναι η πρώτη γενική παρατήρηση. Και δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για γνωμοδότηση, Νομίζω ότι και εσεί και οι σκιώδει θα πρέπει να τα βρείτε και να δείτε πού μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά εμεί ω Επιτροπή. Με άλλα λόγια, δεν νομίζω ότι εμεί σίγουρα και απαραίτητα θέλουμε να διοργανώσουμε μια ευρεία κλίμακα ε, ακρόαση, για αυτό το πράξει η αρμόδια επί Επιτροπή. Εμείς πρέπει να περάσουμε τα βασικά μηνύματά μας. Και όσον αφορά τις νομοδοτήσεις, ε, έχουμε ε, συγκεκριμένα περιθώρια χώρου, τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και πρέπει να τα λάβετε και στις υπόψεις σας. Στα πλαίσια αυτά, αν εσείς και ο κύριος Μπουζόη με τους σκιώδεις μπορείτε να συζητήσετε τα ζητήματα και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και να αποφασίσετε μετά πώς θα προχωρήσουμε και μετά θα επανέλθουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα ικανοποιητικό χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα έχουν συμφωνήσει όλοι και θα μεγιστοποιήσουμε την προστέμενη αξία τη δική μα επιτροπή. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε και με τη δική μα την γνωμοδότηση. Έχω ορισμένου ομιλητέ. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι σκιώδη ή συμβάλλουν με τη γνώση του. Έχω λοιπόν το εξή στον κατάλογό μου και σα υπενθυμίζω ότι στην έκθεση τη κυρία Μπάστο σε, ε, σε λίγο. Fox, So I... Λοιπόν, ακούσατε το κατάλογο μιλητών. Να κλείσει εδώ ο κατάλογο των ομιλητών. Ωραία, κύριε Βάισμπέκερ πρώτα. Σα ευχαριστώ. Ε, μιλώ εξ ονόματο ε, του ΕΛΚ ω εισηγήτρια επί του θέματος. Βεβαίως να περιορίσουμε τη συζήτησή μας στα ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Και προφανώς ε, ε πρέπει να λάβουμε υπόψη τον τίτλο της Επιτροπής μας, εσωτερική αγορά και η προστασία των καταναλωτών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η πρόταση, αλλά έχει δίκιο ο πρόεδρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να δούμε πώ εμεί μπορούμε να βοηθήσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντο και να επηρεάσουμε τι εξελίξει εκεί. Είναι τόσο ευρύ το ζήτημα που απαιτεί συζήτηση επί των θεμελιωδών ζητημάτων. Και άρα, πρώτα απ' όλα να καλέσουμε ορισμένες οργανώσεις καταναλωτών γιατί οι πρώτες επαφές που είχα εγώ και οι πρώτες συζητήσεις για το θέμα έδειξαν ότι υπάρχει ανοιχτό πνεύμα. Τέλος αυτά θα πούμε αργότερα. Ευχαριστώ και τους δύο συγητές για την εξαιρετική τους παρουσίαση και να επαναλάβω κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Έχετε δίκιο κύριε Μπουσόη. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή καλύπτεται ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με απαγόρευση διαφήμισης. Το ζήτημα τη ενημέρωση όμω και τη πληροφόρηση ε, εξετάζεται ε, σε κάθε και χωριστά. Για παράδειγμα, στη Σουηδία υπάρχει περιγραφή στο ίντερνετ που εγκρίνεται από το, από το κράτος και που δίνει πληροφορίες στου καταναλωτές για τα φάρμακα, πώς πρέπει να χορηγούνται κτλ. Σε άλλα κράτη-μέλη όμως οι πολίτε δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου πληροφορίε. Ενώ θα έπρεπε κατά την άποψή μου. Υπό, ε, κατά την οπτική γωνία της προστασία των καταναλωτών. Δεν είναι πάντα δυνατόν να έχουμε τι σωστέ πληροφορίε. όταν ε, ε, ένας ασθενής να παίρνει πάντα τι σωστέ και τι κατάλληλε πληροφορίε. Και αυτή τη στιγμή Μπορεί κανεί να βρει στο διαδίκτυο πολλέ πληροφορίε. Αλλά όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών αυτών, τι να σα πω, είναι πολύ χαμηλή. Εγώ μίλησα με έναν γιατρό, ο οποίο μου είπε ότι περνάει πάρα πολύ χρόνο για να εξηγεί ε, στου ασθενεί ότι αυτά που έμαθαν από το διαδίκτυο είναι λάθο. Και ότι μπορεί να του βλάψουν αυτέ τι πληροφορίε. Καταλαβαίνετε ότι ένα ασθενή. Εάν ένα ασθενή ε, ε, δεν έχει πάρει τι σωστέ πληροφορίε, τότε απαιτείται πολύ χρόνο εκ μέρου του από, από γιατρό. Αν έχει σωστέ πληροφορίε, μειώνεται ο χρόνο ε, συνολικά. Και βεβαίω, ε, σε επίπεδο πρόληψη είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Βεβαίω, αυτό μπορεί να σημαίνει ε, περισσότερο προσπάθειε από περισσότερε προσπάθειε από το κράτο μέλο και σε επίπεδο προπολογισμού. Η προληπτική φύση όμω πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική προ του καταναλωτέ, έτσι ώστε να μπορούν να δράσουν προληπτικά. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θέλουμε πολίτε που να μπορούν να πούν τη γνώμη του και ασθενείς που να έχουν ε, δικαίωμα ε, επιλογής, να έχουν το δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους. Κάθε φορά που έχω ένα πρόβλημα, εγώ τι κάνω, προσπαθώ να ε, μάθω τι φάρμακα υπάρχουν το πρόβλημά μου, τι φάρμακα μπορώ να χρησιμοποιήσω, μπορώ να πάρω. Και ε, οι πληροφορίε αυτέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Μακάρι και εμεί στη Γερμανία να είχαμε το, το σύστημα τη Σουηδία. Το ζήτημα βέβαια είναι αρκετά αμφιλεγόμενο καθώς υπάρχουν και πολλές ε, ενώσεις προστασίας των καταναλωτών που φοβούνται τον αντίκτυπο ή μάλλον το γεγονό ότι θα μπορούσε να υπονομευθεί η απαγόρευση τη ε, διαφήμιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε και πολύ προσεκτικά το ζήτημα τη ιδιαιτερότητα των σχετικών ε, πληροφοριών. Η βάση μα είναι ε, προφανώ πάντα τα στοιχεία τα οποία μα διαβιβάζει η φαρμακομηχανία, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να γίνεται και μια επαλήθευση από την πλευρά των δημοσίων αρχών σε συνεργασία με τον τομέα της των ε, φαρμακείων και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να μην υπάρχει εδώ πρόβλημα. Ε, προς αυτές λοιπόν τις κατευθύνσεις μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς δηλαδή τις πτυχές της προστασίας του καταναλωτή και τις πτυχές του ελέγχου και της παρακολούθησης, της αποπτίας. Σημαντικό λοιπόν το ζήτημα της απαγόρευσης της διαβίβασης. Ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τους διάβλους ε, επικοινωνίας μέσω των οποίων διαβιβάζουμε αυτές τις πληροφορίες. Ε, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε μία ε, ποιοτική ιστοσελίδα η οποία θα ε, εμπίπτει σε πολύ αυστηρούς ελέγχους και προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκω ενδιαφέρουσα την πρόταση που κάνω συζητής, δηλαδή να χτίσουμε πάνω στα ήδη φυστάμενα συστήματα. Και παράδειγμα, στη Σουηδία υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα δικτυακή από την οποία έχουμε αποκομίσει θετικέ εμπειρίε. Ε, άρα λοιπόν θεωρώ πως ε, η εν λόγω πρόταση αποτελεί πρόοδο για τους ε, πολίτες μας και πραγματικά βρίσκω αρκετά περίεργο αυτό που μας λένε τα κράτη-μέλη ότι δηλαδή δεν χρειαζόμαστε διάταξη γιατί ούτε ή άλλως η σημερινή διάταξη περί απαγόρευσης της διαφήμισης καταστρατηγείται ήδη. Ε, δηλαδή ε, αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα ε, και είναι περίεργο το ότι μα το λένε αυτά τα κράτη-μέλη. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με... Δηλαδή στη κατάσταση είναι ότι έχουμε να κάνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο οι οποίε δεν επίπτουν σε κανένα έλεγχο. Άρα λοιπόν επίση θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ποιοτικέ πληροφορίε που διαβιβάζονται από τι φαρμακοβιομηχανίε και οι οποίε έχουν βαχθεί σε έλεγχο από ε, γιατρού. Ε, αυτές είναι οι δικές μας απόψεις και βέβαια θα ε, παρουσιάσουμε και τις δικές μας απόψεις και στις υπόλοιπες σαμβόντες ε, επιτροπές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχω τον κατάλογο των επόμενων μιλητών και πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Φόξ για την πρώτη του εμφάνιση στην Επιτροπή μα και ελπίζω να ακολουθήσουν και πολλέ ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κορέα και τον κύριο Μπουσόη για τι σαφεί εξηγήσει που μα έδωσαν για το ζήτημα αυτό. Ε, με τις οποί... Και συμφωνώ σε γενικέ γραμμέ με τι απόψεις του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών ε, σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, έτσι ώστε η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει ει όφελο των καταναλωτών. Υποστηρίζω την διατήρηση τη υφιστάμενη απαγόρευση για την άμεση ε, διαφήμιση προ τον καταναλωτή όσον αφορά τη, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Έχω όμω δύο ανησυχίε για την πρόταση και θέλω να τι τονίσω. Η πρώτη μου ανησυχία αφορά αυτή την συνολική προσέγγιση ε, ε, όσον αφορά όλες τις πληροφορίες. Δεν ξέρω λοιπόν, μήπως θα πρέπει να ε, δούμε το θέμα, για να, γιατί μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα γραφειοκρατική αυτή η προσέγγιση, δεδομένου του κινδύνου μη συμμόρφωσης. Ε, θα έλεγα, και ο οποίο είναι σχετικά μικρός, θα έλεγα να δούμε κατά πόσο είναι σωστή αυτή η συνολική προσέγγιση. Και δεύτερον, όσον αφορά ε, τους ελέγχους για τη διαφήμιση των ιατρικών προϊόντων. Ε, είναι ε, εθνικό το ζήτημα. Δεν ξέρω. Πρέπει να το ρυθμίσουμε σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το αφήσουμε στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Φόξ, είστε σκιώδης ε, για την ε, εκ μέρους ομάδας ECR. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρόιτοβα. Eh, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, στη σχέση με αυτά τα οποία ελέγξαν προηγουμένως, να σας πω τα περισσότερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν απαγόρευση και Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ορισμένε ανησυχίε όσον αφορά την εναρμόνιση. Να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη λειτουργούσε εδώ και πολύ καιρό και σε άλλα μόλι εισήχθη το μέτρο αυτό. Η διαφήμιση λοιπόν ε, έχει, ε, είναι διασυνορική φύσεως, έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Αλλά τέλος πάντων αυτά είναι θέματα που θα αποφασίσουν οι εμπειρογνώμονε, όχι οι πολιτικοί. Αυτό που πρέπει να πούμε εμείς γενικά είναι να πούμε ότι δεν μας αρέσει η διαφήμιση στον τομέα αυτό. Κάτι άλλο, όσον αφορά τι πληροφορίες που πρέπει να παίρνουν οι ασθενεί. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι Καταλαβαίνουμε ταυτόχρονα και συμφωνούμε ότι ο γιατρό είναι ο βασικό καθοδηγητή του ασθενού, αν θέλετε, και μπορεί να επιλέξει τον γιατρό του για να του έχει εμπιστοσύνη και να ακολουθεί τι συμβουλέ του. Ο γιατρό λοιπόν είναι υπεύθυνο για να δώσει πληροφορίε. Γιατί ένα πράγμα είναι η πληροφορία όσον αφορά τα φάρμακα που παίρνει ο ασθενή, αλλά ο ασθενή ε, χρειάζεται και άλλε πληροφορίε. Παράδειγμα, ε, οδηγίε διατροφή. Ε, Ένα ασθενή ο οποίο ε, παίρνει φαρμακευτική αγωγή πάντα πρέπει να καθοδηγείται από έναν εμπειρογνώμονα. Και εμείς θα πρέπει να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση του γεγονότο αυτού από του ασθενεί η συνειδητοποίηση είναι βασικό, έτσι ώστε να έχουμε ασθενείς καλά ενημερωμένους που να μπορούν να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Συμφωνώ με ορισμένα από τα ζητήματα που ανέφερε και η κυρία Βάισμπεργκερ, κυρίως όσον αφορά το θέμα της παροχής πληροφοριών, που έχουν δικαίωμα να παίρνουν οι ασθενείς, αλλά αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι σωστές. Άρα, τα φυλάδια που πρέπει να δίδονται στου ασθενεί. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να υπόκειται σε αυστηρού ελέγχου. Πρέπει να υπάρχουν οι υπεύθυνοι αυτών των εντύπων των ενημερωτικών. Και μερικέ φορέ. Ε, τι γίνεται με τα έντυπα αυτά. Πάντα πρέπει να τα έχουν στη διάθεση του ασθενεί. Τα παίρνουν μια φορά, μπορεί να τα χάσουν, μα να μπορεί να τα ξαναπάρει. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Τώρα να πω δύο λόγια. Προειδοποίηση, αν θέλετε. όσον αφορά τη διάκριση ανάμεσα στη διαφήμιση και στην ε, ενημέρωση. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προβεί σε ορισμούς. Γιατί το ζήτημα τελικά ανάγεται σε ζήτημα ορισμών. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι η διαφήμιση και τι είναι η παροχή πληροφοριών. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για ε, τους ορισμούς αυτού Ε, κοιτάξτε, τα συστήματα τελευταία ανάλυση συγκλίνουν και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για εναρμόνιση της ποιότητας. Ίσως λοιπόν, επειδή δεν βρισκόμαστε ακόμα στην εναρμόνιση, αυτό το πακέτο να μας ενθαρρύνει για να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Αλλά να έχουμε ε, πλήρως εναρμονισμένη, πλήρως εναρμονισμένη νομοθεσία δεν νομίζω. Σύμφωνα και με τις ειδίκες της Λισαβόνας, αυτό δεν είναι θέμα της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ορισμένα όρια εκ των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άννα. Έχει ε, αρκετή εμπειρία σε αυτό το τομέα και γι' αυτό ε, μα χαροποιεί το γεγονό ότι συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία. Πρωτού ζητήσουμε να πάρει το λόγο ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Παρβάνομα, την οποία καλωσορίζουμε και ω νόμιμο στην δική Επιτροπή. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ε, να συγχαρώ τους ε, κύριους Κορέα και Μπουσό ε, για το τάρος το οποίο έδειξαν το κουράγιο τους για να αναλάβουν αυτό το ζήτημα το οποίο βέβαια θα, θα γίνουν πολλές συζητήσεις είναι ένα από τα πλέον δύσκολα ζητήματα για να βρεθεί μια ισορροπία καθώς δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ των δύο διαφορετικών γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής των Συναρμόδιων διευθύνσεων. Γιατί αν το είχαν κάνει θα ήταν πολύ πιο εύκολο το έργο το δικό μας. Αλλά συμφωνώ με αυτό που είπατε, Πρόεδρε, ότι δηλαδή θα πρέπει να παραμείνουμε ε, μέσα στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων, της δικής μας Επιτροπής και να υποστηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Άρα λοιπόν, ε, σε ό,τι αφορά το δικό μας ε, τομέα, δηλαδή την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή, μιλάμε για καταναλωτές πρώτη φορά σε σχέση με τα φάρμακα αντί για ασθενείς. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε στη δική μας έκθεση γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελέσει ε, μια συγκεκριμένη και ε, αυτή προέδωσε σε ό,τι αφορά ε, τις εν λόγω υπηρεσίες ε, και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, ότι δηλαδή έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με δικαιώματα του ασθενούς, αλλά και με δικαιώματα του καταναλωτή. Δεύτερο σημείο. Είναι πολύ περίπλοκο να ευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ενημερωμένης επιλογής και κατευθυνόμενης επιλογής του ασθενούς. Εάν εγώ είμαι, εγώ είμαι ιατρός έτσι και έχω προφανώς συμφερόντων κατά κάποιο τρόπο. Αλλά εάν μπορεί ένας ασθενής να κάνει ενημερωμένη ε, επιλογή, τότε δεν χρειαζόμαστε όχι μόνο πληροφορίες, αλλά δεν χρειαζόμαστε γιατρούς. Άρα λοιπόν, ο κύριος λόγος λοιπόν για αυτή τη δυνατότητα πρόσβασης σε καλής ποιότητας πληροφορίες είναι να είναι έτοιμο για να λάβει τι κατευθύνσει τη οδηγία από την πλευρά του ιατρού ή ασθενή. Αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην δημιουργήσουμε ένα Φραγκενστάιν, όπω είπε χθε η κυρία Κούνεβα. Και θα σα δώσω δύο παραδείγματα γι' αυτό και θα κλείσω. Το πρώτο παράδειγμα αφορά την Πολωνία και είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, όπου έχουμε μια ομάδα επιστημόνων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προσποιούνται χωρίς να έχουν βάσιμα επιστημονικά στοιχεία ε, ισχυρίζονται λοιπόν ότι μια συγκεκριμένη ενσούλινη δημιουργεί καρκίνο. Και αυτή η φήμη έχει κυκλοφορήσει γενικά και προσπαθεί μάλιστα ασκούν πιέσει αυτή οι επιστήμονε αυτή η ομάδα να μην περιλαμβάνονται στο επίσημο συνταγολόγιο ε, συγκεκριμένε ένσουλε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, σε ό,τι αφορά αυτό που συμβαίνει τέτοιου είδου πληροφορίε. Από εκεί και μετά έχουμε το δεύτερο παράδειγμα μια ε, μιας ένωσης ε, ε, που έχει αποστείλει κάποια ερωτηματολόγηση σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση, σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίες υγεία από χώρα σε χώρα, χωρί να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. Αλλά δημιουργούν πολύ δηλαδή καθόλου ουδέτερε, καθόλου αμερόληπτε απόψει, χωρί κανένα να μπορεί να επαληθεύσει επιστημονικά αυτά τα στοιχεία. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Επιτροπή Ένδυοτο ώστε να έχουμε ε, καλέ τροπολογίε από την πλευρά μα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των πληροφοριών και του διάβλου ενημέρωση, επικοινωνία, αλλά και του αρμόδιε φορεί οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη διάδοση αυτών των πληροφοριών και θα μπορούν να προβάλλουν σε συγκεκριμένε μελέτε. Υπάρχει ε, μια επιστήμη η οποία ασχολείται ακριβώ με την με το έβρο των πληροφοριών και γι' αυτό θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει την γνωμοδότηση αυτών των αρμοδίων, δηλαδή που σχετίζονται με το ζήτημα του εύρου των ε, πληροφοριών, και θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παρμάνοβα. Και δεν θεωρούμε πω ε, έχετε στη δική σα περίπτωση μια σύγκρουση συμφερόντων ε, ίσα ίσα που είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το γεγονό ότι είστε γιατρό και εσείς και κυρία δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά αν θέλει ο κύριος Ρούτινγκ από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις να κάνει κάποια σχόλια, είναι εδώ. Ωραία, θα του δώσουμε το λόγο. Και μετά βέβαια θα δώσω το λόγο και στους κύριους Γορέα και Μπουζό για να κάνουμε κάποια καταληκτικά σχόλια για να κλείσουμε με αυτό το σημείο. Αλλά αν θέλει καταρχήν ε, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσης να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλες αυτές τις, ε, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έγιναν και θα θέλαμε απλώς να επενθυμίσουμε τρία σημεία τα οποία ήδη αναφέρθηκαν εδώ από τους ευρωβουλευτές. Ε, το πρώτο από αυτά είναι η δήλωση ότι η απαγόρευση της ε, διαφήμισης για φαρμακευτικές συνταγογραφούμενα φάρμακα παραμένει ω έχει. Δεν επιθυμούμε να υπάρχει τέτοια διαφήμιση. Αυτό έχει προβλεφθεί στην κοινωτική νομοθεσία και αυτό θα παραμείνει. Δεύτερο, εμείς θεωρούμε πως οι σημερινές ισχύουσες διατάξεις δεν ενδείκνυνται για την ε, διάθεση ποιοτικών ε, και ισορροπημένων αμερόληπτων πληροφοριών στον ε, ασθενή και ακριβώς επειδή θα πρέπει να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισορροπία σε αυτές τις πληροφορίες κάνουμε αυτές τις προτάσεις. Και τρίτον, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι προβλέπει ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα αυτή η Επιτροπή ώστε να μας υποστηρίξει σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Πέρα από αυτά τα τρία βασικά σημεία θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άλλα ακόμα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Ε, ε, πρώτον είναι ότι αυτή η πρόταση έχει οθετηθεί από το σύνολο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή έχει υπογραφεί από τους 27 επιτρόπους, έχει οθετηθεί από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από όλες μαζί τις υπηρεσίες της. Και δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω, επειδή προφανώς έχουν προκύψει εδώ κάποιες παρανοήσεις, σε ό,τι αφορά τις ε, πληροφορίες που συνοδεύουν ένα φαρμακευτικό σκεύασμα. Αποτελεί λοιπόν ε, υποχρέωση και κάθε τέτοιο ενημερωτικό φυλάδιο που συνοδεύει τη συσκευασία έχει εγκριθεί από την Εθνική Αρμόδια Αρχή ή από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας των Φαρμακών. Και αν υπάρχει έστω και ε, μία παραμικρή αλλαγή. Ακόμα και αν αλλάξει ο αριθμό του φαξ που αναφέρεται, θα πρέπει να υποβληθεί είτε στην EMEA ε είτε στην Εθνική Αρμόδια Αρχή και εκ νέου να υπάρξει έγκριση αυτής της, ε, αυτού του φυλαδίου. Και υπάρχει δηλαδή νέα απόφαση μετά ότι πράγματι εγκρίνεται αυτή η αλλαγή του αριθμού φαξ. Δηλαδή πιο αυστηρές ε, διατάξεις σε ό,τι αφορά την αλλαγή πληροφοριών δεν νομίζω πως υπάρχουν πουθενά άλλο από σε αυτό το τομέα. Παρόλα αυτά, διαπιστώνουμε σε σχέση με αυτή την πρόταση ότι σε πολλά κράτη-μέλη οι επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα. και μας λένε αυτά τα κράτη-μέλη ότι δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο γιατί κάτι τέτοιο α, έρχεται σε αντίθεση με το νομοθεσία περί απαγόρευσης τη διαφήμιση. Δηλαδή ένα από τα φυλάδια, τα συνοδευτικά τα οποία διαβάζονται πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο στον χώρο των ε, προϊόντων μα λένε ότι τελικά δεν είναι δυνατό να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο επειδή κάτι τέτοιο έρχεται σε σύγκρουση με τι διατάξει περί απαγόρευσης τη διαφήμιση. Θα πρέπει να γίνει κάτι εδώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπουζόη, κύριε Κορέα, θέλετε το λόγο. Ε, πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ σε επιτοπλίστων με τις απόψεις ε, που ακούσαμε. Βέβαια εύκολο δεν θα είναι να ε, εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη, διότι ε, υπάρχει αντίσταση στο Συμβουλίο, πόσο γνωρίζω. Πάντως, είμαι σίγουρος πως αυτό το θέμα θα πρέπει να το ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Φόξε αναρωτιέται πώ είναι καλύτερα να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη το θέμα. Μα έχουμε εσωτερική αγορά, έχουμε το ίδιο φάρμακο που κυκλοφορεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιείται στα 27 κράτη-μέλη. Δεν είναι δίκαιο σε κάποια κράτη οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλέ πληροφορίε ενώ σε άλλα να μην έχουν καθόλου πληροφόρηση. Άρα θα πρέπει να το χειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από αυτή την πλευρά θα υποστηρίξω την πρόταση της Επιτροπής. Ε, θα συζητήσω με τη συνάδελφό μου την κυρία Κουρβανοβά ε, σχετικά με την διάκριση ανάμεσα στην περιττή γραφειοκρατία και τους αυστηρούς ελέγχους. Φυσικά χρειάζονται αυστηρή ελέγχη να ξέρουμε τι συνιστά επίστημη στο σελίδα, τι ισχύει για, τα, για τις δημοσιευμένες πληροφορίες, αλλά αυτοί οι αυστηροί ελέγχοι δεν συνοδεύονται απαραίτητα από περιττή γραφειοκρατία που είναι επιζήμια ε, για τους παρόχους και για τους πολίτες τους ίδιους. Συμφωνώ επίσης ε, μαζί σας κύριε Χάρμπορ, ε, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή και μα ε, στι πτυχέ τη ιατρική αγορά, τη προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών. Δύσκολο βέβαια είναι να μην συζητήσουμε την πρόταση ω σύνολο. Έχουμε ε, γιατρού, ε, ε, και εγώ ίδιο ε, έχω σπουδάσει ιατρική και οι δύο συναδελφοί μου και Θα έρθω σε επαφή τη προσεχή ημέρα με τον κύριο Κορέα Ντεκάμπο ε, για να δούμε πώ γίνεται να αναβάλουμε κατά τη, ε, τη συζήτηση. Αλλά άμα γίνει τελική ψηφοφορία 25 Ιανουαρίου στην Επιτροπή, ε, στην αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε. Σα ευχαριστούμε κύριο Κορέα, τώρα. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ιδέες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και προκύπτουν από τη συζήτηση και ε, δείχνουν το βάθος του προβλήματος. Ε, η έννοια ε, της πληροφορίας. Δεν υπάρχει διχοτόμηση ανάμεσα στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση και στη διαφήμιση. Και στην διαφήμιση μπορεί να υπάρχουν καλές και κακές πληροφορίες. Και οι κακές πληροφορίες δεν σημαίνει ότι δίνονται εκ προθέσεως πάντοτε. Και κάτι άλλο που προκύπτει από τη συζήτηση είναι η ευαισθητοποίηση αυτών που ε, παρέχουν τις πληροφορίες. Ε, η αγορά βασίζεται στην ευθύνη των οικονομικών φορέων. Οτιδήποτε διευρύνει την ε, υποχρέωση μέρημνας για τους παρόχους πληροφοριών δεν σημαίνει περί τη γραφειοκρατία. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ε, θα πρέπει να αναλάβουν το ρόλο τους σε αυτό το τομέα. Δηλαδή αυτοί που παρέχουν τις πληροφορίες και ό,τι γίνεται για να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους είναι θετικό και είμαι σίγουρος ότι θα είναι χρήσιμες οι μελλοντικές μας εργασίες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές και όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ πλούσια και χρήσιμη ανταλλαγή προφοριών, ως συνήθως δηλαδή στην Επιτροπή μας. Και θα ήθελα να σας προτείνω το εξής για το χρονοδιάγραμμα. Ε, και ε, να σας πω κάποια πράγματα σχετικά με το πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ως Επιτροπή. Κύριε Μπουζέη, κύριε Κορέη, ε, μπορείτε να με τους κοιόδης της προσεχείς ημέρες και θα σας ε, δώσουμε λίγο χρόνο την επόμενη Τρίτη για να επιβεβαιώσετε απλά το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα καταλήξετε και ίσως να επιβεβαιώσετε και ποια θα είναι η προσέγγισή σας ε, για τα βασικά ζητήματα με τα οποία θέλετε να ασχοληθεί η Επιτροπή μας και οτιδήποτε άλλο έχετε να ζητήσετε, ενημερωτικά σημειώματα κτλ. Καλό θα ήταν να προγραμματίσετε τις εργασίες σας μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Θα προβλέψουμε λίγο χρόνο την επόμενη Τρίτη. Ε, στις 6 Οκτωβρίου για να μας ενημερώσετε. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Έχουμε καθυστερήσει, συνάδελφοι. Όχι ότι θέλω να περικόπτω τις συζητήσεις, απλά ε, θέλω να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 12.30. Προχωρώ σε άλλη μια σημαντική ε, γνωμοδότηση. Κύριε Μπάστος. Ε, θα μας μιλήσει για τα παραποιημένα φαρμακευτικά ε, σκευάσματα, πάλι αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ο κ. Αγγελάκας ε, είχε κάνει πολύ σημαντική δουλειά στην προηγούμενη θητεία και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάστος για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Δεν ξέρω αν έχουμε τους εσκιώδεις εδώ που θέλουν το λόγο, η κυρία Παλπανόβα από το Άλντε, η κυρία Βάιλερ, ε, η ΣΥΑΡ, τα υπόλοιπε πολιτικές ομάδες, ο κύριος Φόξ, ναι, η κυρία Ρούλα για τους Πρασίνους, ναι, ωραία. Θα ακούσουμε τους συναδέλφους που προανέφερα λοιπόν. Από πλευρά Επιτροπή, ο κύριο ε, Φίρινγκ ε, θα χειριστεί και αυτό το ζήτημα. Η κυρία Μπάστο. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να κάνω μια συνθετική παρουσίαση, παρότι είναι εξαιρετικά ευίσθητο αυτό το θέμα και ε, δεν μπορώ παρά να, να δώσω ένα σύντομο ιστορικό αυτής της πρώτης τροποποίησης της οδηγίας Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι όροι, προϋποθέσεις που ορίζουν την τροποποίηση. Ποια είναι η πρώτη. Αιτιολογείται η πρόταση τροποποίησης από το ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρεκβολικά αυξήθηκε ο αριθμός των ψευδεπίγραφων φαρμάκων ε, σε σχέση με την ταυτότητα και με την ιστορία, την προέλευση δηλαδή ε, του φαρμάκου. Επίσης, τα ψευδεπίγραφα ε, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα ε, ε, περιέχουν παραποιημένες ουσίες και μπορεί να μην περιέχουν και καμία ενεργή ουσία ή τουλάχιστον όχι στη σωστή δόση. Αυτό συνιστά σοβαρότατη απειλή για την δημόσια υγεία, για την ασφάλεια των ασθενών που ε, καταναλώνουν αυτά τα φάρμακα και απειλεί για την ίδια τη φαρμακοβιομηχανία. Ε, είναι μεγάλη πηγή ανησυχίας λοιπόν ε, για την κοινή γνώμη αλλά και για τους ιδεοπολιτικούς ηθήνοντες. Να σας πω επίσης ότι το προφίλ κινδύνου της παραποίησης ε, των φαρμάκων ε, τροποποιήθηκε. Ε, πώς άλλαξε ο αριθμός της παραποίησης των νέων φαρμάκων αυξάνεται και έτσι η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική και ακόμη πιο απειλητική. ως προς την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει το κοινό για την φαρμακοβιομηχανία και τους βασικότερους ε, οικονομικούς φορείς της. Υπάρχει επίσης το θέμα της διατροφικής ασφάλειας ε, που αντιμετωπίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεκαετία του 90 που σχετίζεται με αυτό το θέμα. Ε, να λοιπόν, Πρόεδρε, το ιστορικό υπόβαθρο ε, της προηγούμενης έκθεσης του κυρίου Αγγελάκα ένα έγγραφο εργασίας όπου εν γέννη συμπαρατασσόταν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούσε ότι η τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας θα έπρεπε να σχετίζεται όχι μόνο με τα αρχικά πρωτότυπα φάρμακα που καλύπτονται από το, την προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αλλά πρέπει να σχετίζεται και με τα γενώσιμα φάρμακα. Και επιθυμούσε να ε, επεκταθεί η πρόταση για να υπάρχει η δυνατότητα ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να ε, συνεργαστεί με χώρες όπως Κίνα και Ινδία ή ΙΠΑ για να έχουμε μια πιο αποτελεσματική εποπτεία σε αυτές τις χώρες. Τέλος. Για να σας εξηγήσω τι διακυβεύεται με την τροποποίηση της οδηγίας, θα έλεγα επίσης ότι η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών των κρατών μελών τάσσονται υπέρ της πρότασης τροποποίησης και ε, θα πρέπει κάποια σημεία να βελτιωθούν, να διευκρινιστούν. Υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις επιλώνες που πρέπει να επεξεργαστούμε κατά την τροποποίηση αυτής της οδηγίας. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι καλές πρακτικές πρακτικές παραγωγής ε, με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών. Παραδείγματος χάρη μπορώ να σας πω ότι κάποια κράτη-μέλη θέλουν το πεδίο της εφαρμογής της οδηγίας ε, να επεκταθεί και να καλύψει όλα τα φάρμακα. Άλλα πάλι κράτη-μέλη ε, δεν συμφωνούν και υπάρχουν προφανώς ε, και η στάθμιση του κόστους που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κάτι άλλο κρίσιμη σημασία και σημασίας, είναι η απουσία του ορισμού του ψευδεπίγραφου φαρμάκου. Εγώ πιστεύω, ε, επειδή είμαι σκιώδης εισηγήτρια, είμαι εισηγήτρια, συγγνώμη, για την εκνομοδότηση προς την καθήλια αρμόδια επιτροπή, δηλαδή την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι πέραν κάθε αμφιβολίας με πάσα διαφάνεια οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε ορισμό του ψευδεπίγραφου φαρμάκου κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε ορισμό λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνεισφορές όλων των φορέων αυτής της αλυσίδας παραγωγής των φαρμάκων τους διανομής ε, της φαρμακοβιομηχανίας, ε, ε, την εκπροσώπηση φαρμακοβιομηχανίας σε επίπεδο κράτους μέλους, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν για να καταλήξουμε σε έναν ορθό ορισμό των ψευδεπίγραμμων φαρμάκων. Κάτι άλλο, ένας άλλος πυλώνας που πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς κατά την επεξεργασία και την τροποποίηση οδηγία σχετίζεται ε, με την αλυσίδα διανομής ε, και τους οικονομικούς φορείς ε, που εμπλέκονται σε αυτή και τις καλές πρακτικές διανομής. Καλύπτει προφανώς τη χονδρική πώληση, την βάση των δεδομένων για τις καλές πρακτικές διανομής, την εποπτεία της επιθεωρήσης. Ε, και τις απαιτήσει για την εξαγωγή, ε, για τις ενεργές ουσίες, τις δραστικές ουσίες τώρα. Ε, ακούσαμε αμφιβολίες σχετικά με αυτή τη χρησιμότητα του καταλόγου των δραστικών ουσιών, γιατί 90% αυτών των ουσιών προέρχονται από τρίτες χώρες. Κυρίως από δύο χώρες, Ινδία και Κίνα. Τώρα, ε, πριν περάσω στο χρονοδιάγραμμα που προβλέψαμε για την παρουσίαση της γνωμοδότησής μας, θα ήθελα να σας πω ότι η κατάσταση με τη διαπραγματεύση έχει ως εξής. Όλα τα κράτη-μέλη ε, καλωσορίζουν την πρόταση και υπάρχει γενική ε, συμφωνία στην αρμόδια ομάδα εργασίας. Όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται ε, ε, ρυθμιστική, ρύθμιση για να, μην, ε, για να μειωθεί ο αριθμός των ψευδεπίγραφων φαρμακών και επίσης να βελτιώσουμε την ποιότητα των δραστικών ουσιών. Αυτό το ζήτημα είναι πολιτικού χαρακτήρα, αφορά επίσης στη δημόσια υγεία και ε, είναι επίγον το θέμα. Ε, έχει βασική σημασία. Πρέπει να ρυθμιστεί το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης, ε, έχουμε τις αρμόδιες αρχές, τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές που θα εφαρμόσουν τις νέες προτάσεις και αυτό είναι ευαίσθητο ζήτημα. Και εμείς ως πολιτικοί θύνοντες οφείλουμε να συνεισφέρουμε λαμβάνοντας υπόψη την άποψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και τέλος, για να ε, θα έλεγα συνοπτικά ότι προβλέπει το εξή εχνονοδιάγραμμα. Η συζήτηση ε, στην Ολομέλεια ε, προβλέπεται για τις 23 Φεβρουαρίου του 10. Πριν από αυτό θα γίνει παρουσίαση ενός του σχεδίου γνωμοδότησης την 1η Δεκεμβρίου και οι τροπολογίες έχουν καταλεκτική ημερομηνία την 11η Δεκεμβρίου. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, η συγγήτρια είναι από την Γκουέ Μαρίζα Ματίας λέγεται. Ήδη είχα την ευκαιρία να κάνω μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα μαζί της και μου είπε ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί μαζί μας, ούτως ώστε να ε, επιτύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε να επιτύχουμε ε, που ε, θα ε, βάλει την τελευταία πινελιά στις εργασίες μας, ε, ούτως ώστε να έχουμε μια σοβαρή εγγύηση για τους ασθενείς, αλλά και για την φαρμακοβιομηχανία και για την κοινή γνώμη γενικότερα. Θέλουμε να έχουμε ένα ασφαλές εργαλείο εργασίας, επίσης, για τους πολιτικούς ηθήνων. Σας ευχαριστώ. Thank you very much for that Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνολική εισαγωγή. Πριν καλέσω και τους άλλους ομιλητές, Κοιτάξτε, επειδή φοβάμαι ότι ήμασταν μάλλον φιλόδοξοι, προσπαθούσαμε να ομοδοποιήσουμε όλες αυτές τις προτάσεις και έχουμε μια δυσκολία. γιατί τις 12 παρατέταρτο καλέσαμε την Επιτροπή να μας κάνει μια παρουσίαση για, το, για, για τον πίνακα βαθμολογίας της Επιτροπής. Τώρα, έχουμε την κυρία Σαλντεμόζε και δεν θέλω να σας ε, στριμώξω ιδιαίτερα και δημιουργήσω προβλήματα. Ρωτώ, θα μπορούσατε όμως να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή και σε μια εβδομάδα να βρούμε λίγο χρόνο να, κάνουμε μια συνολική παρουσίαση. Θα συμφωνούσατε. Ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Θα ήθελα όμως να σας δώσω την ευκαιρία σήμερα να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση. Και θα σας δώσουμε το χρόνο σας σε μια εβδομάδα. Ε, επιτρέψτε μου λοιπόν να ζητήσω από τους σκιώδες γιατί η κυρία Μπαστό μα έκανε μία πληρέστατη παρουσίαση. Σα παρακαλώ, ε, απευθύνουμε στου κοιόδε, αν, αν θέλετε να είστε ε, σύντομοι. Λοιπόν, ξεκινούμε την κυρία Βάρντ. Κυρία Βάρντ. Ja, ναι, σε κάθε περίπτωση θα μπορούσα να είμαι πιο σύντομη από την προηγούμενη ομιλήτρια, δηλαδή την εισηγήτρια, γιατί βρισκόμαστε σε πλήρη συμφωνία σε ό,τι αφορά το στόχο μας. Και μάλλον συμφωνούμε, δηλαδή μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ως ε, προς ε, το ότι η εν λόγω πρόταση, το εν λόγω στοιχείο ε, όλων των πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει σε αυτό τον τομέα των φαρμάκων Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα, αλλά και πολύ δύσκολο και δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το πρόβλημα ε, και γιατί δεν είχε γίνει κάτι και πριν από τις εκλογές, αφού και το Συμβούλιο ε, συμφωνεί ότι θα πρέπει πράγματι να γίνουν εδώ βελτιώσεις. Άρα λοιπόν ε, μόνο σε ορισμένα επιμέρους σημεία δεν θα οδηγηθούμε σε συμφωνία. Σε καμία περίπτωση, και αυτό το λέω με σαφήνεια για τη δική μου πολιτική ομάδα, δεν θα πρέπει να αποδυναμωθεί ή να τροποποιηθεί δραστικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για το ε, ελάχιστο κοινό παρονομαστή σε ό,τι αφορά μια μελλοντική μεταρρύθμιση. Οπότε ε, θα θέλαμε να ξέρουμε ε, πότε θα λάβουμε και την σχετική έκθεση να μας πει δηλαδή κυρία Μπάστος, τόσο ώστε να έχουμε και κάποιο χρόνο για να κάνουμε κάποια συζήτηση από τη δική μας πλευρά στην πολιτική μας ομάδα. Ε, να πούμε πως οι τροπολογίες προτείνονται σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την πρόταση εκεί στο 5 για τους περισσότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις ε, και στις ίδιες τις μηχανίες να είναι δηλαδή ε, πιο διαφανή τα πορίσματα των διαφόρων επιθεωρήσεων πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι τώρα. Όλες λοιπόν αυτές οι προτάσεις είναι εξαιρετικές και ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ποια είναι, είναι, πώς προέκυψαν οι αριθμοί που έχουν συμπεριληφθεί εδώ στη μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά το κόστος και σε ό,τι αφορά και τις, ε, τα χρήματα τα οποία δεν θα δαπανηθούν, δηλαδή τις εξοικονομήσεις. Ε, ε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν υψηλέ προσδοκίε από την πλευρά του ευρέω ε, κοινού. Αλλά τι σημαίνει προσδοκίε, τελικά είναι μια αξίωσή του, δηλαδή να ελέγχονται εντελεχώς οποιαδήποτε συνταγογραφούμενα ή όχι φάρμακα κυκλοφορούν στην αγορά και ψευδεπίγραφα φάρμακα να υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρέ κυρώσει που να οδηγούν μέχρι και στην απαγόρευση τη διάθεσή του στην αγορά. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο εργαλείο, δεν ξέρω, ένα ψαλίδι για τον κήπο ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για φάρμακα δηλαδή, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ε, τομέα. Κλείνοντα λοιπόν να πω πω οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ καλέ, δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν, ίσω ένα ή δύο σημεία θα πρέπει να αποσαφινιστούν. Από εκεί και μετά αναμένουμε με χαρά τη συνεργασία και βέβαια θα θέλαμε να μας πείτε την ημερομηνία ε, κατά την οποία θα πρέπει να αναμένουμε την ειδική σας έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Παρβάνο. Κύριε Παρβάνο, πρόεδρε. Controversial.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 Ε, είναι προφανές ε, ότι είναι πολύ επιφανειακή συνεργασία ανάμεσα στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ επιχειρήσεων και ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ για αυτήν την πρόταση. Προκύπτει αυτό σαφώ, γιατί εδώ μιλάμε για διοικητικά μέτρα καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Μα στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ε, προσθέτει κύρο στο να καταπολεμεί κανεί την κυκλοφορία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Όλοι υπέρ θα είναι, έτσι δεν μπορεί να είναι κανεί κατά. Απλά δεν ξέρω αν ε, επιτιθέμεθα στο πρόβλημα από τη σωστή σκοπιά. Μιλάμε ε, για μια αγορά 40 δις, μιλάμε για την ανθρώπινη υγεία, μιλάμε για τον προϋπολογισμό, δηλαδή ε, για την έρευνα και την ανάπτυξη για την επόμενη περίοδο μέχρι το 2013. Εφόσον μιλάμε για μέτρα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, πρώτη φορά ε, στον κόσμο ίσως το εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία. Και στην πρόταση δεν γίνεται καμία διάκριση ανάμεσα στους νόμιμους και παράνομους διάβλους. Ε, 3 με 5% ε, παραποιημένων φαρμάκων μέσα στους νόμους ε, διάβλους που αυτή η πρώτα τροποποίησης οδηγίας. Το υπόλοιπο 95% ε, είναι, πρόκειται για παράνομη διακίνηση. Δεν μιλάμε, μιλάμε για διαδίκτυο και παράλληλο εμπόριο. Αυτή είναι η βασική δρόμη εισόδου στην αγορά των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Στο Κοινοβούλιο εμείς επιτρέψαμε την ε, πρόσβαση ε, στο εμπόριο αυτών των φαρμάκων μέσα από το διαδίκτυο και την παράλληλη αγορά. Για τα γενώσιμα φάρμακα τώρα, ε, μόνο 1% είναι ψευδεπίγραφα. 17% της αξίας των γενώσιμων είναι η βασική αγορά μόνο και τα υπόλοιπα είναι τα ethical products. Ε, σίγουρα κάποιο θα πληρώσει το τίμημα. Όπου και αν βάλουμε τι πληροφορίε, στο φυλάδιο του φαρμάκου κτλ., όποιο έλεγχο και αν ζητήσουμε από τη φαρμακοβιομηχανία, τελικά όλα αυτά θα μπουν μέσα στην τιμή του φαρμάκου και θα τα πληρώσει ο ασθενή. Εάν θέλουμε αυτά τα μέτρα ε, να γίνουν, να εφαρμοστούν για 70% των φαρμάκων, μόνο το 1%, ε, ενώ το 1% είναι ψευδεπίγραφα, δεν υπάρχει καλή σχέση κόστους-οφέλους. Είναι προφανές. Τώρα, αυστηρότερη έλεγχη έναντι της ε, βαρύτερη γραφειοκρατίας. Μα δεν είναι τρόπος αυτός για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στη γνωμοδότησή μα για τι δραστικέ ουσίε και ποιο φέρει την ευθύνη. Ε, σίγουρα αυτοί που παράγουν τα φάρμακα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τι ουσίε που χρησιμοποιούν και δεύτερον ευθύνη, ε, υπεύθυνη, πλήρω υπεύθυνη ε, για τα διοικητικά μέτρα που θα εφαρμόσουμε σε αυτούς γιατί γνωρίζουν ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία διοδότηση. Για την αξιολόγηση, όπω είπε και η κυρία Βάιλερ, Πρέπει να δούμε από πού προέρχονται αυτά τα δεδομένα και γιατί ε, μιλάμε μόνο για το κόστος και την εξοικονόμηση χρημάτων για τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά δεν αναφέρονται πουθενά οι ασθενεί. Ε, το κόστος για τους ασθενείς ε, δηλαδή, που εκείνοι θα φέρουν το μεγαλύτερο βάρος στο μέλλον. Εφόσον έχουμε την αξιολόγηση αντικτύπου σε τέτοιου είδους πρόταση, ας ξέρουμε ποιος θα πληρώσει τελικά το λογαριασμό. Και η προσωπική μου άποψη και η άποψη πολιτικής μου ομάδας είναι ότι για την επόμενη επιτροπή ε, θα ήταν λογικότερο να μπει στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ ή στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ καταναλωτών ε, το θέμα αυτό. Ε, ευχαριστούμε. Ήταν πολύ εύστοχα τα σχόλιά σας και θα τα λάβουμε υπόψη. Βέβαια υπάρχουν ζητήματα ε, υλοποίηση εφαρμογή είναι δυσκολότερα για τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν την εφαρμογή. σου. θα έπρεπε να το γράψουμε και αυτό στην γνωμοδότησή μας. Απλά είναι γνωμοδότηση, το θυμίζω έτσι. Δεν είμαστε εμεί ε, καθήλυνα αρμόδιοι για το φάκελο. Τώρα ας ακούσουμε τον κύριο Φόξ, την κυρία Ρότα, τον κύριο Σαρτόρη και την κυρία Ρούλα. Αν ναι, έχουμε χρόνο. Κύριος Φόξ. I will be brief. Um, I'm Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω τις προτάσει αυτέ και επίση υποστηρίζουμε, υποστηρίζω το γεγονό ότι δεν θέλει να διευρύνει και στα φάρμακα μέσω διαδικτύου. Αν γίνει στο μέλλον πολύ ωραία, αλλά δεν θέλω να συνδέσουμε αυτή την πρόταση με τη ρύθμιση του διαδικτύου. Επίση, με απασχολεί κάπω το συμπληρωματικό κόστο προ τη βιομηχανία, που τελικά θα το υποστούν οι φορολογούμενοι και οι πρέπει επίσης να δούμε το ζήτημα της ε, ε, Σαφώς είναι αντιπαραγωγικό η βιομηχανία ε, να μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες για την ασφάλεια, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να φροντίσουμε έτσι ώστε όταν γίνεται ανασυσκευασία των φαρμάκων, να πρέπει να υπάρχει απέτηση για ε, εφαρμογή των ίδιων μέτρων και όσον αφορά ε, αυτά τα ανασυσκευασμένα προϊόντα. Τέλος, δεν συμφωνώ ότι πρέπει να δώσουμε αρμοδιότητες σε έναν εξάρτητο οργανισμό για να επιθεωρεί ε, τις άδειες διανομής σε χοντρικό επίπεδο. Αυτό είναι θέμα που αφορά τις εθνικές αρχές. Σταματώ εδώ προς μη Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την αξιοθαύμαστη ε, περιεκτικότητα τον λόγο σας. Ελπίζω να είστε παράδειγμα και τους υπόλοιπους. Κύριε Ροϊτόβα, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μα. Θα περιοριστώ λοιπόν και εγώ σε δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε συνολικά το πρόβλημα αυτό. Πάντως, ε, ε, καλωσορίζω την εισαγωγή της παρακολούθησης και του ελέγχου των διανομέων πρέπει να φροντίσουμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία των ασθενών. Αν δηλαδή ε, αγοράζουν μέσω των επίσημων διάβλων τα φάρμακά τους, να είναι σίγουροι ότι 100% τα φάρμακά τους είναι σωστά. Δεύτερον, όσον αφορά τους ε, διάβλους, ε, πραγματικά είναι λυπηρό το χάος που υπάρχει. Έχουμε δει πόσο το Σέγγεν είναι ανίκανο να προβεί σε προστασία ε, από ε, τα πλαστά φάρμακα. Άρα, ό,τι αποτελεί αντικείμενο διανομής μέσω των επισήμων διάβλων, εκεί τουλάχιστον θα υπάρξει πρόοδος και η προστασία θα είναι καλή. Αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να εκπέμψουμε. Και επίση, και εγώ θέλω να απευθύνω έκκληση στο θέμα της συνειδητοποίηση, γιατί και αυτό είναι βασικό θέμα. Θα με ενδιαφέρει και εδώ έχω να κάνω μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Το πώς φαντάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μπορέσουμε να πετύχουμε βελτίωση των ελέγχων ή να το πω διαφορετικά. Πώς... Ε, τι γίνεται όταν έχουμε να κάνουμε με μεταφορά φαρμάκων τα οποία δεν αποτελούν το σήμανση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι ο κίνδυνος. Εδώ ανοίγει η πόρτα για πλαστά φάρμακα. Δηλαδή τι γίνεται. Περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πολλούνται εδώ, αλλά εδώ υπάρχει κίνδυνος ε, να διαρρεύσουν και στην ε, δική μας αγορά ε, πλαστά φάρμακα. Ευχαριστώ κύριε Σατόρη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω και η πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με την φυστάμενη κατάσταση. Αλλά το βήμα αυτό είναι μικρό και δειλό σε σχέση με τις απαιτήσει των Ευρωπαίων καταναλωτών που εμείς έχουμε καθήκον να υπερασπίσουμε. Εάν δεν επιδείξει το απαιτούμενο θάρρος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει να υποβάλει πρόταση που να προβλέπει την υποχρεωτική ανιχνευσιμότητα όλων ε, των συστατικών των φαρμάκων από τη στιγμή της παραγωγής μέχρι το σημείο πώλησης δεν πρόκειται να πετύχουμε διαφάνεια σε συγκεκριμένο τομέα. Επομένως δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, πράγμα το οποίο αποτελεί δικό μας καθήκον. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό ακόμα. Γνωρίζουμε ότι τα φάρμακα αποτελούνται από πολλέ ουσίες, δραστικές ουσίες, δραστικά συστατικά και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα, δεν ασκείται ακόμα πραγματικός έλεγχος όσον αφορά την ανεχνησιμότητα και όσον αφορά τον, ε, την επιθεώρηση των σημείων παραγωγής. Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορά ε, την πλαστοποίηση ε, και αυτή που είναι προφανής, αλλά αυτό το οποίο είναι πιο δύσκολο είναι ότι δεν γίνεται έλεγχος ε, των, ε, της διαδικασίας παραγωγής. Ακόμα και όσον αφορά τα φάρμακα τα γνήσια, τα οποία φτάνουν σωστά ε, μέσα από τους διάβλους διανομής. Αυτά, είναι προβλήματα, τα, αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζει η πρόταση, αλλά με δειλό τρόπο, όπως σας είπα, και όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Θέλετε να κάνετε μια σύντομη παρέμβαση, ε, να σας βολέψουμε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 Κατά τη δική μου άποψη, το ζήτημα των παραλλήλων εισαγωγών δεν συζητήθηκε επαρκώ. Ε, και επειδή ένα από του προηγούμενου ομιλητέ μα είπε ότι στο διαδίκτυο και στι παράλληλε εισαγωγέ έχουμε τι ε, περισσότερε απάντε, ε, θα συμφωνήσω με, το, με τα όσα είπα για το διαδίκτυο, αλλά όχι με τι παράλληλε εισαγωγέ, καθώ έχουμε εδώ πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά πρέπει να πω ότι ήταν ιδιαίτερα πλούσια η ανταλλαγή απόψεων, πολύ ενδιαφέρουσε οι παρεμβάσει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ε, πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν πρέπει να πείτε δύο λόγια και απευθύνομαι και στην εισηγήτρια. Πρέπει να συζητήσετε με του σκιώδει για να δείτε πού θα εστιάσουμε την προσοχή μα στην Επιτροπή. Ξέρω ότι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντο ενδιαφέρονται πολλοί συνάδελφοι. σω λοιπόν θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την ευρωγνωμοσύνη σα για να δούμε ποια είναι η προσθέμενη αξία, η πραγματικά προσθέμενη αξία τη Επιτροπή μα. Αυτά θα τα βρείτε μεταξύ σα. Κύριε Φίρινγκ, θέλετε να ε, δώσετε, κάνετε κάποια συγκεκριμένα σχόλια και να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα είμαι πολύ σύντομο. Πέντε πολύ σύντομε παρατηρήσει θα ήθελα να κάνω. Καταρχήν, το πεδίο αυτή τη πρόταση. Το ζήτημα των ψευδοφάρμακων φαρμάκων προφανώ και αφορά πολλού ε, κλάδου, ε, δηλαδή τον τηλεωνιακό κλάδο, τον ποινικό κλάδο, γενικά το ζήτημα των αγορών και ούτω καθεξής. Ε, αυτή η πρόταση εστιάζει τώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μια πτυχή, δηλαδή την αλυσίδα αν θέλετε πώληση ε, και την ε, παραγωγή των φαρμακευτικών συσκευασμάτων, ένα τομέα ο οποίος έχει τύχει επαρκούς εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό πεδίο ε, μέσω της οδηγίας 2083 ε, και αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να περιλάβουμε και άλλους ε, τομείς ούτως ώστε να διασφαλίσουμε αυτήν την αλυσίδα της διάθεσης στην αγορά ούτως ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνο ψευδεπίγραφων. Μιλάμε λοιπόν για ένα πολυδιάστατο ζήτημα και εδώ εμείς ασχολούμαστε με μία από αυτές τις πολλαπλέ διαστάσεις. Το δεύτερο σημείο, σε ό,τι αφορά το κόστος, πάντα κάνουμε εδώ μία σύγκριση μεταξύ του κόστους ε, της πρότασης και του κόστους ε, που θα προέκυπτε σε περίπτωση που δεν γινόταν μια πρόταση. Σε ό,τι αφορά το κόστος το οποίο θα προκύψει αν δεν υπάρξει πρόταση, ε, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να υπολογίζουμε το status quo, δηλαδή τα όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή. Αλλά το πρόβλημα είναι, είναι ότι δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσα ψευδεθήρα φάρμακα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην, ε, που διατίθενται στην αγορά, γιατί πρόκειται για έναν ε, τομέα ο οποίος είναι προφανώς ε, παράνομος ε, και γι' αυτό μόνο μέσω extrapolation και με ευρύτερε εκτιμήσεις μπορούμε να γνωρίζουμε περίπου τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη δική μας πρόταση, μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα νούμερα ως προς το κόστος Και προβήκαμε λοιπόν σε μια πρόταση σε ό,τι αφορά και ζητήματα στα οποία έχουμε σταθμίσει τον κίνδυνο. Δεν είπαμε για παράδειγμα ότι το σύμβολο ασφαλείας θα πρέπει να το έχουν όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ορισμένα φάρμακα που να το φέρουν με βάση μια αξιολόγηση που θα έχει γίνει ως προς ορισμένους παράγοντες ε, κινδύνου. Ακριβώς επειδή είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία ε, γενική ε, μεταχείριση των ε, φαρμάκων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το κατά πόσο θα πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένες διατάξεις ασφαλείας για επιμέρους φαρμακευτικά σκευάσματα ανάλογα με το τι αυτό σημαίνει βέβαια και για τον ασθενή ή για το ασφαλιστικό ταμείο ή το φορολογούμενο γενικά. Το τρίτο σημείο τι συμβαίνει στον χώρο διαμετακομιστικού εμπειρίου, δηλαδή του transit με τα φάρμακα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα καθώς αυτή τη στιγμή η σχετική νομοθεσία καλύπτει μόνο εκείνα τα φάρμακα τα οποία προορίζονται για διάθεση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αν έχουμε ένα εμπορευματοκιβώτιο το οποίο καταφθάνει στην Αμβέρσα ή κάπου αλλού ε, και μετά ε, μεταφορτώνεται για να συνεχίζει το ταξίδι του αλλού, οι δικέ μα οι μας διατάξεις δεν ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. Και το δικό μα σκεπτικό, και έτσι έχουμε διαμορφώσει αυτή την ε, πρότασή μας, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά την ποιότητα των λόγων φαρμάκων, ακόμα και στις περιπτώσει όπου τα λόγω φάρμακα ε, διέρχονται μόνο μέσα από την Ευρώπη, χωρίς δηλαδή να προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Ε, αυτό το λέω επειδή καταρχήν χρωστάμε τις, ε, το χρωστάμε στις χώρες εκείνες που παραλαμβάνουν αυτά τα φάρμακα γιατί πολύ συχνά πρόκειται για αναπτυσσόμενες χώρες και από την άλλη πλευρά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν εδώ κάποια, σε, ε, παραθυράκια, κάποιες πίσω πόρτες μέσα των οποίων δηλαδή παρότι προορίζονται για, για μετακομιστικό εμπόριο τέτοιες ε, αποστολές τελικά να φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Μία ακόμα παρατήρηση αυτή η πρόταση δεν καλύπτει ε, το λιανικό εμπόριο μέσω του διαδικτύου. Ε, γνωρίζουμε πως υπάρχουν εκατομμύρια ε, online φαρμακεία, δηλαδή μια σχετική έρευνα στο Google μας δίνει 22 εκατομμύρια αποτελέσματα και προφανώς έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους φαρμακευτικά σκευάσματα ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Η περίπτωση όπου κανείς ε, προσφέρει σε ένα, στο διαδίκτυο, μια τρίτη χώρα προσφέρει ε, στο διαδίκτυο τέτοια φάρμακα και τα ε, λαμβάνει κανείς χωρίς συνταγή και τα οποία αποστέλλονται σε μια απλή συσκευασία στον ε, ασθενή ε, είναι μια πρακτική η οποία ε, ουσιαστικά συνιστά παράβαση 15 διαφορετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μια αποτελεσματική εποπτεία αυτής της κατάστασης. Δηλαδή παρακολούθησης μίας-μίας των επιμέρους αποστολών από σκιώδεις αν θέλετε προμηθευτές οι οποίες βρίσκονται κάπου αλλού ε, ε, εντός ή εκτός της Ευρώπης. Και εκεί βέβαια υπάρχει πράγματι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος ο ασθενής τελικά να καταλήξει στο να ε, χρησιμοποιεί ψευδευτικά φάρμακα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι καλύφθηκαν μια σειρά από ορισμένα σημεία πολύ σημαντικά. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο η οδηγία αυτή έχει ενδιαφέρον. Κύριε Βάστος, θέλετε να επανέλθετε. Και επιβεβαιώνω το ότι συμφωνούμε με το χρονοδιάγραμμά σα, το οποίο βεβαίω και αυτό συνδέεται με την ψηφοφορία τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, που από ό,τι καταλάβαμε δεν θα γίνει πριν το Μάρτιο τον Απρίλιο. Άρα έχουμε άπλητο χρόνο. Θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να κλείσω τη συζήτηση. Θα μιλήσω επιγραμματικά. Το χρονοδιάγραμμα ήταν σαφέστατο. Υπάρχει μεγάλη διαφάνεια για την παρουσίαση της ε, γνωμοδότησης. 1η ε, Δεκεμβρίου είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, ε, γιατί χάρη σε αυτές είναι πιο προφανές το τι διακυβεύεται με αυτή την πρόταση. Ακούσαμε και την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με το διαδίκτυο, της παράλληλης εισαγωγής ε, ότι χρειάζεται και θα προβλεφθεί ένας αυξημένος έλεγχος. Έτσι καθησυχάζονται διάφορες ανησυχίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοι. Για την αξιολόγηση του αντικτύπου και του τελικού κόστους, η πρώτη τροποποίηση της οδηγίας απαριθμεί, ε, ε, συμπεριλαμβάνει ένα πλήρη κατάλογο ε, των αντικτύπων. Πάντως, στο τέλος ξέρουμε ποιος θα φέρει το βάρος, η φορολογούμενη και η φαρμακοβιομηχανία. Τέλος, θα ήθελα να πω, απευθυνόμενη στην Επιτροπή, ότι στην παρέμβαση του εκπροσώπου ε, δεν ε, έγινε καμία αναφορά στην επίκρισή μου. Δηλαδή ε, ότι δεν υπάρχει ο ορισμός του ψευδεπίγραφου φαρμάκου. Θα ήθελα ο εκπρόσωπος Επιτροπής που είναι εδώ μαζί μας να μου εξηγήσει γιατί δεν υπεραμείνεται αυτή της ιδέας αυστηρού ορισμού των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Σας ευχαριστώ. Okay, well... Πολύ ωραία. Θα δημοσιεύσουμε το χρονοδιάγραμμά σα. Πάντω επιβεβαιώνω αυτό που είπατε και πριν από λίγο, ότι μέχρι την 1η Δεκεμβρίου θα υπάρχει το σχέδιο γνωμοδότηση. Προφανώ οι σκιώδει θα συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια θα έχουμε μια προθεσμία για τροπολογίε 11 Σεπτεμβρίου και εξέταση τροπολογιών 25 Ιανουαρίου και 23 Φεβρουαρίου ψηφοφορία. Εάν θέλετε περαιτέρω ανταλλαγή απόψε, που νομίζω ότι ίσω θα ήταν σκόπιμο, θα μπορούσαμε να προβούμε σε αυτήν την ανταλλαγή σε μία από τι προσεχεί. Όχι την επόμενη εβδομάδα, αλλά μία από τι επόμενε. Ε, ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στο το χρονοδιάγραμμα και σας είπα ότι πρέπει να το δείτε το θέμα και με τις κοιόβε. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και τώρα, κυρία Σαλτεμόζε, ε, είχε την ευγενή καλοσύνη να συμφωνήσει να συζητήσουμε το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα. Μήπω θέλετε απλά και μόνο να κάνετε μια σύντομη εισαγωγή τώρα, να κάνετε μια παρουσίαση, ή δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω, θέλω να σα δώσω το λόγο, αλλά ε, ότι εσεί αποφασίζετε. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή τη στιγμή μια εισαγωγή στη συζήτηση. Θα ήθελα τουλάχιστον πέντε λεπτά. Και αν θέλετε την επόμενη εβδομάδα να μας δώσετε τον κατάλληλο χρόνο, τότε καλύτερα περιμένουμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ζητώ για άλλη μια φορά στη γνώμη. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να το συζητήσουμε με την άνεσή μα την επόμενη εβδομάδα παρά να το συζητήσουμε πάρα πολύ βιαστικά. Και ελπίζω, ε, και κοιτάξτε, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και του σκιώδει, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε όλο το θέμα. Σα υπενθυμίζω σε όλου ότι στην περασμένη Κοινοβούλια συζητήσαμε το θέμα αυτό και καταλήξαμε σε μια γνωμοδότηση που δεν τη χρησιμοποίησε ποτέ η Επιτροπή Περιβάλλοντο, γιατί ε, δεν προχώρησε η ψηφοφορία. Άρα λοιπόν έχουμε στοιχεία για να δουλέψουμε. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα η πρώτη ε, ε, ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας επί νέας θητείας. Πρόκειται για το πίνακα βαθμολογίας από το σκόρμπορ της εσωτερικής αγοράς. Uh, λοιπόν, ε, βλέπω ότι η κυρία Μπράμπτον είναι εδώ, η οποία και θα πει δύο λόγια. Και στο μεταξύ να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι εδώ έχουμε αυτές τις νέες αίθουσε που υποτίθεται ότι έχουν ε, όλα τα τεχνολογικά μέσα. Οι οθόνες είναι τόσες μικρές ε, για τις διαφάνειες που είναι σχεδόν άχρηστες. Τι κάναμε λοιπόν. Ε, θεωρητικά πήρατε όλοι αντίγραφα των διαφανειών. Άρα λοιπόν πάμε στην παλιά καλή τεχνολογία με τα χαρτιά που δεν είναι και φιλικές προς το περιβάλλον Φροντίστε όμως όλοι να πάρετε αντίγραφα των διαφανειών. Θα μιλήσουμε για δύο σχέδια. Το ένα είναι οι υποδείξεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, του Ιουνίου για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεύτερον θα μιλήσουμε την πίνακα βαθμολογίας της εσωτερικής αγοράς. Οι συντονιστές συμφώνησαν να έχουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για τα ζητήματα αυτά που αφορούν τον πίνακα βαθμολογίας εσωτερικής αγοράς και ρωτήσω ιδιαίτερα την κυρία Τούν στην Επιτροπή, είναι νέο μέλος και διορίστηκε εισηγήτρια για την πρόταση αυτή. Δεν ξέρω ποιο θέλει το λόγο. Μήπω θέλετε πρώτα να ακούσετε την παρουσίαση και μετά να σχολιάσετε. Ό,τι προτιμάτε. Κυρία Τούν, εσεί αποφασίζετε. <clears throat> Maybe the presentation first. Ίσως πρώτα να ακούσουμε την παρουσίαση. You agree. Okay. Όχι, εγώ ε, συμφωνώ. Απλά δεν ήθελα να νομίσετε ότι σας αφήνουμε έξω από τη συζήτηση. Ωραία. Θα τοποθετηθεί η κυρία Τούν μετά από την παρουσίαση της Επιτροπής. Και αν έχουμε το χρόνο, θα καλέσω και του χειώδει. Αλλά πρόκειται για μια συζήτηση προσανατολισμού, για να ξεκινήσουμε τη συνολική διαδικασία ε, τη έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Κυρία Βάντερ, θα αρχίσετε. Σας καλωσορίζω με μεγάλη μου χαρά στην Επιτροπή μας. Έχετε το σημαντικό ρόλο του να είστε επικεφαλής ε, ε της συγκεκριμένης ε, ε, μονάδας, συγκεκριμένου τμήματος, στη Γενική Διευθυντική Αγορά. Και με μεγάλη μου χαρά σα δίνω το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα σας παρουσιάσω τις συστάσεις της Επιτροπής για την βελτίωση της λειτουργίας ιστορικής αγοράς και η συνάδελφός μου, η κυρία Καζάης, θα σχολιάσει ε, τον πίνακα βαθμολογίας ε, της ιστορικής αγοράς. Και για τις δύο παρουσιάσεις, ε, πήρατε τις διαφάνειες σε χαρτί. Ε, οι διαφάνειε ε, αναφέρονται λεπτομερώ στη σύσταση. Εγώ θα σχολιάσω με δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, γιατί εκδώσαμε τι συστάσει αυτέ. Διότι, όπω όλοι γνωρίζουμε, δεν ε, λειτουργεί όσο καλά θα έπρεπε η εσωτερική αγορά και στη σημερινή περίοδο κρίση επήγει να συντονίσουμε τι προσπαθίε μα έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση προ όφελο και των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. Επίση, όλα αυτά ακολουθούν την αναθεώρηση της ενιαίας αγοράς ε, που ανεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο χρόνια και ε, τότε εξέδωσε και ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου ζητούσε από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή να μειώσουν το χάσμα ανάμεσα ε, στις δυνατότητες και στην πραγματικότητα που χαρακτηρίζει την εσωτερική αγορά, την ενιαία αγορά. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε να απαντήσουμε απευθεία σε αυτές τις ανησυχίες και ως Επιτροπή και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σύσταση αποτελείται από 10 επιμέρους συστάσεις που αφορούν τις ελλείψεις στην ενσωμάτωση, στην εφαρμογή και ε, στην ε, και στην ε, ε, συμμόρφωση με του κανόνε ιστορικής αγορά, με βάση την έρευνα που διεξήχθη από κοινού με τα κράτη-μέλη. Ε, θα δείτε επίση ε, σε παράρτημα τα συγκεκριμένα μέτρα που καλούνται να λάβουν τα κράτη-μέλη κράτη έτσι ώστε να ε, εφαρμόσουν τι υποδείξει αυτέ. Για να δούμε τώρα το πώ μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, δίδονται παραδείγματα των βέλτιστων πρακτικών στα κράτη-μέλη που απέδειξαν ότι είναι αποτελεσματικά. Αυτό το δίνουμε λοιπόν στο παράδειγμα για κάθε σύνολο μέτρων. Η ε, σύσταση επίσης συνοδεύεται από δύο ε, έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ένα περιγράφει το τι πράττει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα στον τομέα της ενσωμάτωσης, ε, της καθοδήγησης, μηχανισμοί επίλυση προβλημάτων και ένα άλλο έγγραφο το οποίο δίνει μια συνολική επισκόπηση των υφιστάμενων δικτύων για διοικητική συνεργασία σε επίπεδο εσωτερική αγορά. Για την Επιτροπή όλες ε, οι υποδείξεις είναι εξίσου σημαντικές και θα δείτε ε, τι επιμέρους διαφάνειες και τα συνολικά ε, σχόλια. Τονίζω όμως τρία σημεία. Το πρώτο αφορά την καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων και των πολιτών για, τα, για την εσωτερική αγορά και τις συνοριακές ευκαιρίες. Τα προτινόμενα μέτρα αφορούν την χορήγηση πρακτικών πληροφοριών με έναν τρόπο που να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ε, και να γίνεται σύνδεση και με τις εθνικές ε, πληροφορίες, να προωθήσουμε επίση τη συνειδητοποίηση για ε, ε, ότι είναι, τη συνειδητοποίηση ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, στον τομέα τη ε, εφαρμογή και συμμόρφωση με του κανόνε. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συμμόρφωση με του κανόνε τη ενιαία αγορά και να προωθήσουμε του μηχανισμού επίλυση προβλημάτων. Και εδώ τα προτινόμενα μέτρα είναι η εξασφάλιση απλών και μη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών από τα κράτη-μέλη, διαβίου κατάρτιση και εύκολη πρόσβαση σε, ε, των δικαστών στις πληροφορίες που αφορούν τους κανόνες εσωτερικής αγοράς. Και τρίτον, η τρίτη υπόδειξη που είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την εξασφάλιση και την ενίσχυση ε, του, του συντονισμού ε, της λειτουργίας εσωτερικής αγοράς σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα ανάμεσα στις αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εδώ το προτινόμενο μέτρο αφορά την, την πρόθεση της λειτουργίας σε θέματα εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση του συντονισμού σε όλα τα επίπεδα. Ένα σημείο το οποίο θα μας απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για πολύ καιρό. Τώρα το follow-up στη σύσταση, επειδή η σύσταση αυτή δεν επιβάλλει όπως είναι φυσικό καμία νέα υποχρέωση στα κράτη-μέλη, είναι σημαντικό να ε, ε, συνοδεύεται από το κατάλληλο follow-up. Και προβλέπουμε μια πολύ καλά οργανωμένη διαδικασία παρακολούθηση σε follow follow-up με τα κράτη-μέλη και έχουμε μια ομάδα εργασία με τα κράτη-μέλη που θα συναντάται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για να εξετάζει το πώ ε, εφαρμόζεται πρακτικά από τα κράτη-μέλη κάθε μία υπόδειξη ξεχωριστά. Τέλο Πρόεδρε, όπω είπατε και εσεί, το Συμβούλιο ήδη έχει εκδώσει συμπεράσματα για την, ε, σύσταση αυτή. Τα εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και μας ενδιαφέρει το θέμα της εφαρμογής, ε, της σωστής εφαρμογής και του follow-up. Και ζητάμε ιδιαίτερα την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε η όλη προσπάθεια να στεφθεί από επιτυχία και να δώσει όλες τις ευκαιρίες ε, που προσφέρει η εσωτερική αγορά και στους ε, πολίτες και στις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο ευρία παρουσίασή σας και επειδή μας δώσατε και όλες αυτές τις λεπτομέρειες, Έχουμε και εμεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τα οποία έστειλε η Γραμματεία σε όλα τα μέλη, άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε και τι απόψει του Συμβουλίου. Και η αρχική σα πρόταση, νομίζω, απεστάλλει τον Ιούνιο, έτσι. Ωραία. Δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μέχρι στιγμή. Ξέρω την κυρία Μπιούλη. Η πρόεδρο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα, όταν ήρθε να μιλήσει στην Επιτροπή μα αρχέ αυτού του μήνα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ζήτημα αυτό και, το έθεσε στο, και είπε ότι θα το θέσει στο επίκεντρο τη ημέρης τη διάταξης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα το Δεκέμβρη. Η κυρία Τούν βεβαίω μπορεί να θέλει να θίξει το ζήτημα αυτό και οι συντονιστέ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να παρέμβουμε, αλλά παρόλα αυτά σίγουρα θα ε, αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Νομίζω λοιπόν ότι ορισμένε παρατηρήσει σα, ε, κυρίω όσον αφορά το συντονισμό εσωτερική αγορά, καλύφθηκαν πλήρω όταν συζητήσαμε το ζήτημα με τη Σουηδική Προεδρία την περασμένη εβδομάδα και μπορούμε να συμπεριλάβουμε τη συζήτηση αυτή αλλά και συγκεκριμένη τεκμηρίωση που χρησιμοποίησε ε, η Σουηδική Προεδρία σε αυτή την προσπάθεια βελτίωση συντονισμού. Νομίζω τώρα θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε απευθεία με τη συζήτηση και με την παρουσίαση του θέματο ε, του πίνακα τη εσωτερική αγορά. Κυρία Καζάη θα μα το παρουσιάσει και μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Τιούν και θα προβούμε σε ένα γύρο τραπέζι με συμμετοχή των παρευρισκομένων. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής για να μας παρουσιάσει τον πίνακα βαθμολογίας. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Ορισμένοι μπορεί και να μην γνωρίζετε τον πίνακα ε, αποτελεσμάτων ε, της εσωτερικής αγοράς, οπότε, εν συντομία, μου δίνεται η ευκαιρία να σε εξηγήσω ποιος είναι και ο βασικός στόχος του πίνακα και να σε εξηγήσω γιατί αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία παρακολούθησης και τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Χαίρομαι ιδιαίτερος που έχω την ευκαιρία να σας κάνω αυτή την παρουσίαση για τον πίνακα αποτελεσμάτων. Ο βασικός στόχος του πίνακα είναι πρώτον να αυξήσει την ε, ευαισθητοποίηση των κρατών μελών σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στη διαδικασία μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και γενικότερα να, μιλήσει, να δείξει ποια είναι τα προβλήματα κατά τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες για να τηρήσουν τις προθεσμίες μεταφοράς ε, και πριν από 10 χρόνια γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε ότι πρέπει να παρακολουθούμε τις επιδόσεις των κρατών μελών για τη μεταφορά των κοινοτικών νομοθετημάτων στην εθνική νομοθεσία εκδίδοντας, ε, δημοσιεύοντας ε, δει στο χρόνο αυτό το πίνακα αποτελεσμάτων για να έχουν μια επισκόπηση τα κράτη-μέλη στη διάθεσή τους σχετικά με τις επιδόσεις τους και να έχουν και μια ενθάρρυνση έτσι ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους και να επικουρήσουμε και εμείς από πλευρά μας τα κράτη-μέλη. Ε, το, το, κοινό είναι πραγματικά τα κράτη-μέλη και οι, οι εθνικές αρμόδιες αρχές. Είναι ένα έγγραφο εργασίας αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων που τα κράτη-μέλη για να καλύψουν τις ατέλειές τους. Ε, όταν αρχίσαμε το 97 πώς είχε η κατάσταση. Τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, είχαν πολύ υψηλό έλλειμμα για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, πάνω από 6% προσέγγιζε τα 7% το έλλειμμα και γι' αυτό το λόγο δημοσιεύσαν πρώτη φορά το 1997, όπως σας έλεγα, τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς. Έκτοτε το έλλειμμα ε, συνέχισε να μειώνεται, ε, μειωνόταν διαρκώς μάλλον και ο φετινός πίνακας ε, του Ιουλίου δείχνει ότι έχουμε ένα έλλειμμα μόνο της τάξης μόνο του 1%. Ε, φαίνεται λοιπόν ότι έγινε σημαντική προσπάθεια βελτίωσης κατά τη διάρκεια αυτών των ετών και παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία πάρα πολύ χρήσιμη όπως φάνηκε και από τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας. Τι θέλουμε να επιτύχουμε τώρα. Έχουμε φτάσει, είπαμε, στο 1%. Καλό φαίνεται, καλό ακούγεται, είναι καλό, αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να μειώσουν περαιτέρω το έλλειμμα του. Ε, εξακολουθεί να είναι υψηλό, ακόμη και στο 1%. Κάποια κράτη-μέλη, 9 συγκεκριμένα, απέχουν πόρο από ένα τέλειο βαθμό μεταφοράς. Η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση έχει διπλό έλλειμμα, άνω του 2,1%. Παρά είναι υψηλό το ποσοστό. 18 ε, μονοκράτη λοιπόν είναι ε, κάτω του ε, στόχου ελλείμματος του 1% που κρίνουμε ότι είναι εύλογο αν θέλετε. Αυτό συνιστά βελτίωση, αλλά η έγκαιρη μεταφορά, η έγκαιρη υλοποίηση είναι ένα πρώτο βήμα. Ε, τώρα ο στόχος μας ε, θα ε, μετατοπιστεί προς μια ορθότερη μεταφορά. Αν δούμε ποιες οδηγίες δεν έχουν μεταφερθεί και ποιες δεν έχουν μεταφερθεί ορθά, διπλασιάζεται το έλλειμμα, φτάνει στο 2%. Έχουμε υπερβολικά πολλά κενά στο νομικό πλαίσιο και αυτό δημιουργεί έλλειψη ασφάλειας δικαίου σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Και γι' αυτό θα εστιάσουμε, λένε και περισσότερο, την προσοχή μας στην ορθή μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Αυτό κάνει ο πίνακα αποτελεσμάτων δείχνοντας ε, και τις ε, υποθέσεις ε, Διαδικασία για παράβαση που ε, ε, υπάρχουν για τα διάφορα κράτη-μέλη δεν έχει σημειωθεί ε, βελτίωση σημαντική τα τελευταία πέντε χρόνια. Η Ιταλία έχει τις περισσότερες τέτοιες υποθέσεις παραβίασης, ακολουθεί η Ισπανία και αυτό είναι μεγάλη μελλοντική πρόκληση για μας. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των υποθέσεων παραβίασης. Οι περισσότερες οφείλονται σε ε, πλημελή μεταφορά της εθνικής νομοθεσίας και πλημελή εφαρμογή της ε, κοινοτικής ε, νομοθεσίας. Στο μέλλον θέλουμε λοιπόν να εστιάσουμε όλους ιδιαίτερο σε τομείς όπου τα κράτη-μέλη φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες και θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγι στη διαδικασία για να επικουρήσουμε τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Μπρέμτη και κυρία Ρίτσιου για, τις, ε, ε, για τη σαφή παρουσίαση αυτών των ζητημάτων. Κυρία Τούν, είστε η συγγήτριά μας για την έκθεση για τον πίνακα αποτελεσμάτων εσωτερική αγορά και πρόταση μέτρων για τη βελτίωση τη λειτουργία εσωτερική αγορά. Ε, θα σα δώσω το λόγο. Δεν ξέρω αν έχουμε σκιώδει συγγητέ που έχουν οριστεί. Εν πάση περιπτώσει, όποιο θέλει το λόγο μπορεί να τον ζητήσει. Η κυρία Τούν πρώτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους. Και ευχαριστούμε βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συστάσεις της. Ε, προφανώς ε, για κάτι τέτοιο αυτές οι πρωτοβουλίε ε, ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και ε, προσφέρουν κίνητρα για αναπτύξει στην Ευρώπη, τα οποία χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Οι οδηγίε για την εσωτερική αγορά αποτελούν ε, το, ε, το βασικό στοιχείο της σπονδυλικής στήλη για μια αγορά και βέβαια η σωστή ε, εφαρμογή και η συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες της εσωτερικής αγοράς οδηγούν στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ενδυναμώνουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το, αυτό θεματικό πεδίο και για μας ε, και αφιερώνουμε σε αυτό πολύ χρόνο. Αναφερθήκατε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ε, της τελευταίας εβδομάδας ε, που έλαβε χώρα εδώ στις Βρυξέλλες. Ναι, συμφωνώ με τα συμπεράσματα. Εκείνα και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο από αυτά υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη και συνεκτική ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της πλήρους ε, και ε, έγκαιρης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες και θεωρούμε πως ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο. Χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευρύνει και εργαλεία στη διάθεσή τη και ε, την καλή να συνεχίσει να ε, σημειώνει την πρόοδο που ε, σημειώνεται σε ορισμένου τομεί. Άρα λοιπόν μόνο να χαιρετίζουμε μπορούμε τέτοιου είδου συμπεράσματα και ω προ την έκθεση να πούμε πω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο. Ελπίζω πω θα το εξετάσετε λίγο πιο προσεκτικά. Απευθύνομαι στου συναδέλφου μου. Είναι ο πίνακα 19, ο οποίο καταρτίζεται δύο φορέ το χρόνο και παρά ε, όλες τις προκλήσεις ε, που ε, αντιμετωπίζουμε καταδεικνύει τις επιτυχίες της εσωτερικής αγοράς. Τρεις προκλήσεις αντιμετωπίζουμε σήμερα και επιτρέψτε μου να τις αναφέρω ξανά. Πρώτον, οι καθυστερούμενες οδηγίες. δηλαδή για αυτές τις οδηγίες που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα έχει ήδη περάσει η προθεσμία των δύο ετών ε, και το Συμβούλιο έχει θέσει συγκεκριμένε ε, ε, κυρώσει για κάτι τέτοιο. Και παρόλα αυτά έχουμε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμα με αυτέ τι προθεσμίε περί μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, παρότι αυτέ έχουν συμμορφωθεί από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Δεύτερη πρόκληση Ε, όλα τα κράτη-μέλη επιτυγχάνουν ε, το στόχο. Δηλαδή αυτό το στόχο του λιγότερου από 1%. Εδώ στο πίνακα αποτελεσμάτων έχουμε 9 κράτη όμως μέλη τα οποία δεν επέτυχαν αυτό το στόχο. Και το τρίτο ε, σημείο είναι αυτό που αναφέρατε. Η συνοχή της νομοθεσίας. 1,8% των οδηγιών είναι αυτές οι οποίες δεν εφαρμόζονται στο ακέραιο ή με τον σωστό τρόπο. Πράγματι θα πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτό, το αναφέρετε και εσείς στη δική σας παρουσίαση. Καθώς ε, η συνέπεια της μη εφαρμογής, της ελπούς εφαρμογής, είναι ο κατακαιρματισμός της ε, εσωτερικής αγοράς. Ε, κατακαιρματισμός σε επίπεδο 6% που σημαίνει ότι 100 οδηγίες της εσωτερικής αγοράς δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δικαίωμα των Κρατωμενών Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δημιουργεί νομική αβεβαιότητα και ε, βέβαια συνεπάγεται ε, διαφορετικούς ευκαιρίες ε, για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη. Στις χώρες εκείνες όπου δεν εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες η εσωτερική αγορά δεν αποτελεί πραγματικότητα. Οι τομεί στου οποίου σημειώνονται οι παραβάσει είναι πάρα πολλοί. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι κλάδοι στου οποίου έχουμε τι περισσότερε διαδικασίε κατά παράβαση είναι αυτή τη φορολόγηση τη Τελωνιακή Ένωση και του περιβάλλοντο, καθώ ε, συνιστούν περίπου ή αντιστοιχούν περίπου στο 50% των ε, διαδικασιών παραβάση. Αυτό λοιπόν αποτελεί σημαντική πρόκληση και για να κλείσω να πω ότι χαιρετίζω τις συστάσεις που ε, μας ε, ε, προέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ πως η τακτική κατάρτιση των σχετικών ειδικών από την των κρατών μελών και ανταλλαγή απόψεων θα οδηγήσει σε καλύτερα ε, αποτελέσματα και η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να ελέγχεται διαρκώς ε, από κοινού με την ε, παρακολούθηση της ευρωπαϊκής νομολογίας θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, για παράδειγμα, ε, σε πλατφόρμες όπως το Solvit, ε, την πλατφόρμα δηλαδή για την αποκοινού επίλυση των ε, προβλημάτων λαθασμένης ή ελλειπούς εφαρμογής κοινοτικής νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες κατά παράβαση, είναι πολύ σημαντικό να επιταχύνουμε την διαδικασία της επίλυσης των διαφορών σε ένα πρόμοιστο πρώιμο στάδιο και να έχουμε μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων ώστε να ασχολούμαστε με εκείνε τι περιπτώσει παραβάσεων οι οποίε είναι οι πλέον σημαντικέ για του Ευρωπαίου πολίτε. Όπω ήδη αναφέρθηκε, ο πίνακα αποτελεσμάτων θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο σε ένα χρήσιμο εργαλείο για του ε, αρμόδιου για τη χάραξη τη ε, πολιτική ω προ τον εντοπισμό εμποδίων στη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Ε, μέσω αυτής της έκθεσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση ε, στην ε, διάδοση ε, αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων και να, θα πρέπει να αυξηθεί η προσβασιμότητά του από τους πολίτες αλλά και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα πρέπει δηλαδή να είναι διαθέσιμος αυτός ο πίνακας των αποτελεσμάτων και στις ισοσελίδες των σχετιζόμενων φορέων με ένα διαφανή και εύκολα κατανοητό τρόπο. Ε, και χρειάζεται εδώ να υπάρξει ε, ενδιαφέρον από την πλευρά ε, και των εκατομελών και της Επιτροπής ούτως ώστε να δούμε πώς σχετίζονται οι αγωνισμοί με τους πίνακες αποτελεσμάτων. Αυτή η σχέση είναι πολύ σημαντική για μένα και αναμένω πως όλοι μας εδώ οι συνάδελφοι θα έχουμε να μοιραστούμε μεταξύ μας εμπειρίες σε αυτό το τομέα, καθώ ε, όλοι σχετιζόμαστε με τον ένα τον άλλο τρόπο με τι φορολογικέ αρχέ τη χώρα μα. Και άρα λοιπόν αναμένω ε, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα με όλου σα και μου ζητήθηκε από την ε, γραμματεία να σας κοινοποιήσω το εξής χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε σε ό,τι αφορά τη συζήτηση και τις τροπολογίες. Σήμερα λοιπόν συζήτηση, προθεσμία 15 Οκτωβρίου για να αποσταλεί για μετάφραση το σχέδιο εξέταση του σχεδίου 5 Νοεμβρίου, προθεσμία αποβολή τροπολογιών 9 ε, Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου, ε, ψήφιση ε, της έκθεσης εδώ, στην ΙΜΚΟ και ε, τον Ιανουάριο στην Ολομέλεια. Και να σας πω ότι είμαι βέβαια πάντα εδώ στη διάθεσή σας για να το συζητήσω αυτό το ζήτημα τόσο με τους κοιόδης συζητητές ή οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο ενδιαφέρεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Τούν και για το χρονοδιάγραμμα και για τις διευκρινήσεις. Ε, δεν έχουμε τους σκιώδες εδώ. Ο κύριος Λούχεγκαρντ ε, έχει ζητήσει πρώτο το λόγο. Νομίζω πρώτη φορά θα πάρει το λόγο στην Επιτροπή. Αλλά ήταν πολύ δραστήριο την περασμένη εβδομάδα που ήμασταν στη Σουηδία. Μετά η κυρία Γκέπχαρτ. Ποιος άλλος? Η κυρία Ράπτη, μάλιστα, και ο κύριος Μπίλεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτη φορά παίρνω το λόγο και θα μιλήσω στα δανέζικα. Øh, er, er Νομίζω πως ε, πρόκειται εδώ για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, τομέα και ως ε, Δανός ενδιαφέρομαι πάρα πολύ ε, για το ζήτημα του πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο την ενιαία αγορά. Εγώ δεν έχω διαβάσει ακόμα την έκθεση, η οποία μας παρουσιάστηκε εδώ, αλλά ε, έχω να θέσω κάποια ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω πως ε, οι απαντήσεις θα μας δώσουν νέα ρεθίσματα για σκέψη. Συχνά αναφερόμαστε ως προς την αποτελεσματικότητα εδώ της νομοθεσίας και ε, σε κάποια ε, νούμερα, δηλαδή κάποια χρήματα τα οποία μπορεί να αντλήσει από τέτοιου είδους διατάξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε εδώ για αριθμούς οι οποίοι φτάνουν ε, τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως δηλαδή εξοικονομήσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε αν πράγματι είχαμε καλύτερη εφαρμογή, καλύτερες πρακτικές εδώ έχει ακούσει τέτοιου είδους νούμερα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρησιμοποιεί δηλαδή τέτοιου είδους εκτιμήσεις, κάτι τέτοιο βέβαια προφανώς και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό, για την κοινή γνώμη, το να ακούσει συγκεκριμένα νούμερα, ούτως ώστε να έχουμε κάτι μετρήσιμο. Κάτι αυτό ως προς το τι μπορεί πράγματι να μας φέρει ως κέρδος η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε αν έχετε τέτοια συγκεκριμένα νούμερα. Ε, άλλο ερώτημα. Ε, τι θα συμβαίνει σε περίπτωση όπου δεν ε, ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του στα κράτη-μέλη. Προβλέπετε Θα υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες επιβολής ε, κυρώσεων στα εν λόγω κράτη-μέλη. Και αν έχουμε επιτύχει κάποιες σχετικές προόδους, αν υπήρξαν κάποιες επιτυχίες όπως μας λέτε, τι κάνατε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, υπήρξαν δηλαδή κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν, ε, χρειάστηκε να ασκήσετε πιέσεις με άλλους τρόπους. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με το ζήτημα της επικοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό θεωρώ πως ε, τόσο εμείς όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τονίζουμε ε, ξανά και ξανά ότι θα πρέπει να κοινοποιούνται αυτές οι επιτυχίες στο ευρύ κοινό, ε, στις επιχειρήσεις, σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την εύρυθμη λειτουργία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. Uh, Mrs. Ευχαριστούμε, κυρία äh, äh, Ευχαριστώ. Ε, εμείς από την πλευρά της δικής μας πολιτικής ομάδας ε, ε, δεν έχουμε ακόμα ορίσει εισηγητή ή εισηγήτρια, αλλά μόλις θα ορίσουμε θα σας το κοινοποιήσουμε βέβαια, την εισηγήτρια. Να πούμε λοιπόν καταρχήν πως πράγματι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό εργαλείο προκειμένου να καταγράψουμε την κατάσταση όπως αυτή ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχετε δίκιο όταν λέτε ε, πως δεν μπορεί ο νομοθέτης ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ε, υιοθετούν κάποια, ε, κάποια νομοθεσία, κάποιε νομοθετικέ πράξει και στη συνέχεια αυτέ να μην εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, κάτι πρέπει να γίνει εδώ. αυτό αναφέρεται και θα πρέπει να αναφέρεται μέσα στη δική σα έκθεση. στη συνέχεια αναφερθήκατε στην ΟΔΙΕ για τις υπηρεσίες, μια από τι πλέον σημαντικέ νομοθετικέ πράξει του τελευταίου καιρού σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά. Ε, θα πρέπει να πω σε σχέση με αυτό το τομέα στην εισηγήτρια ότι θα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εφαρμοστεί πράγματι αυτή η οδηγία. Συζητήθηκε επί μακρόν και γι' αυτό και στην ε, συζήτηση των ε, συντονιστών που κάναμε αποφασίσαμε να αποστείλουμε γραπτή επερώτηση στο Συμβούλιο μέσα στο Νοέμβριο, εάν μας το επιτρέψει το χρονοδιάγραμμά μας, ως προς την κατάσταση που ισχύει στα κράτη-μέλη ως προς την εφαρμογή της. Προφανώς και η προθεσμία τους ε, τέλει αυτού του χρόνου, αλλά με βάση τις πιέσεις που βλέπουμε θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα ήθελα εδώ να ε, θυμίσω κάτι. Ως εισηγήτρια, όταν βρισκόμαστε στη φάση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, είχαμε προτείνει στο Συμβούλιο των Υπουργών να ξεκινήσει η εφαρμογή ένα χρόνο πιο αργά. Γιατί πραγματικά η οδηγία ε, για τις υπηρεσίες ε, αφορά ένα πολύ ευρύ πεδίο σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ε, σχετικές νομοθεσίες. Και οι υπουργοί μας λένε, μας είπανε τότε ότι όχι, δεν χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Είναι λοιπόν τώρα ευθύνη τους να διασφαλίσουν ότι πράγματι θα υπάρξει αυτή η εφαρμογή. του είχαμε δώσει αυτή τη δυνατότητα να υπάρξει μεγαλύτερη ε, προθεσμία μέχρι την έναρξη της εφαρμογή. Και μάλιστα ε, είχα φροντίσει ούτως ώστε αυτό να περιληφθεί στην έκθεσή μας, δηλαδή αυτή η πρόταση που είχαμε κάνει, ούτως ώστε να είναι αυτό ορατό από όλους. Ε, ένα τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω το οποίο βασικά αποτελεί ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ίσως βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε ξανά, κυρία είναι η αξιολόγηση ε, όλων εκείνων των στοιχείων, τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά ή ελλιπώς. Ε, με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Γιατί προφανώ έχουμε εδώ να κάνουμε μια πολιτική φύση απόφαση και γνωρίζουμε πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ή και το Συμβούλιο δεν ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο τα νομοθετικά κείμενα. Άρα λοιπόν, σε ποιο βαθμό λαμβάνεται υπόψη αυτός ο παράγοντας αυτή η διαφορετική δηλαδή ερμηνεία στην κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις παραβάσεις, τα infringements ή όταν η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσφέρει στο δικαστήριο για να αξιώσει τα δικαιώματα εκείνα τα οποία θεωρεί πως αντλούνται από το κείμενο ε, μια συγκεκριμένη νομοθετικής πράξης. Θα πρέπει να λαμβάνουμε κάποιες ε, πληροφορίες στο πλαίσιο αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων ως προς το σε πόσες ε, περιπτώσεις τελικά είχε δίκιο ως προς την ερμηνεία που έδωσε στην ε, νομοθεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ποιες περιπτώσεις δεν είχε δίκιο. Γιατί πραγματικά ε, η εφαρμογή μιας νομοθετικής πράξης αποτελεί και πολιτικού χαρακτήρα ερμηνεία των όσων έχουμε αναφέρει μέσα στο νομοθέτημά μας. Γιατί συχνά ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένο ένα νομοθέτημα ε, αφήνει τέτοια περιθώρια και συχνά τελικά ε, είναι αρμόδιο το δικαστήριο να αποφασίσει μέσω της νομολογίας τι συμβαίνει. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε και κάτι τέτοιο στον πίνακα αποτελεσμάτων. Αυτό θα μας βοηθούσε να ε, διαπιστώσουμε πώς θα ερμηνεύσουμε αυτούς τους αριθμούς στην πραγματικότητα, τους αριθμούς δηλαδή που έχουμε λάβει τώρα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τέσσερις ομιλητές και οχτώ λεπτά και ε, δεν, μπορεί, δεν υπάρχει χρόνος για να κλείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τους τέσσερις ομιλητές ε, μπορείτε, σας παρακαλούμε, να κάνετε μονόλεπτες παρεμβάσεις ε, για να απαντήσει κάπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτως ή άλλως, κυρία Τουν, θα ξανασυζητήσουμε το θέμα. Κυρία Ράπτη, ένα λεπτό σας παρακαλώ, δεν θα βάλω χρονόμετρο. Μία ερώτηση μόνο στην Επιτροπή. Επειδή αναφέρθηκε στην Ελλάδα και στους όχι καλούς αριθμούς που παρατηρούνται στους πίνακες, τους κοίταξα κι εγώ, η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ μικρή. Γιατί διστάζετε να χρησιμοποιήσετε ως Επιτροπή και να κινήσετε τη διαδικασία επί παραβάση. Τίποτα άλλο. Very short, sharp question. Mr. Πολύ σύντομη η ερώτησή σας, όντως, ε, και πολύ συγκεκριμένη. κύριος Μπίλεν. Πρόεδρε, ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει μεγάλη επιτυχία. Στη διαφάνεια 3 βλέπουμε αποδείξεις σχετικά με τη μείωση του ελλείμματος ως προς ε, την ε, περίοδο μεταφοράς σε τελευταία δεκαετία. Είμαι από την Πολωνία και βλέπω ότι είμαστε από τους χειρότερους μαθητές, αλλά δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Έχουμε τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, που είναι πρώτη-πρώτη βάσει των στατιστικών. Συχνά παρουσιάζεται, θυματοποιείται η Πολωνία στα ΜΜΕ, ε, παρουσιάζεται ως θύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντάξει, εκδίδει αυτά τα εσωτερικά έγγραφα, αλλά θα πρέπει να ασχοληθεί και με την κοινή γνώμη. Ο κύριος Σβάπ. Ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να πω πως η δουλειά που έχει κάνει άλλη ε, σχέση με αυτό το έγγραφο είναι πολύ καλή και θα ήθελα να το ευχαριστήσω και ε, σήμερα το απόγευμα όταν θα συζητήσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε πολύ λίγες ε, τέτοιου είδους αξιολογήσεις, δομημένες αξιολογήσεις ως προς το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ιστορική αγορά, για τους καταναλωτέ, αλλά πολύ λίγα υπάρχουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ε, και την πρακτική που ακολουθείται σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Πράγμα βέβαια το οποίο μας δημιουργεί δυσκολίες στο να περιγράψουμε το πώς έχει κατάσταση στα 27 κράτη-μέλη. Ε, και γι' αυτό, σε σχέση με την, ε, ε, με την εφαρμογή των οδηγιών, θα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, ώστε να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε καλύτερα την αγορά με όλη την περιπλοκότητα. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βερνιώτη, την Αντιπρόεδρο, πολύ σύντομα, ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ε, ύψιστα πολιτικό και πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίου πολίτες. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρόκειται και το είπαν και όλοι για αύξηση ε, του περίπλοκου χαρακτήρα ε, και του διοικητικού άχθους το οποίο το βλέπουν με πολύ κακομάτι και οι επιχειρήσει και οι πολίτες. Αντίθετα να αποδείξουμε και εδώ είναι πολιτικό το σημείο, άσχετο με το αν περνάει μέσα από τεχνικέ λεπτομέρειε. Να δείξουμε λοιπόν ότι η εσωτερική αγορά βεβαίω και αποτελεί ευκαιρία για την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη, δηλαδή και των επιχειρήσεων, αλλά είναι και στην υπηρεσία των πολιτών στην καθημερινή του ζωή. Όλοι μιλήσαμε για την απουσία σωστή ενσωμάτωση. Και όταν βλέπουμε ότι υπάρχει 22% ε, των οδηγιών που δεν έχει μεταφερθεί ε, από τα κράτη-μέλη, πράγματι εδώ, όπω ε, είπε και η συγκήτρια, έχουμε πολλά να κάνουμε θα πρέπει εντάξει, να μην βιαστούμε, αλλά να σημειώσουμε πρόοδο. Γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ε, το οποίο ε, είναι πολύ σημαντικό σε περίοδο κρίση και σε οικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και θα πρέπει να εξαλείψουμε την νομική ασάφεια που είναι αβάσταχτη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και για του πολίτε και του καταναλωτέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα αυτό, το οποίο μπορεί να φαίνεται σαν κάτι ε, και δεδαλώδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για μας σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς θα μπορέσει να αποτελέσει ένα εργαλείο επικοινωνίας για αύξηση του γοήτρου της Ευρώπης. Αλλά εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που είναι τεράστιες φυσικά. Uh, right. Ευχαριστώ. Έχει περάσει ο χρόνος. Ίσως όμως ε, θα μπορούσαμε να καλέσουμε την κυρία Μπράπτον αν θέλει να απαντήσει σε ορισμένα από τα ζητήματα αυτά πολύ σύντομα. Και μετά θα δώσω και στην εισηγήτρια το χρόνο. Α, όχι, στην κυρία Καζάη. σα ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, εάν μπορούμε να μετρήσουμε το κόστο τη καθυστέρηση στην ενσωμάτωση. Προσπαθήσαμε στο παρελθόν, αλλά φάνηκε σχεδόν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε το πόσο κοστίζει δηλαδή στην ουσία η έλλειψη έγκαιρης ενσωμάτωσης. Γιατί είναι σχεδόν αντίνετο. Γιατί πρέπει να δούμε τους δείκτες που θα, θα λάβουμε ε, ως βάση. Πώς θέλουμε να μετρήσουμε το κόστος. Ανάλογα με τη σημασία της οδηγίας, με την οικονομική αξία της συγκεκριμένη οδηγία. ή με, το, με την επίπτωση της οδηγίας στους πολίτες, αν είναι τεχνικής φύσεως ή όχι επίσης κτλ. Προσπαθήσαμε λοιπόν, όπως σας είπα, να το κάνουμε στο παρελθόν, αλλά οι οικονομικοί εμπειρογνώμονές μας ε, και οι άλλοι εμπλεκόμενοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί τρομερή αβεβαιότητα και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να επιδοθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά την ερώτηση για τις κυρώσεις, τι κάνουμε σε σχέση με τα κράτη-μέλη τα οποία δεν ενσωματώνουν έγκαιρα. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι εύκολη. Η μη, ε, ε το να μην ακολουθεί κανεί ε, τη διαδικασία ενσωμάτωση, ε, η διαδικασία είναι αυτόματη. Δηλαδή, αν δεν ενσωματώνει μέσα σε ένα μήνα το κράτο μέλο μετά την εκνοή τη προθεσμία, για την ενσωμάτωση, αμέσως ξεκινάμε τη διαδικασία παραβάση. Άρα στέλνουμε το, το κράτος μέλος στο δικαστήριο. Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να δράσουμε. Και επανειλημμένα το έχουμε κάνει. Σας είπα ότι είναι σχεδόν αυτοπαιματοποιημένη η προσέγγιση αυτή. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία για το ότι τα κράτη-μέλη θα τιμωρηθούν σε περίπτωση μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο μη ενσωμάτωση ε, των ε, οδηγιών. Τώρα, γιατί έχουμε αυτόν τον, βαθμο, ε, τον πίνακα και γιατί τα, τα κράτη-μέλη έχουν καλύτερε επιδόσει. Γιατί δημιουργώντα αυτή την peer pressure, την πίεση των ομοτήμων στα κράτη-μέλη και με τη μεγαλύτερη διαφάνεια, να προβάλλουμε τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν καλέ επιδόσει θετικά και αρνητικά εκείνα τα οποία δεν έχουν καλέ επιδόσει, καταλαβαίνετε ότι δείχνουν προθυμία τα κράτη-μέλη. Γιατί σα διαβεβαιώνω, κανένα κράτο-μέλο δεν θέλει να βλέπει ε, τον ε, εαυτό του ε, στο κάτω μέρο του πίνακα. Αισθάνονται μεγάλη μηχανία και προσπαθούν να βελτιώσουν τι επιδόσει του. Γιατί η πίεση σε εθνικό επίπεδο είναι μεγάλη. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα αποτελέσματα. Κάθε φορά που εκδίδουμε τον πίνακα βαθμολογίας είναι τεράστιες οι εντράσεις ε, μας έρχονται email ε, από τα κράτη-μέλη και από τον τύπο, μας ρωτούν ε, πού βρίσκονται κτλ. Είναι όλοι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να βελτιώσουν τα πράγματα για να μην είναι και οι κακοί μαθητές της τάξης. Η πίεση λοιπόν των ομοτήμων αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο και θέλουμε να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, Σα ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Λυπάμαι, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μα. Ε, ε, δεν θα έχουμε πλέον διερμηνία. Ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε διεξοδικά. Μήπω ε, θα μπορούσατε να μα στείλετε ένα σύντομο σημείωμα γιατί προφανώς έχετε πάρει σημειώσεις και κρατήσατε τις ε, απαντήσεις. Θέλετε να, μιλήσετε, να απαντήσετε την κυρία Γκέφχαρτ, έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ε, λυπάμαι ιδιαίτερα που σας στερώ την δυνατότητα απάντησης, αλλά θα, μπορώ, θα πρέπει να συνεχίσουμε χωρίς διερμηνία. Σας ευχαριστώ πάντως ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και μας κάνετε την παρουσίαση αυτή. Μήπως μπορείτε να μας στείλετε ένα σημείωμα. Και η κυρία Τούν είμαι σίγουρος ότι ε, θα χαρεί ιδιαίτερα να συνεργαστεί μαζί σας και με την εισηγήτρια. Κυρία Τούν, θέλετε να πείτε δύο λόγια, τελευταία λόγια πριν διακόψουμε και το μεσημεριανό διάλειμμα. Απλά θα ήθελα να πω ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή, για την παρουσίαση και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και το αποτέλεσμα θα είναι τελικά να βρούμε περισσότερα ε, κίνητρα προς τα κράτη-μέλη για να μεταφέρουν γρηγορότερα και ε, καλύτερα τις οδηγίες στην εσωτερική νομοθεσία και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστώ όλους. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, γιατί αναλάβατε αυτή την πρώτη σας εργασία ως συγγήτρια. Περιμένουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Θα περιμένουμε και την τελική ε, δομή της πρότασής σας για το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα προτείνεται ψήφο την 1η Δεκεμβρίου, θα μας επιστρέψει να στείλουμε το σωστό μήνυμα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις απόψεις για ε, το πακέτο μέτρων που θα βελτιώσουν τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Ε, παρόλο που δεν θα έχουμε ψηφίσει στην Ολομέλεια, νομίζω θα αναλάβουμε το κίνδυνο και το ρίσκο. Θα το συζητήσετε το χρονοδιάγραμμα. θέλετε και άλλα πράγματα να κάνουμε σε συνεργασία με τι πολιτικέ ομάδε εντάξει, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι ίδιε οι πολιτικέ ομάδε. Πάντω, νομίζω θα, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμά σα και να πετύχουμε το στόχο μα. Ε, οι συντονιστέ συνέχεια θα αποφασίσουν. Πάντω, εμεί σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σα ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε την Επιτροπή που ήρθε εδώ σήμερα για να ε, παρουσιάσει το ζήτημα. Περιμένουμε ε, να τα πούμε και το απόγευμα στι 3 η ώρα. Ο κύριο Βάμπ θα ε, έρθει για να έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση για την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ όλους.